So, um, Κυρίες και κύριοι, με χαρά ξεκινάω την απογευματινή συνεδρία. Θα με συγχωρέσετε, θα μιλήσω γαλλικά. Με μεγάλη μου χαρά προεδρεύω της πρώτη συνόδου του απογεύματος. Ευχαριστώ τους οργανωτές, την οργανώτρια, μάλλον αυτής της ε, διάσκεψης, που μου ζήτησε να προεδρεύσω για ένα θέμα που τόσο πολύ με νοιάζει. Βλέπω τη νέα διάσταση στο δίκτυο Monnet. Χαίρομαι διότι βλέπω όλους αυτούς τους συμμετέχοντες και μιλάμε για υψηλό ποιοτικό επίπεδο πάντα. Οπότε είναι τιμή μου και χαρά μου που προεδρεύω αυτή συνόδου πολύ ενδιαφέρον το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Το θέμα βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών τη στιγμή της ηθίκης της Λισαβόνας. Περνάμε πλέον σε νέα φάση, οι δύο όροι, θεμελιώδη δικαιώματα και ηθαγένεια, είναι όροι προβληματική από πλευράς περιεχομένου και ορισμού και πάρα πολύ σημαντική για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Τώρα τους έχουμε από κοινού, ενώ και ξεχωριστά θα μπορούσαμε να τους αφιερώσουμε ολόκληρη διάσκεψη. Λοιπόν, έχουμε από κοινού τα δύο σημεία. Εντάχει θα μιλήσω βεβαίως, για να μην χάνουμε χρόνο εξαιτία μου. Έχουν κοινά στοιχεία η συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει λύσεις, επιφέρει βελτίωση. Μιλάμε για νέες προοπτικές, κατά κάποιο τρόπο ναι. Η συνθήκη της Λισαβόνας επιβεβαιώνει κάποιες αξίες, υπογραμμίζει τις δημοκρατικές αξίες, αναγνωρίζει μέσω της χάρτας των δικαιωμάτων. Υπάρχει και κεφάλαιο ξεχωριστό για την Ιθαγένεια και τα πρωτογενή δικαιώματα και άλλες σημαντικές πτυχές των θεμελιών δικαιωμάτων που κατά κάποιο τρόπο μάλιστα η συνθήκη της Λισαβόνα ε, παρέχει με κάποια ανανέωση. Η συνθήκη της Λισαβόνα ρυθμίζει τις εκκρεμότητες. Όχι, προφανώς. Παραμένουν κάμποσα προβλήματα. Εξού και η σημασία της απογευματινής συζήτησης. Παραμένουν προβλήματα, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε κάμποσα. απειλούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα και η ηθαγένεια λόγω της τρομοκρατίας, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής ύφασης, λόγω της μετανάστευσης, λόγω θεμάτων που ξεπερνάνε την ε, Ευρώπη. Επανέρχονται τα ίδια προβλήματα. Και άλλο θέμα που θα πρέπει να προσέξουμε. Το πεδίο της ηθαγένειας και το πεδίο των θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν είναι απαραίτητο στα ίδια. Έχουμε το τεράστιο πρόβλημα της μετανάστευσης των υπηκών τρίτων χωρών στον ευρωπαϊκό χώρο. Άρα, τι μπορούμε να πούμε για τους δύο αυτούς όρους, δηλαδή δικαιώματα και η ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Αυτά είναι που όλα αυτά μας προβληματίζουν. Όντως έχουμε νέες προοπτικές. Ήδη η Κομισιόν προχωρά σε προβληματισμό για τον χώρο ελευθερίας, ε, δικαιοσύνης και ασφάλειας για την ε, κατάρτιση του προγράμματος Στοκχόλμης. Ποιο χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας θέλουμε για τον Ευρωπαίο πολίτη. Αλλά το θέμα πάει και πέρα σε σχέση με τον Ευρωπαίο πολίτη. Το είδαμε και σήμερα στο πλαίσιο των νέων θεσμικών ισορροπιών διαθέτει τα μέσα όντω η Κομισιόν ε, για να προτείνει κάποιες λύσει. Ιδού κάποια από τα ερωτηματικά που έχουμε κατά νου. Θα έχουμε σίγουρα πολύ καλές συνεισφορές από τους συμμετέχοντες. Στα δεξιά μου έχουμε τον καθηγητή Ινίκο Μέντεθ Ντεβίγο με όλους του τους τίτλους που μπορείτε να τους δείτε στο πρόγραμμα Ποτέ δεν θα ξεχάσω πάντω τους αγώνε μα υπέρ τη χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και μετά του συνέχισε και στη συνέλευση και σε χίλια δυο άλλα μέτωπα. Μετά, έχουμε μαζί μα τον κύριο Ορέλ Τσαμπάνο Ντορντέα, είναι διευθυντή, έχει την αρμοδιότητα σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, στην Κομισιόν. Αφιερώσαμε πολύ χρόνο για το θέμα της υποψηφιότητας της χώρας σας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θυμάστε γι' αυτό. Μετά έχουμε δύο ακαδημαϊκούς μαζί μας, την ε, καθηγήτρια Elspeth Guild, έχει την έδρα Ζαμονέ και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Νίμεκ και ο καθηγητής Σιντάνσκι, που θα είναι ο πρώτο τελευταίο μας ομιλητής και μετά ο Πιάγ Λεμουάν, ο οποίο είναι εκδότη για ε, τη, στο Europolitics. Ευθύσαμε στο λόγο στον ε, κύριο Μέντες Δεβίγκο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, πράγματι. Δέκα χρόνια πέρασαν, α, για, σένα, για σας, εσάς δεν φαίνεται, πέρασαν πάντως δέκα χρόνια από τότε που είχαμε τη τιμή και τη μεγάλη χαρά να συμμετάσχουμε σε μία από τις πλέον συναρπαστικές περιπέτειες, σε ευρωπαϊκό επίπεδο τουλάχιστον, όπως η σύνταξη της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ο Ρόμαν Χέρτσοχ προείδρευσε τη συνέλευση. Και κατόπιν αυτού περάσαμε στη δεύτερη συνέλευση που κατήρθησε πλέον τη συνταγματική συνθήκη. Και μετά τα γνωστά επεισόδια προέκυψε κάποια στιγμή και η συνθήκη της Λισαβόνας. Ήταν ένα είδος γενικής δοκιμής ας πούμε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο συνελεύσεων. Η πρώτη συνέλευση που κατήρθησε τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ήταν με καθηγητές. Με συμμετοχή καθηγητών. Οι τεχνικές πτυχές δηλαδή ε, έπαιξαν ρόλο καθοριστικής σημασίας. Θυμάμαι τις πρώτες μας συζητήσεις ε, το Δεκέμβριο του 1999 κατά πόσον θέλαμε χάρτη νομικής, χάρτα νομικής εμβέλειας ή χάρτα που να αποτελούσε πολιτική δήλωση. Θυμάμαι πολύ καλά τι μας έλεγε ο πρόεδρος Χέρτσοκ. Προσπαθούσε να βρει λύσεις. Τι μας έλεγε. Θα δουλέψουμε ως να επρόκειτο να προσαρτηθεί η χάρτα στις συνθήκες. συμμετείχαν ακόμα και πολιτικοί που ταυτόχρονα ήταν και καθηγητές. Δουλέψαμε με βάση να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα που τελικά ε, ήταν αποτέλεσμα νομικών. Μέσα σε δέκα μήνες καταρτήσαμε τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Θυμάμαι ότι θεωρήθηκε ενδιάμεση φάση. Ο πρόεδρος Μπαρόν θυμάται πώ ε, πρώτο ξεκινήσαμε. Αντί να αποδοθεί μεγάλη πολιτική σημασία στην πρώτη χαρτά θεμελιωδιών δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το DNA την αποκαλούσαμε τότε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώ αυτά συμβαίνουν καμιά φορά στην πολιτική. Λόγω τη θέση κάποιων κρατών μελών μην, μην τη δώσετε μεγάλη σημασία γιατί μετά θα έχουμε εσωτερικά προβλήματα. τελικά σε ένα διάδρομο της Νίκαιας εγκρίθηκε μπροστά από μια σημαία και υπέγραψαν κάποια αρχή και υπέγραψαν αρχή κρατών και κυβερνήσεων. Αλλά ο χρόνος απέδειξε ότι είχαμε δίκιο. Η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σήμερα είναι μέρος των συνθήκων, μέρος της συνθήκης της Λισαβόνας και χρειάστηκε να δώσουμε και άλλη μάχη, το θυμάται ο για να δημοσιευθεί ο δήλωση. Γιατί κάποιοι θέλησαν να υποσκάψουν την νομική και πολιτική σημασία της χάρτας. Σήμερα την έχουμε, φίσταται. Τι έγινε με τη χάρτα. Έπαθε αυτό που έπαθε και η συνθήκη της Λισαβόνας η χάρτα. Τόσο καιρό δώσαμε μάχες για την επικύρωση της ε, συνθήκης, λυσαλές μάχες. Πέντε χρόνια μας πήρε επικύρωση, πρώτα για τη συνταγματική συνθήκη, μετά για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Με αποτέλεσμα τελικά όταν ετέθησε ισχύ, σχεδόν χωρίς καν να το αντιληφθούμε πριν από μερικούς μήνες, η προσπάθεια που κάναμε για να πετύχουμε την επικύρωση της Λισαβόνας ήταν τόσο μεγάλη που τελικά ξεχάσαμε το περιεχόμενο της ηθίκης της Λισαβόνας. Παράδοξο θα σας φανεί αυτό, αλλά συμβαίνει πολλές φορές ε, στη ζωή. Δίνει κανείς μάχη για κάτι και μετά όταν το πετυχαίνει ε, ξεχαχανάει το επίτευγμά του. Σήμερα αυτό το παράδοξο ζούμε και το βλέπουμε σε θεσμικό επίπεδο. Η συνθήκη της Λισαβόνας επιφέρει εκβάθρων αλλαγές ε, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις θεσμικές ισορροπίες. Θα πρέπει να εξοικειωθούμε βεβαίως με τα νέα δεδομένα. Οι ήδη οι παίχτες δεν έχουν αντιληφθεί τις ε, αλλαγές που θα επιφέρει. Και να το συσχετίσω και με την πρωινή σας συζήτηση. De facto πλέον καταργούνται οι εκπεριτροπείς σαν ανά εξάμεινο. Αυτό είναι μεγάλη πολιτική σημασία. Τώρα πλέον αποκτάει νέο ρόλο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έχει μόνιμο πρόεδρο. Άρα αλλάζει η πολιτική δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πράξη καταργείται η εκπεριτροπή προεδρία. Και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι που δίνει πλέον την πολιτική κατεύθυνση τη Ένωση. Ταυτόχρονα το Συμβούλιο Υπουργών μετατρέπεται σε όργανο βασικά που θα είναι απλά συνομοθέτης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την εκτελεστική εξουσία σαφώς την έχει η Κομισιόν. Ευχαριστούμε την Κομισιόν με την ευκαιρία αυτή που οργανώνει αυτή τη διάσκεψη. Η Κομισιόν έχει μια μοναδική πολιτική ευκαιρία να παίξει ε, το ρόλο που της ανήκει. Οι ευκαιρίες είναι σαν τα τρένα ε, που περνάνε. Είτε το προλαβαίνεις είτε το χάνεις. Ε, και άμα χάσεις το πρώτο δεν ξέρεις πότε θα ξανάρθει το δεύτερο. Μιλάμε για μια ήσυχη επανάσταση που είναι Φώνα. Έχει μια χρυσή ευκαιρία η Κομισιόν να παίξει το ρόλο που θεωρούμε ότι θα πρέπει να παίξει εμεί οι φιλοευρωπαϊστέ. Και άμα δεν τον παίξει η Κομισιόν, θα τον παίξουν άλλοι στη θέση τη. Διότι πώ να το κάνουμε, ε, αυτά γίνονται στην πολιτική. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, λόγω της χρηματοπιστωτικής ύφεση, πώς θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτή την ύφεση. Είτε, είτε με περισσότερη Ευρώπη, είτε με λιγότερη Ευρώπη. Είτε με περισσότερη Ευρώπη, είτε με περισσότερα ε, κράτη-μέλη, εθνικά κράτη. Όταν μιλάμε για χρηματοπιστωτική εποπτεία, λέμε είτε το αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είτε το αναλαμβάνουν τα εθνικά κράτη. Ποιο είναι το δίδαγμα στο οποίο εγώ καταλήγω από την ύφεση. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εξελίξη εργασία και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Οπωσδήποτε θα έχουμε μελλοντικά περισσότερη υποπτία χρηματοπιστωτική, στι ε, ασφάλειε, στι αγορέ. Το πολιτικό στοιχείο θα είναι πιο σημαντικό κατά επόμενα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ότι τα τελευταία χρόνια. Και ποια είναι η συνέπεια όλων αυτών. Τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο, διότι για πολιτική μιλάμε. Δεν στέκει αυτό το επιχείρημα που τόσες φορές έχουμε ακούσει εδώ πέρα. Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αγορά. Έχει, έχει οικονομική σκοπιμότητα. Την έχει, αλλά όχι μόνο. Δεν είναι μόνο αγορά είναι και πολιτική ένωση. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε τις αξίες μας. Είναι το DNA των Ευρωπαίων αυτές οι αξίες. Εμείς ε, προερχόμαστε από μακρά παράδοση σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα πρέπει οπωσδήποτε αυτό να το λέμε και να το τονίζουμε. Έχει να παίξει το ρόλο της λοιπόν η χάρτα. Οι συμμετέχοντες στο πάνελ επίσης θα το αναφέρω σίγουρα. Το θέμα της μελλοντική προσχώρησης της Ένωσης στην ε, Σύμβαση της Ρώμης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει πρωτοπορήσει ανέκαθεν σε αυτό το με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το έχουμε και στο άρθρο 7 της τη Λισαβόνας Τεχνικέ δυσκολίε υπάρχουν και γι' αυτό βρίσκεστε εδώ πέρα για να μα βοηθήσετε. Τεράστιε τεχνικέ δυσκολίε. Η σύμβαση του Στρασβούργου απευθύνεται σε κράτη. Τα συμβαλόμενα μέρη είναι κράτη. Η Ένωση δεν είναι κράτο. Άρα, πώ προσαρμόζουμε τα όργανα και τι διαδικασίε τη σύμβαση στα δικά μα δεδομένα και ποιο θα έχει την εποπτεία της συμμόρφωση με τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα. Τα έχουμε δει και εδώ πέρα στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα. Ότι υπάρχουν πολλές τεχνικέ δυσκολίε. Λύσεις όμως υπάρχουν. Και ένα τελευταίο για να ολοκληρώσω, Πρόεδρε. Ζούμε σε μια στιγμή όπου η πολιτική καλείται να παίξει νέο ενισχυμένο ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι τάσει ε, τίνουν υπέρ ε, της περισσότερη Ευρώπης. Όσο περισσότερη πολιτική Ευρώπη έχουμε, το σημείο αναφοράς είναι αυτά τα δικαιώματα και ελευθερίες που προβλέπονται στην χάρτα. Όπως και εσείς αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερέφηνος που συμμετείχα στις εργασίες ε, για την κατάρτιση αυτή τη χάρτα. Ευχαριστώ πολύ. Η συντονιστρία, σας ευχαριστούμε για τα λόγια σας και το ζήλο σας. Ο κύριος Τσομπάνου Ντορντέα τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με τη σειρά μου να ευχαρίσω τους οργανωτές αυτής της διάσκεψης. Πολύ ευγενικό εκ μέρους τους που μας προσκάλεσαν και μας. Δυστυχώς η αντιπρόεδρος μας Βιβιάν Ρέντινγκ που έχει την αρμοδιότητα για την, ε, το χώρο αυτό δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας δυστυχώς δεν παρίσταται. Πάντως, ε, σαφώς και την ενδιαφέρει η μερισσίας διάταξη, καθώς και τα συμπεράσματά σας ε, την ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Να συνεχίσω τώρα στα αγγλικά. Θα ήθελα να δούμε το βαθμό στον οποίο η Κομισιόν ε, προσπαθεί να κρατηθεί στο ύψος της ατζέντα για την ηθαγένεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα που έχουν ε, σχεδιαστεί και που απορρέουν από την συνθήκη της Λισαβόνας και από το πρόγραμμα της Στοκχόλμης που υιοθετήθηκε το προηγούμενο Δεκέμβρη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η Κομισιόν όντως ε, κατανοεί ότι έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει που της δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας όπως ε, είπε και ο καθηγητής Δαβίγκο αλλά βέβαια η Κομισιόν ε, δεν έχει την ίδια ελευθερία έκφρασης ή δεν απολαμβάνει τον, της ίδιας ελευθερίας έκφρασης όπως η ακαδημαϊκή. Οπότε η δική μου παρέμβαση σήμερα θα είναι περιορισμένη. Θα περιοριστεί στη συζήτηση των πρωτοβουλειών που θα αναλάβει η Κομισιόν, που ανέλαβε τους προηγούμενους μήνες και ίσως και θα αναλάβει και τα επόμενα χρόνια. Να πω εξ αρχής ότι όλα τα στοιχεία για την ανάπτυξη ενός εκπόνηση μιας πολιτικής φιλόδοξης για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν με την θέση σε ισχύ της ε, Συνθήκης Λισαβόνας πέρσι τον Δεκέμβρη και βέβαια με τη Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση που γίνεται και νομικώ δεσμευτική. Δεύτερον, η προώθηση των, ανθρωπίνων των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι μία από τι ε, προτεραιότητε του προγράμματο τη Στοκχόλμη, σα το ανέφερα ήδη, το οποίο καθορίζει τι κατευθυντήριες γραμμέ, την ατζέντα για τι δράσει που πρέπει να αναλάβουν όλα τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα πέντε χρόνια στον τομέα τη ε, ελευθερία, ασφαλεία και δικαιοσύνη. Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν τις διαπραγματεύσει ένταξης ε, για την, ε, προσχώρηση για την, στην Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Συζητήσεις για το περιεχόμενο αυτό της εντολής για τις διαπραγματεύσεις ε, έχουν ξεκινήσει και διεξάγονται μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να συμβάλλει ώστε να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό μέσω μιας αυστηρής πολιτικής η οποία, την οποία θα υποβάλει η Κομισιόν στα μέσα του έτους, τον Ιούλιο δηλαδή. Η Επίτροπος Ρέντινγκ ήδη έχει παρουσιάσει κάποια βασικά σημεία κατά τη διάρκεια της διάσκεψης του Interlaken που έγινε από το Συμβούλιο της Ευρώπης για την μεταρρύθμιση της, του, ανθρωπίνου το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πέρσι το Φλεβάρι. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπερνά την, τα εσκαμμένα όταν, κάνει, όταν υποβάλλει δικαιοσύνη, όταν υποβάλλει προτάσεις, συγγνώμη. Το έχει πει και η ε, Αντιπρόεδρος η χάρτα θα είναι η πηξίδα για, όλη την, για όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το είπε και ο κύριος Μέντες Δεβίγκο, όντως πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η χάρτα και τα ανθρώπινα θεμελιώδη δικαιώματα θα περιλαμβάνονται στο DNA της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χάρτα θα αποτελέσει τη βάση για αυστηρές, πιο αυστηρές αξιολογήσεις επιπτώσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα αφορούν όλες τις νέες νομοθετικές προτάσεις. Δεύτερη προτεραιότητα, όχι μόνο της Κομισιόν, αλλά αν μου επιτρέπετε και όλης της Ένωσης, θα είναι να εξασφαλίσει ότι τα κείμενα που θα προκύπτουν από την νομοθετική διαδικασία θα συνάδουν με τη χάρτα. Θα είναι συλλογική ευθύνη όλων των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών να εξασφαλίσουν ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι και παραμένει συναφές με, με τα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της νομοθετικής. Και θα θυμάστε πριν από λίγα χρόνια ότι υπήρξαν κάποιες, κάποιες στην όλη διαδικασία. Κάποια σημάδια τα οποία μας, είπαν, μας έδειξαν ότι δεν υπήρχε απόλυτη συνάφεια μεταξύ της νομοθεσίας και της χάρτας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τρίτη προτεραιότητα, επίπεδο εφαρμογής στα κράτη-μέλη. Η χάρτα των, ανθρωπινών, των θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν εφαρμόζεται και δεν αφορά μόνο τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, αλλά και τα κράτη-μέλη, τα οποία την εφαρμόζουν ή εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε, που μα προσφέρει η συνθήκη, ώστε να εξασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τη χάρτα τη εθνική νομοθεσία, στην οποία θα ενταχθεί το ευρωπαϊκό δίκαιο. Όπω είπε η Επίτροπο Ρέντινγκ πολλές φορές, η, η Κομισιόν θα δείξει μηδενική ανοχή σε παραβάσει τη ε, χάρτα και όταν θα είναι αυτό απαραίτητο θα ξεκινήσει διαδικασία σε παραβάση. Ε, από αυτή λοιπόν την οπτική προσπαθούμε να αλλάξουμε έτσι λίγο την νοοτροπία της όλης διαδικασίας ε, παράβασης για αυτόν τον τομέα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο βασικός μας στόχος είναι να είναι πιο, όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά τα δικαιώματα που θα ε, υπάρχουν μέσα στην χάρτα για όλους τους ανθρώπους που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε να υπάρχει υψηλό επίπεδο αμοιβαίας εμπιστοσύνη στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, καθώς επίσης απαραίτητο και για την αξιοπιστία τη εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για να μπορέσουμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε αυτέ τι προτεραιότητε, η Κομισιόν θα προετοιμάσει και θα παρουσιάσει από το φθινόπωρο μια ετήσια έκθεση για το θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα επικεντρώνεται στη συμμόρφωση με τη χάρτα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο κρατών μελών. Στα πλαίσια βέβαια και των αρμοδιοτήτων ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η, αίτηση, η έκθεση θα είναι μια μεθοδολογική έκθεση, η πρώτη. Η έκθεση αυτή θα δίνει πληροφορίε για το τι έχει γίνει από την Κομισιόν, για την εφαρμογή τη πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στα πλαίσια των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει στα πλαίσια της ελευθερίας δικαιοσύνης και ασφάλειας. Και η έκθεση επίσης θα δείχνει ποιες είναι οι βασικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης θα δώσει μια ευκαιρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να έχουν μια ετήσια συζήτηση για το τι έχει γίνει στους τομείς όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητες να δράσει και τι θα πρέπει να γίνει στο μέλλον έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα ε, εφαρμοστεί ε, αποτελεσματικά η χάρτα. Η Κομισιόν θα εργαστεί ε, ώστε να προετοιμάσει αυτή την έκθεση σε συνεργασία με τα κρατημέλη, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να παρερμηνεύσουν την προσπάθεια της Κομισιόν για να συμβάλλει στην, ε, πολιτική, στην εκπόνηση πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην, ε, σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Δεν υπάρχει ε, κανένας, ε, δεν υπάρχει καμία ανάγκη να υπάρξει νέα επιπλέον νομοθεσία. Το θέμα είναι να δώσουμε μια κατεύθυνση στην ε, πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να την καταστήσουμε κομμάτι όλων των πολιτικών και να, την, να διορθώσουμε πράγματα ίσως που ήδη υπάρχουν στο κεκτημένο και κυρίως προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε πλήρη συμμόρφωση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας με τη Χάρτα. Επίσης προσπαθούμε να βελτιώσουμε την εφαρμογή επιτόπου στα πλαίσια του ευρωπαϊκού δικαίου για την επίλυση των πραγματικών ε, προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ως προς το θέμα αυτό οι πολίτες μας. Η προσπάθεια λοιπόν όλη αυτή που γίνεται για την εκπόνηση πολιτικής σε επίπεδο ευρωπαϊκό έχει να κάνει και με την ε, σωστή λειτουργία μιας ε, ε, διευρυμένης και διαφοροποιημένης ένωσης έτσι ώστε να, να διατηρήσουμε την ισχύ της ένωσης που νομίζω ότι θα πρέπει να είναι και ο στόχος μας για να μπορέσουμε να ενοποιήσουμε την πολιτική συνοχή της πρέπει να εξασφαλίσουμε μεταξύ άλλων ένα υψηλό επίπεδο αμοιβαίας εμπιστοσύνη που θα βασίζεται σε μια δέσμευση για την προώθηση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων που θα αντικατοπτρίζει πλήρως τις αξίες πάνω στις οποίες βασίστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενοποίηση της αμοιβαίας ε, εμπιστοσύνη μεταξύ δικαστικών και αστυνομικών αρχών είναι προαπαιτούμενο για να έχουμε έναν ισχυρό χώρο ασφάλειας δικαιοσύνης και ελευθερίας. Τέλος, η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση για τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι υψή της πολιτικής σημασίας και νομικής σημασίας. Θα αγγίθει ότι οποιοδήποτε θύμα δράσης που λαμβάνεται στα πλαίσια των ευρωπαϊκών αρμοδιοτήτων θα μπορεί να αναφερθεί ενώπιον του δικαστηρίου στο Στρασβούργο με τις ίδιες συνθήκες που εφαρμόζονται για όλους όσους ε, υποβάλλουν ε, ε, εφέσεις στο δικαστήριο. Οπότε επανεπιβεβαιώνουμε τον σημαντικό ρόλο που έχει να παίξει το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την προστασία αυτών σε όλη την Ευρώπη. Η προσχώρηση στην σύμβαση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί μεμονωμένη πρωτοβουλία, αλλά ως ακόμα μία πρωτοβουλία, ώστε να υπάρξει μία φιλόδοξη πολιτική ευρωπαϊκή για να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των οποίων πρέπει να απολαμβάνουν οι πολίτες της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα έχει λιγότερες ε, πιθανότητες να παρέμβει σε θέματα που άπτονται του ευρωπαϊκού δικαίου, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν, ε, είναι, ε, δεν είναι υπόλογη όταν εκπονεί ε, πολιτική. Τώρα, αλλάζω λίγο απότομα θέμα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Πάμε στην ε, ιθαγένεια, την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, Στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της 3ης Σεπτεμβρίου 2009 ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Χωσέ Μανουέλ Μπαρόσο, τόνισε την ανάγκη που υπάρχει να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή ηθογένεια και τη συμμετοχή, δίνοντας όντως υπόσταση στα δικαιώματα των πολιτών. Η συνθήκη της Λισαβόνας ε, παρουσίασε πολλά, ε, μια δέσμη μέτρων που ενισχύουν την ε, δράση του ως και την δημοκρατική συμμετοχή. Καταρχήν, αναγνωρίζει το δικαίωμα των πολιτών να συμμετέχουν στην, στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης. Δεύτερον, ο διάλογος με την κοινωνία των πολιτών ε, γίνεται μια γενική αρχή που ισχύει σε όλες τις ε, σφαίρες της κοινωνικής ζωής και, αποτελεί τα, και περιλαμβάνει τα βασικά πρότυπα πάνω στα οποία πρέπει να βασίζονται. Ε, επίσης δημιουργεί μια δέσμη δικαιωμάτων που, των οποίων απολαμβάνει κάποιο που έχει την ε, ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Η Κομισιόν δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει όλες τις πιθανότητες, δυνατότητες που έχει από την συνθήκη για να δώσει στους ε, πολίτες βήμα και να δημιουργήσει μια πιο ανοιχτή, έναν πιο ανοιχτό χώρο, έναν ευρωπαϊκό δήμο. Μία από τις βασικές πρωτοβουλίες ήταν η πρόταση που παρουσιάστηκε στις, 20, στις 31 Μαρτίου για την ε, πρωτοβουλία των πολιτών που έχει ως ε, στόχο να δημιουργήσει τις συνθήκες που θα είναι απλές, θα είναι φιλικές προς το χρήστη, θα είναι προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εξασφαλίζει ότι αυτός ο μηχανισμός θα παραμείνει αξιόπιστος και δεν θα τύχει κατάχρησης. Οι συζητήσεις για την πρόταση αυτή έχουν προχωρήσει όπως ξέρετε, οπότε ελπίζουμε ότι αυτός ο μηχανισμός ε, θα ξεκινήσει να λειτουργεί σύντομα. Τα νέα αυτά εργαλεία που προσφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας θα είναι, αποτελεσμα... Ε, σημαντικά έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή και να, είναι πιο... να έχει περισσότερο νόημα η ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Επίσης, τα δικαιώματα που ήδη ισχύουν θα πρέπει να ενισχυθούν και να διευρυνθούν παραμένει ένα κενό μεταξύ των εφαρμοστέων ε, κανόνων και της πραγματικότητας. Οι πολίτες αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ε, ζωή, ειδικά σε θέματα διασυνοριακά που εμάς μας ενδιαφέρουν, ε, με πολλά, αντιμετωπίζουν πολλά προσκόμματα. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο φάσμα πρωτοβουλειών ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η προσβασιμότητα σε αυτά τα δικαιώματα. Και θα τονίσω μερικά για να σας δώσω έτσι μια γεύση του τι γίνεται και τη σημασία που αποδίδεται σε αυτά τα θέματα. Είναι σημαντικό οι πολίτες να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και τις ε, ε, δυνατότητες που έχουν. Η Κομισιόν λοιπόν θέλει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των πολιτών ως προς τα δικαιώματά τους και πώς μπορούν να τα χρησιμοποιούν πλήρως. Στα πλαίσια αυτά, ο πρόεδρος Μπαρόσο έχει ζητήσει από την αντιπρόεδρο Ρέντινγκ να ηγηθεί της ε, προσπάθειας ε, ε, για την παρουσίαση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους πολίτες. Δεύτερον, και των επιπτώσεων αυτών στους πολίτες. Δεύτερον, πρέπει να δούμε και, τις, άμεσα, και τα άμεσα και τα έμεσα προσκόμματα που δημιουργούνται από τα εθνικά όρια όταν οι πολίτες προσπαθούν να εξασκήσουν τα δικαιώματά τους και να αναλάβουμε δράσεις έτσι ώστε να αποφύγουμε τα προσκόμματα αυτά, να τα απαλείψουμε. Αυτό θα γίνει σε απάντηση και της έκθεσης Λαμασούρ, που δημοσιεύτηκε πριν από δύο χρόνια, και της πιο πρόσφατης έκθεσης Μόντι για τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς. Ως προς αυτό λοιπόν, και προ αυτόν τον σκοπό, η Κομισιόν τον προηγούμενο μήνα ξεκίνησε μια δημόσια διαβούλευση που επικεντρώνεται στο πώ τα δικαιώματα ηθαγένεια μπορούν να ενισχυθούν και να ολοκληρωθούν. Είναι λοιπόν ουσιώδε να υπάρξει η πιο ευρεία συμμετοχή ε, αρχών, ε, ακαδημαϊκών, κοινωνίας των πολιτών, πολιτών, μεμονωμένων, ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν, να δώσουν τις απόψεις τους, να συμβάλλουν με τις ιδέες τους. Στα πλαίσια αυτά, ελπίζουμε να επωφεληθούμε και από την εμπειρογνωμοσύνη όλων των α, συμμετεχόντων στην σημερινή διάσκεψη. Αργότερα, τον Οκτώβρη του τρέχοντος, η Κομισιόν θα υιοθετήσει μια, μια ανακοίνωση για, την, ε, για τον ορισμό ε, ε, της ηθαγένειας θα σημειώσουμε τι έχει γίνει, αλλά θα τονίσουμε και ποια είναι τα μέτρα που προτιθέμεθα να λάβουμε, έτσι ώστε να ενισχύσουμε του πολίτε για να μπορούν να απολαμβάνουν των δικαιωμάτων του πλήρω. Θα παρουσιάσουμε επίση έναν οδικό χάρτη για το πώ αυτό θα γίνει εφικτό. Ο νέος αυτός ε, στόχος λοιπόν θα είναι να εξασφαλίσουμε ότι σε όλες τις πτυχές της καθημερινής τους ζωής οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν, να εξασκήσουν τα, ευρωπαϊκά, τα δικαιώματά τους ως Ευρωπαίων πολιτών όπως χρησιμοποιούν και εξασκούν τα δικαιώματά τους ως ε, πολίτες του κράτου, του έθνους τους. μια, ένα γενικότερο θέμα στην προσέγγιση της Κομισιόν ε, και για την εκπόνηση των, ε, της πολιτικής για, την, ε, για τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ηθαγένεια είναι να έχει πολιτικές που θα, που θα έχουν ως στόχο τα, τις ανάγκες και τα δικαιώματα των πολιτών. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν ένας διάλογος και στενότερη συνεργασία και σε τοπικό και σε περιφερειακό, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ όλων των συσχετιζόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικών εταίρων και της, των τοπικών, της κοινωνίας των πολιτών και των ακαδημαϊκών. Πρέπει να σκεφτούμε και να συζητήσουμε πώς αυτός, αυτή η νέα καινοτόμα πτυχή της ε, ευρωπαϊκής τεθαγένειας θα μπορέσει να δώσει αυτά αποτελέσματα για τους πολίτες και πώς η, ε, η κοινωνική καθημερινότητα αλλάζει. Βασισμένη λοιπόν σε αυτά που είπε η κυρία Ντελαροσέρ, πρέπει να έχουμε διεθνικές συζητήσεις για το πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα στα πλαίσια των αθεμελίων δικαιωμάτων. Οι προκλήσεις για τη δική μας την ε, κουλτούρα με βάση τι ε, εμπειρίε που έχουμε από τη δική μα την κουλτούρα και οι οποίε ε, ε, προκύπτουν από την εξέλιξη των ηθών, από τι διαδικασίε που ξεκινούν από την παγκοσμιοποίηση, από τα μεταναστευτικά, τις μεταναστευτικές ροές, από τις μοντέρνες τεχνολογίες, από ασύμετρε απειλέ, όπω τρομοκρατία ή από την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση. Όλε αυτέ οι προκλήσει που σε μεγάλο βαθμό είναι φυσικέ, έχουν τρομακτικές συνέπειες και σε πολιτικέ στις πολιτικές ε, θέσεις ε, και στις, στην, στην ε, διαχείριση που, την οποία αποφασίζουν να λάβουν διάφορες αρχές για προβλήματα που προκύπτουν και για περιπτώσεις τέτοιες. Πρέπει λοιπόν από κοινού να το σκεφτούμε, να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε καινούρια νοοτροπία που θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Θα είναι μακρόπνοες αντί να, κάνουμε, να δίνουμε ad hoc λύσεις, όπως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια αρκετές φορές. Και επίσης πρέπει να αξιολογήσουμε το βαθμό στον οποίο επηρεάζονται οι, αξία, οι αξίες μας, θεμητά ή όχι, από τέτοιες νέες τάσεις. Οι καθηγητές Jean Monnet έχουν, ε, είναι, ε, έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να συζητήσουν ε, δημοσίω τα θέματα αυτά και θα παίξουν σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά τα θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων και ηθαγένειας. Είναι λοιπόν μεγάλες οι προκλήσεις που μας περιμένουν, αλλά έχουμε και πολλές ευκαιρίες μπροστά μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Διότι μας παρουσιάσατε τις προθέσεις της Επιτρόπου, κυρίας Ρέντινγκ, Όταν δει κανείς τους τομείς ε, όπου η Κομισιόν έχει την πρόθεση να παρέμβει, βλέπει κανείς ότι υπάρχει τεράστια προοπτική. Θα αλλάξουμε τώρα οπτική και θα δώσουμε το λόγο στους πανεπιστημιακούς και θα καλέσω την κυρία Ελίζαμπεθ Κίλτ, εδραζόμενη στο Πανεπιστήμιο της Νιτμέγ ε, και καθηγήτρια οικονομικών στο London School of Economics, να πάρει πρώτο το λόγο. Σας ευχαριστώ. Είναι ιδιαίτερη η τιμή που είμαι σήμερα μαζί σας ε, και μιλώ για ένα τόσο σημαντικό θέμα και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους την ομάδα Ζόμονε για την πρόσκληση και να τονίσω τη σπουδαιότητα του προγράμματος Ζόμονε ως ξεχωριστό αλλά και θεμελιώδες σκέλος της πανοπλίας των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης διότι ε, συγκεντρώνει τους ε, διάφορους πανεπιστημιακούς ε, και τους βοηθά να καταλάβουν το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας έρθουμε στο θέμα μας θεμελιώδη δικαιώματα και ε, ενουσιακή ηθαγένεια. Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς αυτή τη στιγμή την πλήρη, το πλήρες νόημα και τον αντίκτυπο που θα έχει η συνθήκη της Λισαβόνας στα θεμελιώδη δικαιώματα και την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι γι' αυτό. Πρώτον, η ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, απέκτησε τα πλήρη της δικαιώματα στα πλαίσια μιας νομικά δεσμευτικής χάρτας. Ο σκελετός της ηθαγένειας αυτής τώρα αποκτά ε, σάρκα και οστά ώστε να αποκτήσει την πλήρη του σημασία. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων προβλέπει και την ηθαγένεια διότι επανακαθορίζει και ε, ε, ορίζει ένα, μια δέσμη δικαιωμάτων για τους ε, υπηκόους. Η Ευρωπαϊκή χάρτα των θεμεσιλιωδών ε, δικαιωμάτων δεν είναι ένα ε, μέρος ε, των θεσμικών κειμένων, ούτε διεθνές όργανο όπως ας πούμε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο νέος μηχανισμός για την τήρηση των δικαιωμάτων μετατρέπει τη σχέση μεταξύ των ατόμων και του κράτους μέσα από ένα διαφορετικό πακέτο δικαιωμάτων που εδρεύουν, που, που καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην παρουσίασή μου θα παρουσιάσω μία από τις, κάθε, κάθε, μία από αυτού, κάθε έναν από αυτούς τους λόγους για τα θεμελιώδη δικαιώματα και ε, τα, την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Τρία είναι τα βασικά στοιχεία. Το να είναι κανείς πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πιο ελκυστικό πλέον σε υπηκόρους των κρατών μελών, διότι τα δικαιώματα, τα οποία, στα οποία δεν θα είχαν δικαιώματα, θα μπορούν να τα απολάβουν μέσα από την εθνική τους, ε, για να απολάβουν αυτόν μέσω της εθνικής τους υπηκότητας, μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση σε αυτά μέσω της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Καθορίζοντας σε μία χάρτα ποιος έχει δικαιώματα, ποιος έχει δικαίωμα να απολάβει αυτά τα δικαιώματα, διευρύνει το σύνολο των ε, κατόχων των δικαιωμάτων, οπότε περιλαμβάνονται όχι μόνο οι πήκοοι άλλων κρατών μελών, ακόμη και αυτούς που υπόκεινται σε μεταβατικές ρυθμίσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων, αλλά επεκτείνεται και σε υπηκόους τρίτων χωρών. Τρίτον, τα δικαιώματα αυτά δεν εξαρτώνται πλέον είτε σε εθνικές ρυθμίσεις ή συνταγματικές ρυθμίσεις είτε σε συνθήκες διεθνούς εμβέλειας με όλες τις ε, δυσκολίες που συνδέονται με την πρόσβαση στα δικαιώματα. Μπορούν πλέον τα άτομα να τα χρησιμοποιήσουν με την υποστήριξη ε, των κρατών μελών και την ε, δέσμευση καλής πίστης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα παρουσιάσω τώρα τις βασικές πτυχές ε, της Χάρτας Θεμελιωτών Δικαιωμάτων και στη συνέχεια θα δω πώς αλλάζουν, αλλάζει η έννοια της ε, υπηκότητας. Η, η ε, Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθετήθηκε από τους τρεις θεσμικούς φορείς το 2000. Η Σύμβαση είναι πραγματικά εξαιρετικό επίτευγμα και όπως όλα τα μεγάλα γεγονότα συνοδεύονται και ε, από αντίλογο και συζήτηση. Ε, η χάρτα κωδικοποιεί τα δικαιώματα των οποίων ήδη απολάβουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και ε, δεν υπήρχε αρχικά ο στόχος να διευρυνθούν, αλλά οποιαδήποτε δράση όμως για την εδραίωση δικαιωμάτων που ήδη έχουν τα άτομα από τη στιγμή που μπαίνουν σε ένα έγγραφο δημιουργεί μία φυγόκεντρο δύναμη προς ε, τα δικαιώματα, των, ε, τα δικαιώματα αυτά. Το να μπορεί κανείς δηλαδή να ε, θεμελιώνει κάποια δικαιώματα για να μπορεί να έχει πρόσβαση και σε άλλα εμφανίζει ακριβώς αυτή την, αυτή την προσπάθεια. Η χάρτα δεν συμπεριελήφθηκε στις τροποποίησεις της συνθήκης αλλά ε, από το 2000 μέχρι σήμερα αυξήθηκε η σπουδαιότητά της μέχρι σήμερα που εντάχθηκε στην ένωμη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις πολιτικές συζητήσεις γινόταν λόγος για τη χάρτα αυτή και από τους δικαστές των κρατών μελών και έτσι σιγά σιγά απέκτησε μεγαλύτερη σημασία και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καθότι ο ε, Γενικός Εισαγγελέας άρχισε να στηρίζεται σε αυτήν. Παρ' όλα αυτά όμως έμεινε εκτός νομικών δεσμευτικών, νομικός δεσμευτικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν ε, πολύ λίγο ικανοποιητική η κατάσταση αυτή και για τα κράτη-μέλη και για τους χρήστες, για πολλούς λόγους. Θα παρουσιάσω κάποιες από αυτές. Πρώτον, τα κράτη-μέλη χρειάζονται εμπιστοσύνη, ότι δηλαδή οι εθνικές τους ρυθμίσεις, συνταγματικές ρυθμίσεις δεν θα υποσκαφθούν από κοινοτικής φύσεως μέτρα λόγω της έλλειψης ε, συνολικών διατάξεων σε Ευρωπαϊκή Ένωση που να καλύπτουν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα ενιαίο έγγραφο το οποίο να ορίζει ποια δικαιώματα υπάρχουν δυνάμει του κοινοτικού δικαίου ώστε να είναι ξεκάθαρο και για τις αρχές των κρατών μελών και για τους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεδομένου ότι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα εργαλείο επιβολής και εφαρμογής των δικαιωμάτων αυτών, το οποίο δεν θα είναι εις βάρος των ε, ατόμων. Η επέκταση του, του χώρου ελευθερίας και δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δείχνει ότι χρειάζεται ε, ένα εργαλείο που να υποδεικνύει την, πώς θα συντάσσεται η νομοθεσία σε αυτό το τομέα. η σύσταση, η σύνταξη των νομικών κειμένων προβλέπουν τα θεμελιώδη δικαιώματα αλλά, ε, μέχρι στιγμής στο προήμιο, αλλά στο μέλλον θα πρέπει να ορίζεται αυτό ξεκάθαρα ώστε οι, ε, οι πολίτες να έχουν γνώση των δικαιωμάτων των οποίων, τα οποία μπορούν να επικαλεστούν. και βεβαίως δεν πρέπει ε, οι διατάξεις που υπάρχουν σε διεθνείς ε, συμβάσεις να υποσκαφθούν από το ε, από μια κοινοτική εμβέλεια συνθήκη. Τι σημαίνει ο θεμελιώδη χάρτα. Καθορίζει ένα χάρτη δικαίων σε 7 κεφάλαια που έχουν τον αντίστοιχο τίτλο, δηλαδή αξιοπρέπεια, ελευθερίες, ισότητα, αλληλεγγύη, δικαιώματα των πολιτών, δικαιοσύνη και γενικές διατάξεις μεταξύ των νομικών έγινε μεγάλη συζήτηση ε, αν τα διάφορα κεφάλαια θα έχουν διαφορετικές νομικές επιπτώσεις. Και βέβαια αυτή η συζήτηση θυμίζει τις συζητήσεις για το φύλλο των αγγέλων Έχω την εντύπωση ότι ε, η ανάγνωση της χάρτας και η εξέταση των γενικών διατάξεων που μας καλεί να κάνουμε η συνθήκη της Λισαβόνας δεν υπάρχει λόγος να θεωρήσουμε ας πούμε ότι οι διατάξεις που υπάρχουν στο κεφάλαιο περί αξιοπρέπειας είναι νομικώς διαφορετικές από αυτές που υπάρχουν στα άλλα κεφάλαια. Για παράδειγμα, το άρθρο 2 το οποίο βρίσκεται στο κεφάλαιο αυτό αφορά το δικαίωμα στη ζωή και αντικατοπτρίζει αντίστοιχε διατάξεις στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και το ΔΕΚ δεν ε, ε, αμφισβήτησε ποτέ το δικαίωμα αυτό και το ε, ερμήνευσε πολλές φορές σε πολύπλοκες και ευαίσθητες υποθέσεις. Καθορίζει λοιπόν ένα πακέτο δικαιωμάτων ανεξάρτητα από το σε ποιο κεφάλαιο έχουν τοποθετηθεί. Τα δικαιώματα που υπάρχουν στη χάρτη προέρχονται από δύο πηγέ κυρίω. Δικαιώματα τα οποία ήδη υπήρχαν στο κοινοτικό δίκαιο, α πούμε για τους πολίτες τη Ευρωπαϊκή Ένωσης, το δικαίωμα ελεύθερη κυκλοφορίας και στην ε, Ευρωπαϊκή Σύμβαση ε, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τα πρωτόκολλα, η οποία ορίζει ότι ε, στο βαθμό που περιλαμβάνει δικαιώματα τα οποία αντιστοιχούν αυτών της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η εμβέλεια αυτών θα είναι η ίδια με αυτή που προβλέπεται στην ε, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όμως αυτή η διάταξη δεν εμποδίζει το κοινοτικό δίκαιο να προβλέψει και ευρύτερε διατάξεις. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι το πεδίο του άρθρου 7 της χάρτας, το δικαίωμα ε, σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωή, θα πρέπει να πηγαίνει τόσο μακριά όσο τουλάχιστον το έχει ορίσει η απόφαση του, του στις 12 Ιανουαρίου του 2010 στην υπόθεση Γκίλαν κατά του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, δηλαδή οι αστυνομικοί δεν μπορούν να σταματήσουν κάποιον ε, για να ε, τον ερευνήσουν διότι αυτό έρχεται σε, παραβιάζει την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή. Υπάρχει και μια απόφαση του Δεκεμβρίου, 4η Δεκεμβρίου του 2009 που έχει σαφείς επιπτώσεις για τις εξελίξεις στον τομέα ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας η, απόφαση ότι βρήκε ότι η βάση δεδομένων DNA του, της Βρετανικής αστυνομίας ε, περιελάμβανε στοιχεία ατόμων τα οποία δεν ήταν ποτέ καν ύποπτα για εγκληματικές επιθέσεις και αυτό ήταν παράβαση της ιδιωτικής ζωής. Ε, κάποιες παρεμβάσεις που ακούσαμε σήμερα το πρωί ε, ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσουν εάν οι αρχές ενός κράτους μέλους μπορούν να δώσουν πληροφορίες γρήγορα από δημόσιες αρχές άλλου κράτου μέλους χωρίς να χρησιμοποιήσουν καταναγκαστικά μέτρα ή χρήση ή μέτρα που έχουν προκύψει από αντίστοιχες αρχές άλλου κράτους μέλους. Το θέμα του πώς μπορεί να επιταχυνθεί η αστυνομική συνεργασία ώστε να καλυφθεί η οποία ασυμβατότητα των συστημάτων πληροφορικής ε, και επέκταση θα πρέπει να συναχθούν και τα σχετικά αποτελέσματα. Κατά την διενέργεια αυτών των δραστηριοτήτων, η Κομισιόν θα πρέπει να λάβει υπόψη την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διασφαλίσει ότι οι δράσεις της δεν θα ενθαρρύνουν ούτε θα δικαιολογούν ε, παραβιάσεις κατά της ε, ιδιωτικής ζωής των ατόμων, λήψη δειγμάτων ή ε, όπου και η κατοχή αυτών των δειγμάτων αντίκειται στο άρθρο 7 της χάρτας. Το δεύτερο σημείο που θέλω να κάνω στην παρουσίασή μου είναι το εξή. Η χάρτα δεν περιορίζεται στο πεδίο εφαρμογής μόνο στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λίγες από τις διατάξεις έχουν αυτό τον περιορισμό στους υπηκόους και αυτό μόνο στο κεφάλαιο 5. Ε, ειδικά περιορισμένους τους ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το δικαίωμα ψήφου και η συμμετοχή στις εκλογές για το κοινοβούλιο ε, στα κράτη-μέλη όπου κατοικεί ο πολίτης. Ε, το στοιχείο για την ελεύθερη κυκλοφορία, τη διπλωματική και προξενική προστασία είναι μόνο δικαιώματα για τους πολίτες. Αλλά ακόμη και σε ένα κεφάλαιο που έχει τον πολίτη ως τίτλο υπάρχουν πολύ σημαντικά δικαιώματα τα οποία αφορούν οποιονδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε είναι υπήκοοι, είτε είναι υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτους μέλους ή είναι υπήκοοι τρίτων χωρών. Για παράδειγμα, το άρθρο 41 έχει ένα δικαίωμα για την σωστή διακυβέρνηση. Είναι στο κεφάλαιο για τα δικαιώματα του πολίτη, αλλά λέει ότι ο καθένα έχει το δικαίωμα ε, να τύχει ε, ε, σωστή και δίκαιη διεκπαιρέωση των υποθέσεων και μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα από του φορεί τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, οποιοδήποτε εδώ σημαίνει οποιοδήποτε, όχι μόνο πολίτη, αλλά οποιοδήποτε κατοικεί τακτικά στην επικράτεια ενό κράτου μέλου κατά λιγότερο τακτικά διαστήματα που είναι παρόν στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου, εάν οι υποθέσεις του απαιτούν δράση από μια κοινωτική αρχή. Οι φορείς ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνουν και τις αρχές των κράτους μέλους που διεκπεραιώνουν το κοινοτικό δίκαιο. Έτσι δηλαδή, ο ετών άσυλος σε ένα κράτος ε, μέλος έχει δικαίωμα να στηριχτεί στο άρθρο 41 της Χάρτας για να ζητήσει ε, η αίτησή του να αντιμετωπιστεί και να διεκπεραιωθεί με, τον, με δίκαιο τρόπο σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, διότι η αίτηση ε, ασύλου θα πρέπει να διεκπεραιώνεται σύμφωνα με την δευτερογενή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η T.H. Marshall, ε, η Βρετανή κοινωνιολόγος, η οποία δραστηριοποιήθηκε στο δεύτερο ήμιση του 20ου αιώνα, δίνει μια σημαντική αφετηρία για να καταλάβουμε την έννοια τη υπηκότητα. Το έργο του μάλλον ήταν, ε, είχε ιδιαίτερη επιρροή, διότι δίνει έναν τρόπο σκέψης για την υπηκότητα, ο οποίο ε, ξεφεύγει από τι μη ικανοποιητικέ ιδέες για το φύλλο και το έθνο, τα οποία ε, κυριάρχησαν στο 19ο αιώνα. Σύμφωνα με τον Μάρσαλ, η υπηκότητα περιγράφει μια διαδικασία δεσμών και δικαιωμάτων ε, για τους ανθρώπους. Ω άτομα τα οποία βρίσκονται σε μια επικράτεια και κάτω από μια αρχή και ισχυρίζονται ε, ότι έχουν κάποια, κάποιες δέσμες δικαιωμάτων, αναγνωρίζουν έτσι την έννοια της υπηκότητας και στο έργο το οποίο αφορούσε το Ηνωμένο Βασίλειο ε, εξέτασε πως τα αστικά δικαιώματα τα οποία αποκτήθηκαν στους αγώνες του 18ου αιώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθήθηκαν από πολιτικά δικαιώματα του 19ου αιώνα με βαθμιακή επέκταση της ε, γενικής ε, δικαιώματος ψήφου και κατέληξαν σε πλήρη δικαιώματα τον 20ο αιώνα. Έτσι λοιπόν μπορούμε να δούμε ότι τα δικαιώματα τα οποία αποκτήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρασαν μέσα από τις συνθήκες επεκτάθηκαν και σήμερα βρίσκει κανείς ε, διάφορα δικαιώματα για την εργασία και τη δυνατότητα να μετακινείται και να ζει κανείς οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τα πολιτικά δικαιώματα και πιο πρόσφατα τα κοινωνικά δικαιώματα οπουδήποτε πάει το άτομο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα οι υπήκοοι τρίτων χωρών απολαύουν δικαιώματα Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω πολλών μέσων τα οποία έχουν εγκριθεί, τα οποία περιλαμβάνουν την οδηγία για τους ε, υπηκόους τρίτων χωρών που είναι μακράς διαρκείας διαμένοντες, που προβλέπουν ε, ένα δικαίωμα ασφαλούς διαμονής και ελεύθερη κυκλοφορία για οικονομικούς και άλλους λόγους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον οι υπήκοοι τρίτης χώρας έχουν περάσει πέντε χρόνια ε, νόμιμης διαμονής σε ένα κράτος μέλος. Ε, η ενοποίηση, η επανένωση οικογενειών, είναι το δικαίωμα σε υπηκόους τρίτων χωρών να ζήσουν με την οικογένειά τους. Οι φοιτητές, ερευνητές και σχετικές οδηγίες προβλέπουν ότι θα μπορούν ε, ε, να εισέρχονται και να διαμένουν υπήκοοι τρίτων χωρών κλπ. Η ε, απέλαση υπηκών τρίτων χωρών θα τεθεί τώρα στη χάρτα. Το δικαίωμα δηλαδή του ατόμου για σεβασμό της ιδιωτικής και κοινωνικής ε, και οικογενειακής του ζωής ε, πολλές φορές από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κρίθηκε ότι είναι ένα δικαίωμα για την προστασία κατά της απέλασης. Αυτή η νομολογία πρέπει να ισχύσει και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο μέσω της ε, χάρτας. Ήδη μέσα στην δευτερογενή νομοθεσία για τους υπηκόους τρίτων χωρών είναι σαφές ότι αυτοί αποκτούν δικαιώματα σύμφωνα με την έννοια της υπηκότητας που έχει υπηρετήσει ο Μάρσαλ. Σχεδόν όλα τα δικαιώματα που υπάρχουν στη χάρτα ισχύουν όχι μόνο για του υπηκόου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε υπηκόου τρίτων χωρών. Αυτοί αποκτούν δέσμε δικαιωμάτων μέσα από τη χάρτα ε, με τρόπο που παρομοιάζεται με αυτόν του τρόπου σκέψη ε, του Μάρσαλ σχετικά με το κομβικό νόημα τη ε, υπηκότητα. Θα μπορούσε να πει κανεί ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δικαιούνται να ενεργοποιήσουν την υπηκότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από την άσκηση των δικαιωμάτων της και έτσι σιγά σιγά η διαφορά μεταξύ των δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών τρίτων χωρών έχει περιοριστεί και υπάρχει μια εξισορρόπηση των δικαιωμάτων. Η μετατροπή των δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τη χάρτα ε, θεωρούσαμε ότι είχαμε ένα ε, συνταγματικό πακέτο δηλαδή όχι μόνο ένα μηχανισμό με τον οποίο καθορίζεται και ε, επιτελείται η διακυβέρνηση, αλλά έχουμε και ένα Bill of Rights ε, που είναι μέρος των εθνικών συνταγμάτων και επομένως είναι ε, καθήκον των κρατικών αρχών να το προστατεύουν. Οι αρχές πέρα από το κράτος μπορεί να μην ε, συμπίπτουν ή να συμπίπτουν με ένα εθνικό κανόνα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με την υποχρέωση να, τηρεί, ε, τον, ε, να τηρούνται τα δικαιώματα. Εναλλακτικά, σύμφωνα με τις, ε, μετά από τις ελλείψεις του συνταγματικών συστημάτων να προστατεύσουν τα άτομα σε πολλά μέρη της Ευρώπης, όπως τονίστηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αναπτύχθηκαν διάφορα ανθρώπινα δικαιώματα σε διάφορα στάδια και το κράτος αναλαμβάνει να τηρήσει και να διασφαλίσει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία υπάρχουν στην ε, διεθνή συνθήκη για οποιονδήποτε υπόκειται στην δικαιοδοσία του κράτους. Ο μηχανισμός για τον καθορισμό του περιεχομένου των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στις συνθήκες είναι πρώτα οι εθνικές διοικήσεις οι οποίες μπορεί να έχουν διαφορετική ερμηνεία σχετικά με το περιεχόμενο και την έκταση κάποιων δικαιωμάτων. Δεύτερον, τα εθνικά δικαστήρια αποφασίζουν ποια είναι, ποιο είναι το νόημα μιας διεθνούς συνθήκη στα πλαίσια των δράσεων των εθνικών ε, διοικήσεων και ορισμένες φορές ε, υπάρχει και ένα δικαστήριο, όπως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο δημιουργήθηκε και το οποίο ουσιαστικά οποιοδήποτε άτομο θεωρείται ότι έχουν ε, πληγεί τα δικαιώματά του μπορεί να προσφύγει όταν έχει εξαντλήσει όλες τις άλλες δυνατότητες. Όμως η χάρτα δεν είναι ούτε εθνικό, ε, εθνική συνθήκη, ούτε συνθήκη διεθνούς εμβέλειας. Είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιούργημα και εξαρτάται για την εφαρμογή και την την ερμηνεία από τους μηχανισμούς του ευρωπαϊκού δικαίου και υπ' αυτή την έννοια επιβάλλει υποχρεώσεις στις κρατικές αρχές οι οποίες δεν μπορούν ε, να ε, υποστούν τροποποίησης. Η τελική τους ερμηνεία είναι δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου προς το οποίο μπορεί να προσφύγει οποιοδήποτε εθνικό δικαστήριο για ερμηνεία. Αυτή η ερμηνεία όμως όταν παρέχεται είναι δεσμευτική και για τις εθνικές διοικήσεις σε όλα τα κράτη-μέλη και τα εθνικά δικαστήρια. Εάν ξεκινήσουμε με αφετηρία το κράτος του Βέμπερ, το οποίο καθορίζεται από μια επικράτεια, το λαό και τη γραφειοκρατία, η οποία ε, έχει ε, δημιουργήσει ένα, έναν ισχυρισμό για το μονοπόλιο εναντί της ε, νόμιμης ε, χρήσης βίας, η χάρτα, ε, δείχνει σημαντικές τροποποίησεις στην Ευρώπη. Πρώτον, είναι αποτέλεσμα διακρατικών διαπραγματεύσεων, συζητήσεων και έγκρισης. Έχει επικυρωθεί από τα κράτη-μέλη, αλλά δεν είναι το προϊόν εθνικού συνταγματικού συστήματος κάποιου κράτους μέλους ή οποιοδήποτε κράτους μέλους. Η εξουσία να δημιουργηθεί αυτό το σύνολο δικαιωμάτων περιγράφει μια αρχή η οποία δεν είναι μια του κράτους τύπου Βέμπερ. Παρ' όλα αυτά η χάρτα έτσι όπως τροποποιήθηκε τροποποιεί ε, την, αξίωση των κρατικών αρχών να έχουν το μονοπόλιο για τη την νόμιμη χρήση βίας. Και πάλι θα σας παραπέμψω στα σχόλια που έκανα πιο πριν για την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Ηνωμένου Βασιλείου και το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και τον αντίκτυπο που θα έχει για τις, αρχές, το, τις κρατικές αρχές σχετικά με την νομιμότητα και την νομιμοποίηση για τη χρήση βίας. Αυτοί προς τους οποίους ισχύουν τα δικαιώματα της χάρτας δεν μπορούν να είναι περιορισμένες με τις, από την πράξη μιας εθνικής αρχής Δηλαδή, οι αρχέ ενό κράτου μέλου δεν μπορούν να αποφασίσουν ότι το δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή θα ισχύει μόνο για του δικού του υπηκόου. Απαιτείται από τη χάρτα να δεχτούν ότι αυτά τα δικαιώματα ισχύουν για του υπηκόου οποιοδήποτε άλλου κράτου μέλου που τυχαίνει να βρίσκονται στην δικαιοδοσία του. Και επίση απαιτείται μέσω τη χάρτα να διασφαλίσετε ο σεβασμό αυτών των δικαιωμάτων και για του ε, υπηκόου τρίτων χωρών οι οποίοι πληρούν τον κανόνα περί δικαιοδοσία. Και αυτό είτε βρίσκονται σε τακτά χρονικά διαστήματα είτε όχι στην επικράτεια. Έτσι, αυτοί οι οποίοι έχουν δικαίωμα στα δικαιώματα της χάρτας δεν είναι τα άτομα του κράτους του Βέμπερ και ούτε μπορούν να περιοριστούν σε αυτή την ομάδα. Τέλος, η επικράτεια στην οποία ενισχύουν τα δικαιώματα της χάρτας δεν μπορεί να τροποποιηθεί από οποιοδήποτε κράτος μέλος. Η ικανότητα ενός κράτους να καθορίσει τα ότι τα δικαιώματα της χάρτας δεν θα ισχύσουν σε μέρος της επικράτειας. Για παραδείγμα, το χάρη οι Αυστραλιανές αρχές όταν ε, εξαίρεσαν το Christmas Island, το οποίο είναι μέρος της Αυστραλίας, αλλά όχι για την ε, υποβολή αίτησης ασύλου. Οι αρχές όμως των κράτους μέλους είναι υποχρεωμένες να διασφολήσουν την ε, πλήρη τήρηση των δικαιωμάτων της χάρτας για όλα τα άτομα που έχουν δικαίωμα σε αυτά. Σε αυτή την παρουσίαση προσπάθησα να παρουσιάσω τι βασικέ αλλαγέ τι οποίε επιφέρει για του πολίτε η συνθήκη τη Λισαβόνα. Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών είναι η πρόσβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της νομικής δράσης ε, ε, που δίνει η συνθήκη τη Λισαβόνα στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Και υπάρχουν τρει βασικέ συνέπειε. Πρώτον, οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τώρα μια χάρτα δικαιωμάτων που είναι νομικά δεσμευτική και θα πρέπει να τηρούν οι κρατικές αρχές σύμφωνα με το καθήκον της καλής πίστης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερη συνέπεια, οι υπήκοοι τρίτων χωρών μοιάζουν όσο, όλο και περισσότερο με τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι συμπεριλαμβάνονται ως δικαιούχοι των δικαιωμάτων της Χάρτας με τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και οι πολίτες της Ένωσης. Τρίτον, η Χάρτα προβλέπει ένα νέο και ε, πιθανώς ε, σημαντικό πακέτο ε, δικαιωμάτων για διάφορα άτομα στην Ευρώπη που δεν μπορεί να τροποποιηθεί από οποιοδήποτε κράτος μέλος και τις σχετικές αρχές με βάση την όχληση που μπορεί τα δικαιώματα αυτά να δημιουργήσουν στο κράτος αυτό. Υπήρξε δηλαδή μια διάσπαση κατά κάποιο τρόπο, ένας διαχωρισμός αρχών και δικαιωμάτων, τα οποία θα βοηθήσουν τις αρχές των κρατών μελών, των κρατών μελών να έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μεταξύ τους και στους πολίτες βεβαίως να έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις κοινωτικές αρχές. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σχολαστική νομική ανάλυση της δυναμικής των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του όλου πλαισίου εφαρμογής τους. Θα ακούσουμε τώρα τον Ειδικό Σύμβουλο και επίτιμο καθηγητή ε, στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εντάχει από εντελώ διαφορετική οπτική γωνία να σας κάνω την παρουσίασή μου. Θα παρουσιάσω τις πολιτικές μάλλον πτυχές της ηθαγένειας. Πολύ απλή η δομή της παρουσίασής μου. Πρώτα θα δούμε τον ευρωπαϊκό πολιτικό χώρο, λέει ο καθηγητής Σιντάνσκι, που τώρα δημιουργείται. Μετά θα δούμε τη δημοκρατία από δύο οπτικές γωνίες. Την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, που γνωρίζετε πολύ καλή, καλά, αλλά και την άμεση δημοκρατία, που τώρα εισάγεται στο ευρωπαϊκό σύστημα. Το δεύτερο κεφάλαιο εντάχει θα το αφιερώσω στα διάφορα είδη διαβούλευσης. Γιατί υπάρχουν μηχανισμοί διαβούλευσης υπάρχουν όργανα διαβούλευση του μηχανισμού που έχει καθιδρύσει η Κομισιόν, είναι τρόποι πρόσβασης ε, των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Και θα συνάγω και κάποια συμπεράσματα. Και κάποιες απαντήσεις στο εξής ερώτημα. Άμεσα τι θα πρέπει να κάνουμε, ούτως ώστε οι νέοι μας να αρχίσουν να ενδιαφέρονται για την Ευρώπη γιατί πολύ σύντομα θα, θα πάρουν τη σκητάλη. Σύντομα εμείς θα αποχωρήσουμε μεταξύ αυτών και φαινόμενος. Θα αναφέρω τρεις άξονες πολύ απλά. Το θέμα του μαθήματος πολιτικής αγωγής, μετά, δεύτερος άξονας. Εν γέννη θα πρέπει να προσέξουμε τη διάσταση της παιδείας, στη σχολεία μας. Τρίτος άξονας, επιστημονική μέθοδος εισαγωγή επιστημονική μεθόδου. Και τέλος θα κάνω και κάποιες καθαρά προσωπικές παρατηρήσεις. Σε σχέση με αυτό που ανέφερε στην παρέμβασή του ο πρόεδρος Μπαρόσο. Βεβαίως ε, πάντα υπό την προσωπική μου ιδιότητα μιλώ όπως θα διαπιστώσετε. Να δούμε τον ευρωπαϊκό πολιτικό χώρο πρώτα απ' όλα σε εισαγωγικά μου σχόλια. Στη συνθήκη αυτή πρώτη φορά, πρώτη φορά ο άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο επί τις βάσεις του οποίου αναπτύσσονται οι ελευθερίες και τα δικαιώματα που ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Ντεβίγκο. Πάνω απ' όλα η ελεύθερη, η ελεύθερη έκφραση, η ελεύθερη σκέψη, η ελευθερία της έκφρασης, η, της ενημέρωσης ε, και η ελευθερία του, και η ελεύθερη σύσκεψη, η συγκέντρωση. Όλα αυτά αποτελούν τα θεμέλια της δημοκρατίας μας. Όλα αυτά τα στοιχεία θα τα δούμε σε λίγο. Άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή στην ε, συνθήκη από πλευράς πολιτικών επιστημών είναι η αναγνώριση του ρόλου των πολιτικών ομάδων. Στο εγγύς μέλλον αυτές οι πολιτικές ομάδες, αυτά τα κόμματα αποτελούν την έκφραση της βούλησης των ε, πολιτών. Αντιπροσωπευτική λοιπόν δημοκρατία. Ε, δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το τι πράττει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το τι εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γνωρίζουμε ταυτόχρονα όμως ότι δυναμώνονται οι εξουσίες του με τη συναπόφαση με τους διάφορους τομείς ε, που προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας. Ενδυνάμωση λοιπόν του Ευρωκοινοβουλίου. Άρα προβληματίζομαι. Ενισχύονται οι εξουσίε του Ευρωκοινοβουλίου. Και τα επίπεδα συμμετοχή δεν ενισχύονται. Τι διαπιστώνουμε. Μειώνεται η συμμετοχή των πολιτών ενώ αυξάνονται οι εξουσίε του Ευρωκοινοβουλίου. Μήπω υπάρχει έλλειμμα ενημέρωση του πολίτη. Γιατί θα πρέπει να γνωρίζει ο πολίτη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι πλέον συμβουλευτικό όργανο. Έχει ουσιαστικές εξουσίες. Πρώτο ενδιαφέρον σημείο. Δεύτερη παρατήρηση. Κάνοντας τη σύγκριση με τη συμμετοχή στα κρατημέλη, βλέπουμε γενικά ότι είναι πιο αυξημένη η συμμετοχή. Αλλά τι διαπιστώνουμε, ότι υπάρχουν δύο ομόσπονδα κράτη όπου η συμμετοχή είναι γύρω στο 50%. Ή, είπα και Ελβετία. Στην Ελβετία έχουμε 45% συμμετοχή συχνά στις εκλογές για την Ελβετική Βουλή, τότε εκφράζουν μεγάλη ικανοποίηση και λένε μεγάλη επιτυχία. Άρα και εκεί πέρα η προσέλευση στις κάλπες ε, είναι πολύ περιορισμένη. Σε δομέ όπου η εξουσία είναι κάπως αφηρημένη, όταν η σχέση δεν είναι άμεση μεταξύ της ψήφου διότι ε, ε, βουλή εκλέγουν οι Ελβετοί, αλλά δεν γνωρίζουν ε, μετά ποιοι είναι οι Ελβετοί έρχονται και εδώ πέρα. Προσερχόμαστε σε ευρωεκλογέ. Α πούμε, έχω ελληνική υπηκότητα, άρα ψηφίζω στι ευρωεκλογέ. Αλλά δεν ξέρουμε μετά ποια θα είναι τα μέλη τη Κομισιόν, ποιο θα είναι ο πρόεδρο τη Κομισιόν. Εξού και η πρόταση του Jacques Delors θα πρέπει να υπάρχει κάποιος συσχετισμός μεταξύ του αποτελέσματος και της επιλογής του Προέδρου. Ποια συνέπεια θα έχει αυτό. Ο Πρόεδρος να μπορεί να απαρτίζει τη δική του Κομισιόν και όχι αυτό να του επιβάλλεται. Και να χρειάζεται ε, να διαπραγματευτεί, να το διαπραγματευτεί. Αυτή είναι η πρώτη πτυχή. Δεύτερον, τι άλλο διαπιστώνουμε. Παρά τις προβλέψεις του ΧΑΣ, θυμάστε στο βασικό του έργο για την Ευρώπη, περί ευρωπαϊκής ε, ολοκλήρωσης, τι έλεγε, ότι ταυτόχρονα θα έχουμε σύσταση πραγματικών ευρωπαϊκών κομμάτων, ενώ όλα αυτά σε εμβριακή μορφή βρίσκονται πάντα και τι άλλο έλεγε. Μαζί με τις οικονομικές, κοινωνικές αρμοδιότητες θα ανθοφορήσουν διάφορες ομάδες ενώσεις πολιτών που θα συσταθούν για συνεχή διάλογο με τη νέα αυτή εξουσία. Τι διαπιστώνουμε ότι αυτό δεν ισχύει. Τρίτη παρατήρηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις ενισχυμένες του πλέον εξουσίες βρίσκεται στο στόχαστρο των ομάδων πίεσης. Παλιά, θυμάμαι, ε, κυκλοφόρουσα στους διαδρόμους του Ευρωκοινοβουλίου και οι ευρωβουλευτές μου έλεγαν «Κανείς δεν νοιάζεται για μας». Και τώρα δεν ξέρουν πώς να γλιτώσουν από όλους αυτούς που τους κατατρέχουν. Ιδού ο δείκτης Τη ε, της σημασίας ενός θεσμικού οργάνου. Αυτέ οι ομάδες πίεσης ξέρουν πολύ καλά σε ποιον απευθυνθούν. Προσπαθούν να επηρεάσουν τη διαδικασία λήψη αποφάσεων οι ομάδε πιέση προφανώ και να ε, επηρεάσουν και στο αποτέλεσμα αυτή τη διαδικασία. και αναλαμβάνουν αποτελεσματική δράση στο βαθμό του δυνατού βέβαια. Αυτός είναι ο στόχος τους τουλάχιστον. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εξέλιξη λοιπόν. Ιδού ένα θετικό στοιχείο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα. Άμεση συμμετοχή. Έχουμε εισαγωγή της πρωτοβουλίας στην, ε, στο ευρωπαϊκό πολιτικό γίγνεσθε. Μιλάμε για μεγάλο επιτεύγμα πολύ ενδιαφέρον σίγουρα. Ένα εκατομμύριο πολίτες δίνεται να αναλάβουν και να καταθέσουν πρωτοβουλία. Υπάρχουν, υπάρχει ειδικό κανονισμό πρώτην η Κομισιόν και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που εξηγεί αυτή τη διαδικασία προτού να αναλάβουν αυτοί οι πολίτες ε, μια πρωτοβουλία. Χρειάζεται και ένα τρίτο των κρατών μελών. Υπάρχουν κάποιοι όροι από πλευράς αριθμού κρατών. Τρίτον, επίπεδα συμμετοχή στα κράτη-μέλη μεταξύ των ε, συμβαλωμένων μερών. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Και διαφορετικό, α πούμε, από την ελβετική περίπτωση, όπου αναλαμβάνεται η πρωτοβουλία ανεξαρτήτως καντονίων ε, κτλ. σε ελβετικό οσποδιακό επίπεδο. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί να γίνει αποδεκτή βέβαια αυτή η πρωτοβουλία Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε προηγουμένως. Αν η πρωτοβουλία βασίζεται σε αξίες που μάλλον σε κάτι που αντίκειται σε βασικές αξίες της Ευρώπης αν τότε δεν μπορεί να γίνει αποδεχτή προφανώς αυτή η πρωτοβουλία. Η πρωτοβουλία επίσης θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά και μόνο το μη αρμοδιότητας της Κομισιόν. Γιατί διότι αυτή η πρωτοβουλία αντίθετα με την ανάληψη πρωτοβουλία στην Ελβετία. Διότι στην Ελβετία τι γίνεται. Από τη στιγμή που περνάει αυτομάτω εγγράφεται στη συνθήκη, στο σύνταγμα, συγγνώμη. Ενώ εδώ πέρα η πρωτοβουλία απλά εξαναγκάζει την Κομισιόν να κάνει κάτι. Την εξα... Εξαναγκάζει την ε, Κομισιόν σε ανάληψη δράσης με συγκεκριμένη πρόταση που την απευθύνει προ το Συμβούλιο Υπάρχει μια διαφορά, ε. Παραμένουμε πάντα στη γνωστή διαδικασία λήψη αποφάσεων. Η Κομισιόν προτείνει, το Συμβούλιο αποφασίζει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, σε πλαίσιο συναπόφασης τουλάχιστον. Στο πλαίσιο πάντα της, ε, και στο πλαίσιο πάντα της νομοθετικής διαδικασίας. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Στην Ελβετία είναι πολύ πιο άμεσα τα πράγματα διότι πώς θα το κάνουμε, παρά τις διαφορές τους, ελβετικός λαός υπάρχει. Ενώ εδώ πέρα γίνονται υπολογισμοί ανά κράτος και με σαφή κριτήρια. Τον έχω διαβάσει το σχετικό κανονισμό. Είναι πολύ περίπλοκος, οπότε δεν θα αναφερθώ καθόλου σε αυτό το κανονισμό. Μιλάμε για βαρύτατη διαδικασία. Ακόμα και σε ένα μικρό κράτος για την Ελβετία είναι βαρύτατη διαδικασία, πόσο δε μάλλον σε επίπεδο ευρωπαϊκό με τις αναλογίες που προβλέπονται ανά κράτος. Πολύ ενδιαφέροντα βεβαίως πάντα όλα αυτά. Άλλη άμεση επαφή μεταξύ του πολίτη και της εξουσίας. Τα πετήσω Πολύ ενδιαφέροντα και αυτά από δύο οπτικές γωνίες. Και εδώ και χρόνια υφίστανται. Χιλιάδες ε, κατατίθεται κάθε χρόνο για μας, τους ε, πολιτολόγους και τους κοινωνιολόγους. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το φαινόμενο. Εξετάζουμε την όλη διαδικασία. Είναι και αυτός ένας τρόπος συμμετοχής της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ότι πάντα, έχουν, ε, πάντα επηρεάζουν την εξουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από πλευράς κοινωνιολογικής ε, είναι ενδιαφέρον για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Πολιτικού Χώρου. Πολλοί συντάκτες ε, και πολλοί συγγραφείς αναφέρονται σε αυτόν τον όρο, όπως γνωρίζετε. Βεβαίως έχουμε το ρόλο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, άμεση πρόσβαση και πάλι για τον πολίτη, ακροάσεις. Βλέπουμε την εξέλιξη σε όλες αυτές τις διαδικασίες Και το ίδιο ισχύει και το θέμα της ενημέρωσης. Άλλο είδος συμμετοχής του πολίτη. Είναι η συμμετοχή στα εθνικά δημοψηφίσματα. Το είδαμε. Στην περίπτωση της Λισαβόνας. Μιλάμε για φοβερή συζήτηση στη Γαλλία. δεν λέω ότι ήταν πάντα σωστή η επιχειρηματολογία, υπήρχε και στρέβλωση. Δεν υπήρχε πάντα σωστή η κατανόηση και αντίληψη της Ευρώπης. Αυτοί που καταψήφισαν καμιά φορά πήγαιναν και έλεγαν εμεί και αν πιστεύουμε στην Ευρώπη. Πώς γίνεται αυτό. Αλλά ήταν και αυτό ένα είδο συμμετοχή έστω. Έγινε πολύ εντόνη συζήτηση στη Γαλλία. Θυμάμαι επίση ε, τη συζήτηση που έλαβε χώρα το 54 Περισέντε. Απίστευτη ιδεολογική συζήτηση. Το αποτέλεσμα δεν σημαίνει απαραίτητος ε, καλύτερη γνώση της επικαιρότητα ή της λειτουργίας της Ευρώπης. Δεν το πιστεύω. Υπάρχει κάτι πάντως που όλους μας ε, πρέπει να μας προβληματίσει. πώς γίνεται να δεχόμαστε ένα δημοψήφισμα που είναι πολύ δημοκρατικό σε εθνικό επίπεδο, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι αντιδημοκρατικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί έχετε μία μειονότητα με συμμετοχή της τάξης που το 60% που όπως έγινε καταφέρουν να μπλοκάρουν το Σύνταγμα, τη Συνταγματική Συνθήκη. Αυτό, μας, ε, αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Εξού και προέκυψαν σχέδια για ενδεχόμενο ευρωπαϊκό δημοψήφισμα. Αν φανταστούμε ότι θα προκύψει νέα συνταγματική συνθήκη, θα είναι τέρμονη οι συζητήσεις, το είπε ο Ζησκάρδεστα. Αλλά, αλλά μην του ακούτε του πολιτικού, διότι εν μέρει ήταν και ο συντάχτης κιόλα. Συγγνώμη για αυτά που λέω, συγγνώμη για την ειλικρινία μου. Το ενδιαφέρον στοιχείο ποιο είναι. Εδώ και χρόνια είχαμε συνθήκες που τροποποιούσαν μια συγκεκριμένη δομή. Και έτσι είχαμε αυτές τις εξελίξεις κατά τα τελευταία 60 χρόνια. Είχαμε πολύ περιορισμένες συνθήκες, ενώ τώρα καλύπτουμε κάθε αρμοδιότητα έως και φεύγουμε νέες αρμοδιότητες σε διάφορους σημαντικούς και καινούριου ακόμα τομείς. έχουν ε, ξεκινήσει ήδη κάποιες εργασίες για το ευρωπαϊκό δημοψήφισμα. Να σας θυμίσω κάτι. Ο στρατηγός Ντεγκόλ ήταν ο πρώτος που πρότεινε, ε, ήταν αυτός που πρώτο πρότεινε το ευρωπαϊκό δημοψήφισμα. Οπότε λίγο σεβασμό στο στρατηγό τουλάχιστον, γιατί όχι να την εξετάσουμε και αυτή τη δυνατότητα. Όταν πρόκειται για εκβάθρον ε, αλλαγές. Ενδεχομένω για νέα συνταγματική συνθήκη μελλοντικά. Ξέρω ότι αυτό θα πάρει πολύ χρόνο. Ένα τέτοιο δημοψήφισμα δυνατόν να εμπνέεται από τα ελβετικά δεδομένα, όπου απαιτείται διτή πλειοψηφία. Πλειοψηφία του πληθυσμού στο σύνολό του και των καντονίων πλειοψηφία. Αν δούμε τη νέα διαδικασία λήψη αποφάσεων της Λισαβόνας, και κάνουμε τον παραλληλισμό, σε επίπεδο συμβουλίου, πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ας πούμε το 2014. Λαμβάνεται υπόψη μια κάποια πλειοψηφία 60% των κρατών και του πληθυσμού και του λαού. Άρα πρόκειται για ομοσπονδιακή διαδικασία. Αντιπροσώπευση ταυτόχρονα των οντοτήτων που είναι μέλη της Ένωσης και ταυτόχρονα του ίδιου του λαού. Παραμένει ανοιχτή αυτή η πόρτα μελλοντικά. Διαβουλεύσεις τώρα. Δεν θα μακρηγορήσω. Διότι ξέρουμε τι έγινε στην Ευρώπη. Πώς διαμορφώθηκε η ευρωπαϊκή εξουσία. Προέκυψαν ομάδες πολιτών, ενώσεις πολιτών, ομάδες πίεσης, επαγγελματικέ οργανώσεις κτλ. Μιλάμε για εκατοντάδες τέτοιες ενώσεις. 1.500-3.000 ομάδες πίεσης λένε κάποιε πηγές. 500 1.000 οι διαφορετικέ επαγγελματικέ ενώσει, όλο και πιο ειδικευμένε τι διαπιστώνουμε και όλα αυτά εδώ και χρόνια τα μελετάμε. Υπάρχει παραλληλισμός μετα... μεταξύ των δύο διαδικασιών. Η συνθήκη τι προβλέπει. Στον τομέα της υγείας προβλέπει αναγνώριση νέων επαγγελματιών, χειροπρακτόρων. Τότε οι χειροπράκτορες αυτομάτως προχωρούσε σύσταση ένωσης και προχωρούσε συνεχή διάλογο με την εξουσία. Ιδού ο παραλληλισμός με τη δημιουργία ενός στρώματος νέων δομών με τη συμμετοχή καμιά φορά άμεση, καμιά φορά έμεση των πολιτών. Είναι γνωστές λοιπόν όλες αυτές οι ενώσεις, οι πολυάριθμες. Μπορεί να είναι και κάτι πιο θεσμοθετημένο. Ας πούμε, σαν η παλιά Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή. Περάστε μπροστά από το χτίριό τους για να αντιληφθείτε τις εξελίξεις. Με ένα ελάττωμα όμως. Δεν είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικό αυτό το όργανο. Είναι ελάχιστα τα μέλη για να εκπροσωπήσουν ισορροπημένα τα διάφορα συμφέροντα. Ποιο είναι το αντιστάθμισμα όμως. Ενώσεις όπως η ΚΟΠΑ, Business Europe, τα συνδικάτα συντονίζουν τα μέλη της ΕΟΚΕ. Άρα, όλες αυτές οι κοινωνικές διαδικασίες, κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Διότι θέτουν τα θεμέλια για την πρόσβαση του πολίτη. Άλλο ενδιαφέρον στοιχείο, η Επιτροπή των Περιφερειών. Ακόμα πιο σημαντικό στοιχείο. Σημαίνει ότι έχουμε αρετού άρχοντες στην Επιτροπή των Περιφερειών. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Επιτροπή των Περιφερειών. Και πάλι το θέμα τη αντιπροσωπευτικότητα. Διότι υπάρχουν μεγάλε ανισορροπίε μεταξύ των περιφερειών μα. Πάρτε τα ομόσπονδα κρατήδια, πάρτε τι περιφέρειε στο Βέλγιο. Αν επιβιώσει δηλαδή το Βέλγιο. Δείτε τι ισπανικέ περιφέρειες αυτόνομε κοινότητε και κάντε συγκρίσει με άλλε χώρε όπω η Γαλλία όπου τώρα αρχίζουμε μόλις, μόλις να μιλάμε για περιφέρειες, με τεράστιες ανισορροπίες. Σε κάποιες χώρες δεν υπάρχει καν τέτοια παράδοση. Στην Ελλάδα, ούτε στην Πορτογαλία δεν υπήρχε τέτοια δομή. Χρειάστηκε βαθμιαία να συσταθούν και σε πολιτικό και σε οικονομικό επίπεδο. Πολλοί δείχτες τι δείχνουν, σύγκληση συμφερόντων δείχνουν. για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωση και για θέματα ευρωπαϊκών διαδικασιών. Δείτε τι γίνεται στα μέσα μαζική ενημέρωσης. Δείτε τι γίνεται στι μεγάλε επιχειρήσει, Δείτε τα think tanks που έχουν συσταθεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν όλες αυτές οι ιδέες που κυκλοφορούν και αυτό το φαινόμενο που διαπιστώνουμε. Και καταλήγω, γιατί όλο αυτό είναι το υπόβαθρο. Για τους νέους τι κάνουμε. Διότι αυτό είναι το βασικό για το μέλλον. Είναι απαραίτητη η ευρωπαϊκή πολιτική αγωγή. Κοιτάμε δεξιά-αριστερά. Πουθενά δεν παρέχεται αυτή η ευρωπαϊκή πολιτική αγωγή. Υπήρχαν κάποια ιδρύματα που ήθελαν να καταστήσουν κάποια χειρίδια. Ξαφανίστηκαν. Η Κομισιόν, η Γενική Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού θα πρέπει να το πάρει σοβαρά υπόψη. Ακούσαμε ενδιαφέρουσες ομιλίες, αλλά θα ήθελα να ακούσω και συγκεκριμένους στόχους. Να τους κουβεντιάσουμε από κοινού και να δούμε γιατί δεν έχουν επιτευχθεί. Στο πλαίσιο αυτού του παιδαγωγικού έργου θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο στοιχείο για να προσελκύσουμε τους νέους. Ας πούμε, να τους μιλήσουμε για το περιβάλλον και να τους εξηγήσουμε. Δεν μπορούμε να το λύσουμε σε γαλλικό, σε ισπανικό επίπεδο και μόνο. Οφείλουμε να το δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να μην, για να πω σε παγκόσμιο δηλαδή. Ιδού πώς ε, γύρουμε, ξυπνάμε το ενδιαφέρον των νέων μας. Γιατί τους ενδιαφέρει ας πούμε πάρα πολύ το περιβάλλον. Και μπορούμε να παίξουμε και παιχνίδια κιόλα ε, προσωμείωσης στα σχολεία, στα διάφορα φόρα παίξουμε το παιχνίδι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι να μάθουμε πώς λειτουργεί στην πράξη. Ευρωπαϊκή παιδεία. Πάρα πολύ σημαντική η διάστασή της. Ας πούμε, στο μάθημα της ιστορίας έχουμε το νέο γαλλογερμανικό εχειρίδιο που είναι αξιοσημείωτο. Με ερωτήματα και που δίνει δύο οπτικές γωνίες του ίδιου φαινομένου. Πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, η διάμεση περίοδος. Γιατί να μην κάνουμε το ίδιο για την ευρωπαϊκή ιστορία. Η Κομισιόν θα πρέπει να αναλάβει τέτοιες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διότι ο καθένας έχει να πει τη δική του ιστορία και έχει τη δική του ερμηνεία των πραγμάτων. Μελλοντικά μπορεί ε, να οδηγήσει σε κρίξεις και σε εντάσεις και σε αντιευρωπαϊκές ακόμα τάσεις. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το στοιχείο. Θα πρέπει να εισάγουμε όλες αυτές τις αξίες, ευρωπαϊκές αξίες και τις δημοκρατικές μας αρχές. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ένα θεωρητικό επίπεδο, έτσι αιωρούνται κάπου, χωρίς να διεισδύουν στο μυαλό των νέων. Ως προς την παιδεία, υπάρχουν και άλλα σημαντικά στοιχεία. Πέραν της ιστορίας, τα σύνορα. Πώς έχουν χαραχθεί τα σύνορα. Σήμερα έχουμε τη νέα Ουγγρική κυβέρνηση που υποσχέθηκε Ουγγρικά διαβατήρια ε, σε Ούγγρους που ζουν σε όμορα κράτη. Αυτό αντίκειται στις ευρωπαϊκές αξίες ή το αντίθετο. Θα πρέπει να αποδώσουμε μεγάλη σημασία στα σύνορα. Να μιλάμε για μεγάλη Κροατία, για μεγάλη Σερβία. Μήπως θα τροφοδοτούμε αυτά τα κινήματα. Ή αντίθετα, θα πρέπει να επιμείνουμε στις δικές μας αξίες. Ε, μελετώντας, ε, εξετάζοντας τα φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα σε τρίτες χώρες. Τρίτο στοιχείο. Εισαγωγή στην ιστορία του της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και του ευρωπαϊκού οικοδομήματος η ιστορία αυτή αρχίζει βεβαίω μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων. Είναι ιδέες που μετά μετατρέπονται σε πολιτικά κινήματα. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο, μόλις αποκαταστάθηκε η ειρήνη, προέκυψαν υπερεθνικά κινήματα. Τα δημοκρατικά κόμματα, τα χριστιανοδημοκρατικά, τα σοσιαλιστικά, ανέλαβαν δράσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο από κοινού για να προωθήσουν τι ευρωπαϊκέ ιδέε. Το ίδιο και σε επίπεδο οικονομικό, το ίδιο και σε επίπεδο εκπαιδευτικό. Θα πρέπει όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη μελλοντικά στις εργασίες μας. Θυμάμαι ότι διάβασα ένα έγγραφο της Κομισιόν πριν από χρόνια που μιλούσε για τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ελοκλήρωσης και ξεκινούσε από το Jean και με την ΕΚΑΧ. Ε, όχι. Η Ευρώπη δεν δημιουργήθηκε από πάνω προς τα κάτω. Δεν ξεχνάμε και τις ρίζες μας. Διότι επί της βάσης αυτής χτίστηκε μετά το ευρωπαϊκό οικοδόμημα το Ζαμονέ που είχε αυτό το όραμα. Φανταστικό όραμα. Τρίτη διάσταση. Επιστήμες. Αυτό και είναι το αντικείμενό μου. Κρίμα που δεν έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο Μπαρόσο. Θα μου έλεγε πάντα τα ίδια λες. Δεν χάνεις ευκαιρία. Ναι, δείτε το 30% των δημοτικών στη Γαλλία εφαρμόσουν αυτή τη μέθοδο. Είναι συμπληρωματική και με πειράματα προσεγγίζει τα επιστημονικά προβλήματα με υποθετικά σενάρια, με αποδεκτικά στοιχεία και με συζήτηση. Πέραν αυτής της τεχνικής πτυχής, να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα, διότι αν θέλουμε να αναβαθμίσουμε το επίπεδο των μελλοντικών γενεών και να επιτρέψουμε όντως τη συμμετοχή τους, να μιλάμε όντως για δραστήριους και ενεργού πολίτες, όχι για που παραγνωρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, δείτε τα χαμηλά ποσοστά ε, ε, ε, δείτε πόσος κόσμος δεν ξέρει τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να τους δώσουμε και τα μέσα της γνώση σε κάθε επίπεδο. Αυτή η μέθος μας επιτρέπει να μάθουμε τι εστί διάλογος, αποδείξεις, επιχειρηματολογία σε τεκμηριωμένη βάση και τελικά Μιλάμε για σεβασμό του καλύτερου. Άλλο αποτέλεσμα. Έτσι μαθαίνει κανεί τι εστί δημοκρατία. Και μιλώ για τα δημοτικά και τα γυμνάσια. Από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Και πριν το δημοτικό ακόμα. Θα πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά μας ε, τι έχει επιτευχθεί. για να δουλέψουν με τη σειρά του υπέρ τη Ευρώπης. Είναι απαραίτητη προπόθεση για να διασφαλίσουμε το μέλλον τη Ευρώπη. Καταλήγω σε κάποιες προσωπικές παρατηρήσεις εντάχει. Με κοιτάει και η Πρόεδρος, με αυστηρό ύφος, αν και πολύ ευγενικό. Μου επέτρεψε να ξεπεράσω το χρόνο αγόρευσης. Θα καταλήξω σε κάποιες προσωπικές, προσωπικές παρατηρήσεις. Δείτε τι λέει το Ευρωβαρόμετρο. Η εικόνα της Ευρώπης ποια είναι. Η ελεύθερη κυκλοφορία πάνω απ' όλα η δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης σε αυτό το χώρο ελευθερίας. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα. Σχεδόν 50% των πολιτών λένε η Ευρώπη είναι αυτή η ελεύθερη κυκλοφορία που απολαμβάνω σε αυτόν τον ε, νέο χώρο. Δεύτερη εικόνα της Ευρώπης. Το ευρώ. Το 37% των πολιτών λέει το ευρώ, το σύμβολο της Ευρώπης. Το γιατί το ξέρουμε. Δεν θα το αναλύσω γι' αυτό. Τι διαπιστώνουμε. Αυτή η ύφεση, η επίθεση, πείτε την όπως θέλετε, κατά του ευρώ, δυνατόν να οδηγήσει και σε κρίση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Πήρε χρόνο στην κυρία Μέρκελ να το αντιληφθεί. Στην αρχή ήθελε να εκδιώξει την Ελλάδα. Μετά είπε να τη βοηθήσουμε την Ελλάδα σε πλαίσιο αλληλεγγύης και στην τελευταία της ομιλία πάει και παραπέρα. Λέει πως εάν αποτύχει το ευρώ τότε θα αποτύχει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Άρα αυτός ο πυρήνας της ευρωζώνης θα παραλύσει και η επιστροφή στα εθνικά νομίσματα θα επέφερε απίστευτο χάος. Φοβερές απώλειες. Και θα αμαυρωνόταν η εικόνα της Ένωσης στο παγκόσμιο προσκήνιο. Η εμπιστοσύνη. Άλλο, άλλο απαραίτητο στοιχείο στην Ευρώπη. Η εμπιστοσύνη του πολίτη είναι γύρω στο 50%. Και σήμερα θα έλεγα ότι θα είναι, είναι ακόμα χαμηλότερη. Καλό θα ήταν να γίνουν τώρα δημοσκοπήσεις. Από τη στιγμή που έγινε αυτός ο διάλογος μεταξύ Ελλάδας, Γερμανίας και λοιπόν κρατών μελών και θέματα αλληλεγγύης, μπορούμε να τη βοηθήσουμε την Ελλάδα, δεν μπορούμε να τη βοηθήσουμε. Λόγω της συζήτησης αυτής μειώθηκε η εμπιστοσύνη του πολίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. παρά τις προσπάθειες της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και άλλων να περιορίσουν τις απάνες τους, παρά τις προσπάθειες τους λοιπόν, δυνατόν επέλθει περισσότερη ανεργία, χαμηλότερες συντάξεις, μείωση των μισθών, χίλιας δυο συνέπειες. Αυτή είναι επίθεση εις βάρος του πολίτη, εις βάρος της ζωής του, του επίπεδου ζωής του. Και ταυτόχρονα τι του λέμε, θα επιβάλλουμε κυρώσεις αν το κράτος σου κάνει διαφορετικό. Άρα, η Ευρώπη είναι ο αστυνομικό. Καθόλου δεν μου αρέσει αυτή η εικόνα της Ευρώπης, το αστυνομικό. Με άλλες αποχρώσεις βεβαίως το έθεσε και ο πρόεδρος Μπαρόσο. Μίλησε για συμμόρφωση με στόχο να δοθούν κίνητρα. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να αντιστρέψουμε την τάση. Θα πρέπει να δούμε τι μας λέει η κοινή μας γνώμη. Θα πρέπει να προσέξουμε τις ε, συζητήσεις σε επίπεδο μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οπωσδήποτε η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει αυτή την εικόνα της αλληλεγγύης, του δυναμισμού. Δηλαδή καλός ο έλεγχος των αγορών, αυτό είναι απαραίτητο, αλλά θα πρέπει να το βλέπουμε πιο σφαιρικά. Δεν θα πρέπει να μιλάμε μόνο για τομεακά επιτεύγματα ή μονομερή επιτεύγματα, όπως συνέβη με την κερδοσκοπία. Το είδαμε ας πούμε τα γερμανικά κρατικά ομόλογα. Δεν είναι σωστό να είναι όλο και πιο αρνητική η εικόνα της Ευρώπης, όπως αυτή που τώρα δίνουμε. Δεν θα καταφέρουμε να βγούμε από την κρίση παρά μόνο να μας στηρίξει η κοινή γνώμη, παρά μόνο να μας στηρίξει ο πολίτης. Δεν, θα, δεν είναι δυνατόν να μιλάμε μόνο για κύρωση και για ποινή στον πολίτη. Ιδού, ε, θα στερηθεί δικαιώματος ψήφου το κράτος μέλος σου. Για χι χρονικό διάστημα. Στην αρχή θα είναι εφοπλισμένος, θα τηρήσει στάσεις υγιής, αλλά μια μέρα θα εμπλακεί σε κοινωνικές αναταραχές που το έχουμε ήδη δει στην Ελλάδα και δυνατόν να προκύψει και σε άλλα κράτη-μέλη. Απευθύνω εκκλησή ούτω ώστε να ληφθούν αυτά μέτρα. Ολοκληρώνω με την ελπίδα να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του πολίτη στην Ευρώπη. Είναι απαραίτητη η συμμετοχή του πολίτη για να εξέλθουμε της ύφεση. Αυτή την αποστολή θα πρέπει να αναλάβει η Κομισιόν και τα θεσμικά όργανα. Η Task Force τελικά είναι σύνοδος των Υπουργών Οικονομικών. Χρησιμοποιούν αυτή την ορολογία, δεν είναι ορθό. Και την Προεδρία την έχει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Για μένα τι σημαίνει αυτό. Ίσως να διαφωνείτε βεβαίως. Διαμάχη εξουσίας. Διακριτική με διαμάχη. Αλλά αυτό βλέπω μεταξύ της διακυβερνητικής διάστασης, μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών και του κοινοτικού επίπεδου, όπου η Κομισιόν και το Ευρωκοινοβούλιο παίζουν θεμελιώδη ρόλο, το γνωρίζουμε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Και όπως είπε και ο πρόεδρος Μπαρόσο, βλέπετε ότι ελεύθερα εκφράζομαι. Είπε σε ένα φίλο του αρχηγό κράτους, Ιδού σου παρουσιάζω τον υποφαινόμενο. Ε, ε, μόνο αυτά είχα να αναφέρω. Σας ευχαριστώ. Merci. Alors, je retiens... Ευχαριστώ. Καλό, ε, κρατώ αυτή την έκκληση για την ιστορική διάσταση από την πλευρά του δικαίου. Ε, τι μας μένει. Ο Πιέρ Λεμουάν ε, αρχή συντάκτη τη πολιτικής Ευρώπης, ε, Ευρώπη πολιτική. Και μετά περιμένουμε να γίνει μια συζήτηση. Μετά από δύο απόψεις πολιτικών και δύο απόψεις ε, δικαιωμένων καθηγητών, εγώ θα κάνω την αντίστοιξη. Είμαι Ευρωπαίος δημοσιογράφος, ασχολούμαι με ένα μέσο το οποίο λειτουργεί ως διεπαφή μεταξύ των θεσμών και των επαγγελματιών που δουλεύουν ε, αυτό. Ε, ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να γίνει μάρτυρας και να θέτει και ερωτήσεις. Αυτό θα κάνω, ε, ελπίζοντας να είμαι πρακτικός, με στόχο να διευκολύνω τη συζήτηση με την αίθουσα, ώστε οι ερωτήσεις να είναι όσο γίνεται πιο πρακτικές και όσο γίνεται λιγότερο ε, ακαδημαϊκές. Ε, να πω ότι μεγάλος υπήκος και Ευρωπαίος υπήκος, γιατί όπως οι περισσότεροι από σας έχω δύο υπηκότητες, έμαθα ότι μία ήταν κάτω από την άλλη και ότι η ευρωπαϊκή υπηκότητα μου χορηγήθηκε γιατί έχω την υπηκότητα ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχω την ευρωπαϊκή ε, ηθαγένεια. Ελπίζω τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου να έχουν αυτή την ευρωπαϊκή προοπτική. Σήμερα, Μάη του 2010, έξι μήνες μετά από την έναρξη ισχύω, τι μου επιτρέπει να πω ότι ναι, είμαι Ευρωπαίος πολίτης, Ευρωπαίος υπήκος και στηρίζομαι στα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία παρουσιάστηκαν εδώ την προηγούμενη ώρα. Πρώτα, το δικαίωμα ψήφου. Έχω το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεστε στις ευρωπαϊκές και δημοτικές εκλογές του κράτους διαμονής που δεν είναι το κράτος καταγωγής μου. Αυτό είναι μεγάλη καινοτομία της συνθήκης του Μάστριχτ Πρέπει όμως να σχετικοποιήσουμε την εμβέλειά της γιατί το ποσοστό συμμετοχής των μεταναστών εκλεκτόρων είναι πολύ μικρό με εξαίρεση το Βέλγιο για, ευλόγους, ε, για ευνοήτους λόγους και επίσης ε, διότι στις ευρωεκλογέ ε, το ποσοστό αποχής ήταν 57% δηλαδή 2,5 ποσοστιαίες μονάδες παραπάνω από ότι το 2005 μετά από τις εκλογές ε, έχουν αυξηθεί τα συναισθήματα και ότι η αποχή δείχνει μία δυσπιστία γενικότερα απέναντι στην πολιτική αλλά όχι ιδιαίτερα ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή ερωτώ, δεν θα πρέπει να θέσουμε ερωτήματα ε, σχετικά με το πώς βιώνουν οι, ευρωπαϊκοί, οι Ευρωπαίοι πολίτες το θέμα της ηθαγένειας. Το θέμα τώρα της ελευθερίας και της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Το χώρο του Σέγγεν. Ο χώρος του Σέγγεν ε, κατήργησε τους ελέγχους ε, στα σύνορα, στα κοινά σύνορα των κρατών που έχουν προσυπογράψει τη συνθήκη της Σέγγεν και συμμετέχουν σε αυτό την 22 εκ των 27 ε, συν τρει συνδεδεμένε χώρε. Συνολικά 25. Οι συμφωνίε ε, του Σέγγεν που χρονολογούνται εδώ και 25 χρόνια μεταφράζουν τη βούληση ε, η Ευρώπη να έρθει πιο κοντά στου πολίτε ακόμη και αν συνήφθησαν μέσα από μία διακυβερνητική συμφωνία. Η ε, βραδύτητα της εφαρμογής είναι το χαρακτηριστικό. Δέκα χρόνια πέρασαν από το 1985 έως το 1995 ε, ε, ανάμεσα στην υπογραφή και την εφαρμογή και από τότε άνοιξαν σιγά σιγά τα σύνορα το 1993. Πέρασαν 17 χρόνια και θα ήθελα να κάνω και μία προσωπική παρατήρηση. Οι ουρές των αυτοκινήτων είναι πάντα εμφανείς στον δρόμο μεταξύ Βρυξελών και Παρίσι και Παρισίου που υποχρεώνουν τους ε, αυτοκινητιστές να πέσουν στα 10 χιλιόμετρα. Γιατί, για να τηρήσουν ένα λεπτό σιγής για να ε, ανάμνηση των θυμάτων των διαφόρων πολέμων ή των στήρων ε, αμφισβητήσεων για τα τσιγάρα ή το αλκοόλ. Ε, εγώ έχω σαφή αντίρρηση με αυτή την ε, συζήτηση η οποία δεν υπάρχει στο γερμανικό χώρο Γι' αυτό το επίπεδο, αν θα είναι το κοινοτικό, το περιφερειακό, το εθνικό, όλοι έχουμε την ευθύνη γι' αυτό το εμπόδιο που με ενοχλεί ως αυτοκινητιστή και πολύ ως Ευρωπαίου πολίτη. Πέρα από αυτή την προσωπική παρατήρηση, η συνθήκη της Λισαβόνας τροποποιεί τους νομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίνει στους πολίτες ένα χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας. Δικαιοσύνη, ασφάλεια, άσυλο, μετανάστευση απασχολούν κυρίως όλο και περισσότερο τους πολίτες και το βλέπουμε και στα ευρωβαρόμετρα που προανέφεραν οι συνάδελφοι. Και όπως υπολόγισε και ο καθηγητής κύριος Μόνα που άκουσα σήμερα το πρωί και που είναι τώρα εδώ και που τον άκουσα στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα, ο καθηγητής Μονά είπε ότι το Συμβούλιο ΔΕΗ που εξακολουθούμε να το αποκαλούμε ΔΕΗ, μολονότι έχει άλλο όνομα πλέον, JLS, το Συμβούλιο λοιπόν ΔΕΗ υιοθέτησε πάνω από 3.300 κείμενα από το 1999 και το τεράστιο πρόγραμμα της Στοκχόλμης που υιοθετήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο για την ε, αστυνομική συνεργασία, τελωνιακή συνεργασία, την ε, συνεργασία για ποινικά και αστικά θέματα, θέματα ασύλου, μετανάστευση πολιτική θεωρήσεων για τα έτη 2010-2014 έχει περίπου 170 προτάσεις που έχει αρχίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μετατρέπει σε προγράμματα δράσης. Η κυρία Μάλστρομ έχει πολλή δουλειά να κάνει. Άρα υπάρχει απόκληση ανάμεσα στο, στην φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ικανότητα των κρατών μελών να μεταφέρουν αυτούς τους κανόνες στο εθνικό επίπεδο επίπεδο χωρίς να μιλήσουμε για τις αντιστάσεις των εθνικών αρχών καθώς επίσης και τις αντιδράσεις των ατόμων που δεν είναι σωστά ενημερωμένα, που είναι καχύποπτα και όπου υπάρχει κίνδυνος παρερμηνίας και απόρριψης. Αντίθετα με αυτό το οποίο επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που άκουσα σήμερα το πρωί να ενισχύσει την αμοιβή εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών ε, μια εμπιστοσύνη η οποία ορίστηκε ως ε, εκ των όνου κάνευ. Άρα τι θα κάνουμε υποχρεωτικά ευρωπαϊκό εράσμους για όλους τους δικαστικούς και τους αστυνομικούς της Ευρώπης είναι τεράστια η ανάγκη κατάρτισης και καθότι η συνθήκη της Λισαβόνας ενισχύει το ρόλο των κρατών μελών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ένωση θα πρέπει να ευκολύνουν το έργο τους. Το διαζύγιο δεν αναφέρθηκε σήμερα. Είναι ε, επίπονη η διαδικασία το διαζύγιο. Οι σύζυγοι που πρέπει να εγκατασταθούν σε διαφορετικό κράτος μέλος από το δικό τους πρέπει να αντιμετωπίσουν και την την νομοθετική ζούγκλα. Το αντιμετωπίζουμε από το 2006 όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε καταθέσει νομοθετική πρόταση με στόχο να δώσει στους διαδίκους τη δυνατότητα να συμφωνήσουν για το εφαρμοστέο δίκαιο. Οι υπέρμαχοι και οι αντίπαλοι ε, αυτή τη ε, διαδικασία έχουν χωριστεί στα δύο. Ε, απαιτείται ομοφωνία και τον, το 2006 η Βιβιάν Ρέντνικ η οποία σήμερα ε, δεν έχει έρθει εδώ, δεν μπόρεσε να ε, βγάλει την παλιά πρόταση να χρησιμοποιείται μια ενισχυμένη διαδικασία για θέματα διαζυγίου. Και αν αυτή η ενισχυμένη διαδικασία ε, έπαιρνε σάρκα και αστά θα ήταν πρωτοφανές ε, φαινόμενο είναι νομικώς δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά δεν υπάρχει αρκετή πολιτική βούληση. Το διασυνοριακό λοιπόν διαζύγιο θα μπλοκάρει ακόμα για πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο πρώτα με ειδική πλειοψηφία έδωσε πράσινο φως για τους μηχανισμούς ενισχυμένης συνεργασίας. Στη συνέχεια τα 10 οι περισσότερα ε, ε, ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη θα ψηφίσουν ομοφόνος το σχέδιο συνεργασίας και θα μπορέσουν να αλλάξουν γνώμη υπόλοιποι και να ε, ενταχθούν και αυτά στην ε, διαδικασία αυτή τέταρτο και τελευταίο παράδειγμα μια, ενός οργάνου για την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Η πρωτοβουλία των πολιτών, είπαμε, η συνθήκη της Λισαβόνας δίνει μια νέα δυνατότητα συμμετοχής στους πολίτες, ε, ένα εκατομμύριο πολίτες από ένα συγκεκριμένο αριθμό κρατών. Η, τον περασμένο Νοέμβριο ξεκίνησε διαβούλευση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έδωσε την εντύπωση ότι θέλει να περιορίσει το νέο μέσο. Όμως μας λένε ότι το σχέδιο κανονισμού του Επιτρόπου για τα διοργανικά θέματα του κ. Σεύκοβιτς που ήταν εδώ σήμερα το πρωί προσπαθεί να ε, περιορίσει τις καταχρήσεις και να αποφύγει οποιοδήποτε υπερβολικό ακτός για τα κράτη-μέλη. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο από ό,τι φαίνεται προχώρησαν και μπορούμε να ελπίσουμε ίσως κάποια συμφωνία στο Συμβούλιο τον Ιούνιο και ίσως να κλείσει το θέμα πριν την εκπνοή της Ισπανικής Προεδρίας και έναρξη ισχύω αν όχι την 1η Δεκεμβρίου ε, επέτειο εφαρμογής της ε, συνθήκη της Αβώνας ή, εν πάση περιπτώσει, αρχές του 2011. Ε, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα γράμματα λαμβάνει μια εφημερίδα σαν τη δική μα. Θα μπορέσει η πρωτοβουλία των πολιτών να αντιστρέψει τη διαδικασία ε, των διατάξεων που λαμβάνονται για να αποφευθεί η αλία του τόνου στη Μεσόγειο. Θα μπορέσει η κοινωνία, η η πρωτοβουλία των πολιτών να αλλάξει την πορεία που παίρνουν διαστάσεις, παίρνουν θέματα όπως είναι ας πούμε η μπουρκα για ολόκληρο το σώμα και η απαγόρευση αυτής. Πώς οι πολίτες της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στις επόμενες πρωτοβουλίες των πολιτών. Αυτοί οι πολίτες έχουν τα ίδια δικαιώματα αλλά όχι τις ίδιες υποχρεώσεις με τους άλλους σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα μείνω εδώ για τις ερωτήσεις. Έχω την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια το 2000 έχει έναν μέτριο απολογισμό, αλλά θέλω να είμαι αισιόδοξο. Η ευρωπαϊκή ηθαγένεια πρέπει να οικοδομηθεί με πολλά πρακτικά βήματα, ακόμη και για τους αυτοκινητοδρόμους και ε, θα είναι το τσιμέντο ουσιαστικά της, του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Δεν συμφωνείτε με αυτή την άποψη. Merci. Ευχαριστούμε για ένα θέμα το οποίο ήταν ευρύτατο ήδη. Εσείς ανοίξατε και άλλες προοπτικές, ε, πάρα πολύ, πολλά θέματα για τα θεμελιώδη δικαιώματα, ε, πώς εμείς οι πολίτες, ευρωπαίοι πολίτες, οι υπήκοοι τρίτων χωρών πώς τοποθετούμαστε σε αυτά τα προβλήματα. Αυτό είναι το είδος της συζήτησης το οποίο μπορεί να προξενήσει χίλια όσα ερωτήματα. Ανοίγει η συζήτηση, όποιο θέλει να πάρει το λόγο. Βλέπω μια ερώτηση εδώ. Thank you very much. Ε, ευχαριστώ. Τρία ερωτήματα έχω. Ένα ερώτημα έχει να κάνει με θέματα που θα μας απασχολήσουν αύριο, αλλά προκύπτει από κάποιες ε, συστάσεις που προέκυψαν από την πρωινή συζήτηση και σε σχέση με το, με το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το πρώτο μου λοιπόν ερώτημα, έτσι γενικά, είναι πώς αντιμετώπισε το Κοινοβούλιο το θέμα των σχέσεων με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα αυτό, ετέθηκε σήμερα το πρωί, αλλά δεν νομίζω ότι απαντήθηκε πλήρως. Να σας υπενθυμίσω ότι το θέμα αυτό των σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο παρελθόν συζητήθηκε πάρα πολύ και μάλιστα με πολύ επικριτικά σχόλια από πλευράς Κοινοβουλίου και στη νέα συνθήκη της Λισαβόνας αυτό είναι ένα από τα θέματα κλειδιά για τις μελλοντικές διοργανικές σχέσεις. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω το Κοινοβούλιο πώς απεδέχθη αυτό το νέο όργανο, αυτή τη νέα κατάσταση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Νέο όργανο αυτό μεταξύ των υπολείπων. Και τώρα περνάω σε, στο θέμα που συζητούμε τώρα εδώ, θα ήθελα μια άποψη για το τι, τι γίνεται με αυτή την ασυνέπεια που υπάρχει μεταξύ του ρόλου του ε, δικαστηρίου που αναγνωρίζει και στον τομέα της ασφάλειας και της ε, εξωτερικής πολιτικής. Βλέπουμε, ας πούμε, στο 215, στο άρθρο της, ε, για την, της για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνει ρόλο, λοιπόν, ε, μετά από συζητήσει, νομικέ ε, ε, συμβολές κτλ. Μια που ήταν φιλογόμενο το θέμα αυτό. Δεν δίνει όμως κανένα ρόλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην, στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής λέει σαφώς στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη και στην Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ένωσης δεν υπάρχει ρόλος για το Κοινοβούλιο. Οπότε υπάρχει συνέπεια εδώ. Μιλάμε για ε, έλεγχο εκ των υστέρων και όχι εκ των προτέρων για την εκπόνηση της, πολιτικής, της εξωτερικής πολιτικής. Και επίσης, ναι, είναι σημαντικό να υπάρχει ασφάλεια, εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δυνάμει του 267, του άρθρου 267. Υπάρχει και η ε, πράξη για την ακύρωση. η οποία είναι ικανοποιητική τροποποίηση και αφορά το ρόλο των ε, ιδιωτών όπως λέει το 267, παράγραφος 3 αν θυμάμαι καλά, που μιλάει για τα για το δικαίωμα των πολιτών να προσφεύγουν έναντι των ευρωπαϊκών, ε, ενώπιον του δικαστηρίου για τις ευρωπαϊκές πράξεις. Αυτά από μένα προς το παρόν. Ευχαριστώ. Ε, could you answer the second question? Μήπως μπορείτε να επαναλάβετε τη δε... Μήπως μπορείτε να απαντήσετε, συγγνώμη, τη δεύτερη ερώτηση, κυρία Γκίλντ. Θα απαντήσω στην ερώτηση για το, ρόλο του Κοινοβουλίου ε, για την πολιτική, εξωτερική πολιτική. Υπάρχει ένα ρητό που λέει ότι η πολιτική είναι θέμα αρχών. Ε, στην εξωτερική υπηρεσία, στον σχετικό κανονισμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή προσυζήτηση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δύο όπλα. Την έγκριση του δημοσιο... της δημοσιονομικής γραμμής και τον κανονισμό του προσωπικού. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα τα χρησιμοποιήσουμε και τα δύο όπλα. Thank you. Ε, une autre question. Άλλη Στο μικρόφωνο, παρακαλώ. Εγώ είμαι από το... Από το Γερμανικό Πανεπιστήμιο. Θα ήθελα να μείνω στα θέματα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ένα ερώτημα έχω. Η χάρτα ονομάζεται Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Στο κείμενο όμως λέει δικαιώματα και αρχές. Και θα ήθελα να ρωτήσω όλους σας μήπως κάνετε κάποιο διαχωρισμό, γιατί νομίζω ότι τουλάχιστον από την γερμανική πλευρά οπτική, ότι δικαιώματα σημαίνει ότι μπορεί κανείς να πάει στο δικαστήριο κατευθείαν και να πάρει απάντηση. Είπε και ο κύριος πιο πριν για τα δικαιώματα που έχουν οι ιδιώτες. Αλλά θυμάμαι ότι μιλήσατε για το θέμα αυτό, οπότε κυρία Γκίλ δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να μου απαντήσετε εσείς. Και ένα δεύτερο σημείο, η χάρτα για τα δικαιώματα των πολιτών. Κάτι που μας φέρνει σε μια διαφοροποίηση μεταξύ πολιτών και μη πολιτών. Αλλά νομίζω ότι η χάρτα διαφοροποιεί μεταξύ τριών ομάδων. Μία είναι οι πολίτες γενικώ, άνθρωποι δηλαδή που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά μιλούμε για μη πολίτες, άνθρωποι δηλαδή που ζουν εκτός Ευρωπαϊκή Ένωση και μιλούμε και για Ευρωπαίους πολίτες. Μήπως λοιπόν μπορούμε να τα ξεδιαλύνουμε λίγο τα πράγματα, ειδικά σε ό,τι το κεφάλαιο για τα ε, δικαιώματα των, των πολιτών, των Ευρωπαίων πολιτών. Γιατί υπάρχουν τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και τα δικαιώματα των πολιτών εν γέννη. Eh, Θα απαντήσω στα ισπανικά. Η διάκριση μεταξύ δικαιωμάτων και αρχών. Έχετε δίκιο. Όταν συντάξαμε τη χάρτα στην εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ε, Κολονίας υπήρχε μία διάκριση μεταξύ των ε, δικαιωμάτων και των κατευθυντηρίων γραμμών. Και υπήρξαν αρκετοί στην ε, συνοδό εκείνη που αρχίσαμε να κάνουμε αυτή τη διάκραση υπήρχε και στο δεύτερο κεφάλαιο τίτλος 2 του Ισπανικού Συντάγματος, αλλά ένα μέρος της συνέλευσης δεν το δέχτηκε. Ε, το έβλεπε το πράγμα ότι οι αρχές είναι δικαιώματα δεύτερης κατηγορίας, ας πούμε και κάποιοι, τι είπαμε, αυτά είναι τα δικαιολογητικά κατά κάποιο τρόπο, είναι ε, δικαιώματα, αλλά κατευθυντήριες γραμμές που είναι πολύ σημαντικές γιατί μεταφέρονται στην νομοθεσία, αλλά ένα μέρος της συνέλευσης δεν το δέχτηκε και γι' αυτό το λόγο χρειάστηκε να βρούμε μια κάπως εξειδικευμένη νομική μορφή. Και λέμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις όπου πρόκειται για μια αρχή βάζουμε ε, και το στοιχείο λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές διατάξεις κάθε κράτους μέλους. Ε, ίσως θα ήταν καλύτερα κάτι άλλο, αλλά πολλές φορές ε, μπαίνει στη μέση η πολιτική και δεν βρίσκουμε και την καλύτερη νομική λύση για να επιληθεί το θέμα. Ευχαριστώ. Μια σύντομη απάντηση για τους, για τους πολίτες και τους μη πολίτες. Ναι. αν δείτε τη διατύπωση της χάρτας. Λέμε τα δικαιώματα των πολιτών, κάθε ε, πολίτης έχει διάφορα δικαιώματα, στο κεφάλαιο 5. Μετά έχουμε τη διατύπωση του ατόμου, άρθρο 41, στο οποίο αναφέρθηκα. Και η άλλη ομάδα που αναφέρεται ρητά είναι στην αλληλεγγύη για τους εργαζόμενους ή εκπρόσωποι εργαζομένων. Οπότε υπάρχει μια, ένας διαχωρισμός τριπλός. Μιλούμε για όλους, ε, πολίτες της Ένωσης αλλά και τρίτους, τρί, υπήκοοι τρίτων χωρών. Μετά έχουμε τους πολίτες της Ένωσης και μετά έχουμε τους εργαζόμενους. Και οι εργαζόμενοι συμπεριλαμβάνουν και πολίτες της Ένωσης και τρίτους ε, υπηκόους τρίτων χωρών που εργάζονται στην Ένωση. Αλλά δεν δέχομαι ότι υπάρχει σαφής αναφορά σε ε, υπηκόους συγκεκριμένων κρατών μελών γιατί αυτό, εδώ μιλούμε για πολίτες της Ένωσης. Ευχαριστώ. Ε, λυπάμαι, λοιπόν, αλλά πρέπει να σταματήσουμε εδώ, γιατί έχουμε και δεύτερη απογευματινή συνεδρία. Σας ευχαριστώ όλους πολύ, γιατί πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι παρεμβάσεις σας. Ε, κάποια θέματα θα μπορούσαν να έχουν αναφερθεί, θα τα θέσουμε όμως ε, τα ερωτήματα σε άλλη ευκαιρία, αλλά αυτή, αυτή συνεδρία πρέπει να την κλείσουμε.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 Υπότιτλοι AUTHORWAVE

Έχουμε αργήσει, έχουμε καθυστερήσει. Μπορείτε να καθίσετε για να ξεκινήσουμε. Ξεκινούμε με 40 λεπτά καθυστέρηση. Και πρέπει να προλάβουμε, να ανακάμψουμε λίγο. So, ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε την απογευματινή συνεδρία. Να ευχαριστήσω τους διοργανωτές που μας φιλοξενούν σήμερα, που μας υποδέχθηκαν τόσο γενναιόδωρα και που προετοίμασαν μια τόσο ενδιαφέρουσα ημερήσια διάταξη. Επίσης προσωπικά να ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μου δίνεται να προεδράψω τη συνεδρίαση σήμερα για το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο και την αντιμετώπιση των παγκοσμίων οικονομικών προκλήσεων, όπως λέει ο τίτλος. Είναι υψηλού επίπεδου το πάνελ μας. Αποτελείται από δύο άτομα που έχουν ε, αναγνωρισμένη καριέρα και σε, στην ευρωπαϊκή αλλά και στη διεθνή πολιτική και δύο ακαδημαϊκούς, τρεις ακαδημαϊκούς καλύτερα, γιατί ένας από τους πολιτικούς μας έχει διπλό πόστο, είναι και ακαδημαϊκός. Τρεις λοιπόν ε, ε, κατόχους του βραβείου Jean Monnet από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν λοιπόν τους δώσω το λόγο, να κάνω κάποια αρχικά σχόλια. Μετά από επίπονη, καμιά φορά και τραυματική, αλλά σίγουρα μακρόχρονη περίοδο, διαβουλεύσεων, διαπραγματεύσεων, επικυρώσεων, με διάφορα δημοψηφίσματα τα οποία δεν είχαν όλα θετική έκβαση ανάλογα το πώς βλέπει κανείς βέβαια το θετική έκβαση σε ένα δημοψήφισμα τώρα λοιπόν έχουμε μια ευρωπαϊκή συνθήκη ένας από τους βασικούς στόχους αυτού του εγχειρήματο ήταν να διευκολύνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικός παγκόσμιος παίκτη. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μια νέα Ευρωπαϊκή Συνθήκη αλλά έχουμε και μια καινούρια, πολύ, ένα πολύ καινούριο, διαφορετικό καλύτερα οικονομικό περιβάλλον σε σύγκριση με αυτό που υπήρχε όταν ξεκίνησε αυτή η μακρά διαδικασία της ε, όλης, της όλης ε, εκπόνησης της συνθήκης της Λισαβόνας. Να σας θυμίσω ότι αυτό που ξεκίνησε ως μια περιορισμένη κρίση ε, στις, στα subprimes των ΙΠΑ μετατράπηκε σε μια παγκόσμια οικονομική κρίση και σε μια κρίση που χτύπησε την πραγματική οικονομία με έναν τρόπο που δεν είχε ζήσει κανένας εδώ και δεκαετίες. Αυτό δεν έχει τελειώσει, δυστυχώς. Είναι μια κρίση που ξεκίνησε χτυπώντας πρώτα τις τράπεζες, τώρα χτυπάει τις χώρες. Και να σας θυμίσω ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει και πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες που ε, καθυστερούν λίγο να προκύψουν αλλά προκύπτουν. Οπότε φοβούμε ότι αυτό που είπε ο Ρόναλντ Ρίγκαν ότι δεν έχετε δει τίποτα ακόμα μάλλον μας αφορά λόγω αυτής της κρίσης. Η κρίση μάλλον δείχνει και το τέλος μιας εποχής, μιας μακράς εποχής που χαρακτηρίστηκε από οικονομική απελευθέρωση, κατά την οποία η απελευθέρωση των οικονομικών αγορών έδρασε ως ε, ρεζέρβα για την παγκοσμιοποίηση. Δυστυχώς αυτό σταμάτησε να συμβαίνει. Με την κρίση αυτή που περνούμε σήμερα έχουμε όχι μόνο το τέλος μιας εποχής αλλά και το τέλος μιας εποχής που μπορεί να μας οδηγήσει σε μια πολύ σημαντική αλλαγή στα όρια μεταξύ κρατών και αγορών. Και αυτό αφορά όχι μόνο τις χρηματοπιστωτικές αγορές, αλλά και αγορές ενέργειας, κλίμα. Ένας τομέας στον οποίο οι αγορές είχαν τη μεγαλύτερη αποτυχία. Το τέλος της κρίσης όμως δεν οδηγεί μόνο σε αυτή την αλλαγή μεταξύ ορίων, μεταξύ κρατών και αγορών. Από ό,τι φαίνεται, συμβάλλει και σε μια επιτάχυνση ε, μια συνεχιζόμενης τάσης προς ε, έναν πιο πολυπολικό κόσμο. Δηλαδή αλλαγή σε, πιο, σε έναν κόσμο που δεν είναι επικεντρωμένος στη δυτική του φύση. Με αυτή λοιπόν την, ε, τον κόσμο που αλλάζει ένα ενδιαφέρον ερώτημα θα ήταν ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ε, αυτή συνθήκη. Και τέλος, το τέλος της εποχής προκάλεσε και το τέλος του μήνα του μέλητος για το ευρώ. Κάποιοι από εμά, εγώ όχι, θεώρησαν ότι αυτός ο μήνας του μέλητος θα κρατούσε για πάντα και ότι οι δομές που είχαμε από το Μάστριχ που ήταν δομές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν μεταμοντέρνες που ε, δεν, δεν εμπίπτουν στους κανόνες της βαρύτητας ε, θα ήταν αρκετοί για να κρατήσουν τα πράγματα όπως ήταν για πάντα. Δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη κρίση που είχαν από την δημιουργία του ευρώ και τη μεγαλύτερη κρίση που είχαμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και δεκαετίες. Αυτά αρχικά. Τώρα έχουμε τέσσερις βασικούς ομιλητές και μετά μια σύντομη παρέμβαση από έναν συνάδελφο δημοσιογράφο. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Κάρελ Ντεχούχτ, που είναι Επίτροπο Εμπορίου, πρώην Υπουργό Εξωτερικών του Βελγίου. Να σα θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Εξωτερική Πολιτική ξεκίνησε με το εμπόριο και το εμπόριο παραμένει ουσιώδες κομμάτι της ευρωπαϊκής πολιτικής ε, εξωτερικών υποθέσεων. Κύριε Ντεχούχτ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ο Jean στο Ζαν Μονέ άρεσε πολύ, ήταν πολύ φιλόδοξος. Όποιος είναι λοιπόν φιλόδοξος και θέλει να βλέπει πράγματα, θέλει να κάνει και πράγματα. Σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν που αλλάζει, το κέντρο βάρους ε, αλλάζει προς την Ανατολή, Η Ευρώπη θέλει να παραμείνει βασικός παίκτη. Θέλει να παραμείνει βασικός παίκτη γιατί πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να εγγυηθούμε την ε, ευημερία μας, την ε, ευημερία της κοινωνίας, να προωθήσουμε τις αξίες μας και τα συμφέροντα και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός αυτής. Επειδή έχουμε την φιλοδοξία να, είμαστε, να ηγηθούμε του αγώνα για την εφαρμογή των, δικαιωμάτων, ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπεια. Είναι μια μεγάλη φιλοδοξία λοιπόν αυτή, αν το σκεφτεί καλά κανεί, και θα έπρεπε να είμαστε φιλόδοξοι. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε φιλόδοξοι και έχουμε όλα τα προσόντα για να εφαρμοστούν αυτές, να πραγματοθούν αυτέ οι φιλοδοξίε μα. Η φιλοδοξία του να, είναι κανείς, να γίνει κανεί κάτι πρέπει να ακολουθείται και από το να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να το επιτύχει. Ε, ο άνθρακας και ο χάλιβας ε, δεν είναι απλά ε, λέξεις. Το να επενδύσουμε στους πολίτες είναι πολύ περισσότερο από το να επενδύουμε σε διεθνείς διασκέψεις κλπ. Για να έχουμε λοιπόν μια επιτυχή πολιτική εμπορίου θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. Δεν μπορώ να σας πω πόσο Σημαντικό είναι να έχουμε ε, ανοιχτό εμπόριο για την ευημερία και την ενίσχυση των οικονομιών μας. Επίσης πρέπει να τονίσουμε και πάλι πόσο απαραίτητο είναι το εμπόριο για, την πολιτική και για τον πολιτικό και γεωπολιτικό ρόλο μας. Να δείξουμε ότι πολιτικός η ε, Ευρώπη είναι ανταγωνιστική τώρα, περισσότερο παραποτέ, σε μια περίοδο που μετά, η, μετά από, την, από τα χρόνια που χρειάστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την συζήτηση που έκανε για τη μεταρρύθμιση των α, δομών της, ο κόσμος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν καταλαβαίνει πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα έπρεπε να λειτουργήσει. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα να δείξουμε πώς λειτουργούμε, ότι σωστά λειτουργούμε, ότι υπάρχουν αποτελέσματα, ότι είναι σημαντικές οι προσπάθειες και κάνουν πραγματική διαφορά. Και γι' αυτό συνεργαζόμαστε, η στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντική. Η ευρωπαϊκή πολιτική δείχνει στον κόσμο ότι μπορούμε να μιλούμε με μία φωνή και μπορούμε να παίζουμε έναν ηγετικό ρόλο ακόμη και σε δύσκολες περιστάσεις. Με τη φωνή αυτή λοιπόν πάντα πιέζαμε τον, τις πολυτομιακές πολυφωνικές συμφωνίες. Αυτό είναι ένας από τους βασικούς μας στόχους που σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε μια ισορροπία για να είναι και επιτυχής ή να εφαρμοστούν επιτυχώς τα αποτελέσματα του γύρου της Δόχα. Σε έναν λοιπόν παγκόσμιο, παγκοσμιοποιημένο κόσμο αναζητώνται και παγκοσμιοποιημένες λύσεις. Ε, απελευθέρωση του εμπορίου στον ε, τομέα της ε, βιομηχανίας, των υπηρεσιών και της γεωργίας. Σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε επιθαρχημένοι για τις επιδοτήσεις, για τους κανόνες και να διευκολύνουμε το εμπόριο για λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Να διατηρήσουμε τους στόχους της Δόχα ώστε να είναι σωστός, ώστε να είναι όντως αναπτυξιακός ο αυτός. Πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μεγάλο ρόλο να παίξει στις διαπραγματεύσεις αυτές που τρέχουν εδώ και 9 χρόνια. Από το καλοκαίρι του 2008 οι συζητήσεις ε, καθυστερούν. Αλλά ε, επειδή δεν είμαστε εμείς αυτοί που προκαλούν την καθυστέρηση, σε αυτή τη φάση των διαπραγματεύσεων δυστυχώς δεν μπορούμε να δώσουμε το κλειδί για να προχωρήσουν. Το πακέτο που προέκυψε το 2008 δεν ικανοποιεί τη ΣΥΠΑ. Άλλοι διαπραγματευτές προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την, Αμερική, την Αμερικανική θέση ώστε να μην χρειαστεί να αλλάξουν ούτε τις δικές τους τάσεις. Και δεν είναι σαφές τι πρέπει να γίνει για να αρθεί αυτό το αδιέξοδο. Σαφές είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να σκεφτεί δημιουργικά και να δράσει αποτελεσματικά ώστε να υπάρξει συμφωνία όταν υπάρξει ένα ανοιχτό παραθυράκι. Ε, εφόσον η επικοδομητικότητα δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε και παραχωρήσεις. Το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι ισόρροπο και, και ε, ικανοποιητικό για όλους όσου βρίσκονται στο τραπέζι. Ε, αργότερα μέσα στην εβδομάδα θα πάω στο Παρίσι. Στα περιθώρια τη υπουργική διάσκεψη του ε, ΟΣΑ θα συζητηθεί το γύρο τη Δόχα. Και επίση υπάρχει και η φιλοδοξία του G20 για την ολοκλήρωση του γύρου της Ντόχας ώστε να υπάρξει όντως ένα σχέδιο μετά από αυτή την, ε, τις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση ε, ώστε οι διαπραγματευτές να μπορέσουν να καταλήξουν σε μία λύση. Όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει ότι ε, δεν μπορούμε από ουσία συμφωνίας από την Ντόχα να μην κάνουμε τίποτα σε ό,τι αφορά την κρατική απελευθέρωση. Η οικονομία μας χρειάζεται καλύτερη σύνδεση με τις αναδυόμενες αγορές, ειδικά μετά από την κρίση που αντιμετωπίζουμε. Η οικονομία πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί. Το εμπόριο είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει να δώσει την όθηση για την οικονομική ε, επάρκεια και να μπορέσει να ε, εξακολουθήσει να είναι λειτουργικό. Αν όλα αυτά καθυστερήσουν, τότε θα πρέπει ε, αυτός ο πολυτομιακός χαρακτήρας να δώσει αυτή την όθηση. Πρέπει να ολοκληρωθούν οι διμερεί συμφωνίε με την ε, Κορέα, πρέπει να ανοίξουμε διαπραγματεύσει με τη Σιγκαπούρη, να, να ξεκινήσει η διαδικασία με το Βιετνάμ, να δούμε κατά πόσο μπορούμε να βρούμε μέχρι το τέλο του χρόνου συμφωνία με την Κολομβία και το Περού. Και την προηγούμενη εβδομάδα ανοίξαμε τι ε, τις συζητήσεις με, την, ε, με χώρες Μέρκοσουρ. Τα οικονομικά ωφέλη και η αναγκαιότητα όλων αυτών των συμφωνιών ξέρω ότι πέρα από αυτά πρέπει να, δείξουμε ότι είμαστε στρατηγική εταίρεια, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δουλεύει παρά τους περιορισμούς που είναι όντως δύσκολοι και περίπλοκοι. Παρά την συνέχεια, τη συνεχεία αναφορά στα ΜΜΕ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει σωστές προσπάθειες, παρόλα αυτά οι προσπάθειες αυτές δείχνουν ότι η Ευρώπη έχει δυναμισμό. Για παράδειγμα, η γεωπολιτική σημασία της, ε, να, του να, να υπογράψει η Κορέα ενώ το, το κογκρέσο τον, ε, τον ΗΠΑ δεν είναι διατεθειμένο να μετακινηθεί από την ε, θέση του μας δείχνει ότι είναι πολύ πιο αργές στην, ή πιο, είναι λιγότερο φιλόδοξες οι προσπάθειες που γίνονται. Η πολιτική για το εμπόριο είναι πολιτική, είναι αυτή η πολιτική που μπορεί να επιφέρει μεγάλες αλλαγές. Και έτσι υπάρχει και πρόκληση αλλά και ευκαιρία, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και για τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ω ε, πρώην Υπουργός ε, και Ευρωβουλευτής ξέρω ότι είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να εμπλακούμε αποτελεσματικά στην εκπόνηση της σωστής πολιτικής. Μετά την συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε τον, το καθήκον να καταλήξουμε σε μια απόφαση, να λειτουργεί η πολιτική στην πράξη, να υποφελούνται και οι βιομηχανίες και οι καταναλωτές και να ενισχύσει τον παγκόσμιο ρόλο μας. Πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη το γενικότερο πλαίσιο. Έχουμε ένα νέο πλαίσιο τώρα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και τώρα είναι ο, το, ο χρόνος για να το χρησιμοποιήσουμε και να αντιμετωπίσουμε όντως αυτές τις προκλήσεις. Μιλούμε για ανοιχτό χαρακτήρα, για ανταγωνιστικότητα και δεν θα πρέπει να είμαστε ε, φιλόδοξοι υπέρ των δέων. Κυρίε και κύριοι, πρέπει να παραδεχτώ ότι δεν είμαι ε, σίγουρος, ε, πεπισμένος για αυτό που σας είπα στην αρχή. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων, αυτοί που θέλουν να είναι κάποιο και αυτοί που θέλουν να κάνουν κάτι. Αν αυτό είναι σωστό, αν αυτό αφορά κατηγορίες ανθρώπων και όχι γενικά φιλοδοξίες, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είμαι από αυτούς που εμπίπτουν στη δεύτερη κατηγορία. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ να είμαι κάποιο. θέλω να κάνω κάτι και να έχω τα καλύτερα αποτελέσματα από τη δουλειά που κάνω. Με είχαν καλέσει στην δυτική πτέρυγα του Λευκού Οίκου την προηγούμενη εβδομάδα για γεύμα. Και το θέμα δεν ήταν ε, η ιστορία του, της ε, τραπεζαρίας όπου α, ε, συμφάγαμε, αλλά το τι προέκυψε από αυτή την συνάντηση. Έγινε λοιπόν πολύ καλή δουλειά, υπήρξαν πολλές υποσχέσεις και ανέφερα ήδη τον ε, ρόλο μας ε, στο να παραμείνει ζωντανό ο γύρος της ε, Ντόχα. Οι διμερεί και οι περιφερειακές συμφωνίες, σας είπα ποιε είναι, για τις εταιρικές σχέσεις σας μίλησα, είμαστε στη διαδικασία διαπραγμάτευση με τις χώρες ΑΚΕ. Μπορούν λοιπόν να κάνουν την διαφορά για όλο το οικονομικό δυναμικό που υπάρχει και για όλου του εταίρους μα. Κάνουμε πολύ σκληρή δουλειά σε ό,τι αφορά τους δασμούς και τα μη, τα μη δασμολογικά προσκόμματα. Ε, έχουμε διάλογο με τους Κινέζους, με τους Ρώσους και, τους, και στο μέλλον θα ζητήσουμε και με τους Ιάπωνες. Επίσης πρόσβαση στην αγορά για πολύ συγκεκριμένους τομείς όπως η, ο τομέας των, της μηχανιών ή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για μένα η παραδοσιακή διπλωματία, η οικονομική διπλωματία και η πολιτική πάντα ήταν ε, θέματα που συνδέονταν άμεσα. Οπότε προσπαθώ να παίξω και εγώ το ρόλο μου ε, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνεργαζόμενος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, ώστε να έχουμε αποτελέσματα. Η εμπορική, αλλιώς η εμπορική πολιτική θα παρερμηνευθεί και θα υπονομευθεί. Εγώ είμαι πεπισμένος κυρίες και κύριοι ότι ε, με βάση και το οικονομικό και ακαδημαϊκό σας υπόβαθρο θα δείτε κι εσείς ποιος είναι ο ρόλος σας στον όλο μηχανισμό των διεθνών σχέσεων. Και γι' αυτό βασίζομαι σε εσά για να είσαστε οι τελευταίοι που θα παρερμηνεύσουν ή θα υποβαθμίσουν τη σημασία της οικονομικής και πολιτικής σημασίας που έχει το διεθνές εμπόριο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Πολύ σημαντικά αυτά που μας λέει ένας Ευρωπαίος Επίτροπος. Τι δράση τονίζει. Είναι γνωστό ποιο το πρόβλημα συνήθως με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι γίνονται ωραίοι λόγοι χωρίς να έχουμε αυτά αποτελέσματα. Τέλειο λοιπόν αυτό που ακούσαμε από πλευρά σα. Ο Μπαρόν Κρέσπον, ο επόμενο μα ε, ομιλητή, πρώην Ευρωβουλευτή, κατέχει την ε, έδρα Ζαμονέ στο Πανεπιστήμιο Καστίγια Λαμάντσα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Στην αρχή είπατε ότι είμαι και ακαδημαϊκός και πολιτικός, της αγωγικά σας σχόλια. Τώρα πράγματι κατέχω την έδρα Ζαμονέ και προτίμασα το παρθενικό μου έγγραφο περί οικονομικής διακυβέρνησης σε σχέση με τη Λισαβόνα και μετά με πήρε η κυρία Κυρός και μου είπε ότι θα πρέπει να μιλήσω ως πολιτικός. Επειδή ήμουνα και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που στράφηκα στο Μάστριχτ και ζήτησα από το Συμβούλιο να κάνει το μέγα άλμα προς τα σε θέματα ηθαγένειας, ενιαίου νομίσματος, συναπόφασης πολιτικών ομάδων και ούτω καθεξής. Και είχα και την ευθύνη εκπροσώπηση του Ευρωκοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για τη συνθήκη της Λισαβόνα, Νομίζω ότι έχω να σας δώσω κάποιες καλές συμβουλές. η προθεσμία ήταν η 3η Μαΐου σε σχέση με το έγγραφό μου. Αλλά η επανάσταση έγινε στις 9 Μαΐου. Επρόκειτο για μεγάλο άλμα προς τα εμπρός. Και πάλι. Κάποιοι ίσως κάνουν τη συγκρίση με το αποτέλεσμα της ε, συνέλευσης Φιλαδέλφειας από πλευρά συγχώνευσης ε, ευθυνών σε θέματα δημοσιονομικά, οικονομικά. Θα το δούμε, θα το δούμε αυτό. Απάντως είναι ένα βήμα προς τα εμπρός. και ομολογώ πως η κατεύθυνση είναι αυτή που αναφέρει το έγγραφό μου. Στο παρελθόν δεν ήμουνα μόνο ακαδημαϊκός, ήταν σύντομη η ακαδημική μου εμπορία και ο Ζαμ είναι το ίδιο. Ουδέποτε πήγε σε πανεπιστήμιο. Ιδού ένα εξαιρετικό παράδειγμα. τι προσθέτει η συνθήκη Λισαβόνας, τη Λισαβόνα σε θέματα οικονομική διακυβέρνησης. Πάνω απ' όλα, έχουμε το άρθρο 3 τη συνθήκη όπου προβλέπει το ευρώ. Προβλέπει ο Στόχο της Ένωσης. Πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Μετά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποτελεί πλέον ε, ένα πλήρη Τρίτον, η Ευρωζώνη καθίσταται ένα απόσπαστο μέρος των θεσμικών οργάνων. Υπάρχει μόλις το πρωτόκολλο 14 με τους κανόνες της Ευρωζώνης με εκλεγμένο πρόεδρο μεταξύ των μελών. Και τέταρτον, και όλα αυτά αναφέρονται στον πολύ ενδιαφέρον έγγραφο που ακούστηκε το πρωί, όχι από τον πρόεδρο Μπαρόσο, η στρατηγική ΕΕ 2020 που η Υπάρχουν δύο άρθρα το 121 είναι το ένα. Και το άλλο είναι το άρθρο 148. Δεν είναι καινούργια. Το 141 υπήρχε και στην ε, συνθήκη του Μάστερ. να υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Δηλαδή τώρα η Κομισιόν διαθέτει εξουσίες να στείλει προειδοποίηση προς ένα κράτος μέλος το οποίο δεν σέβεται τις διαδικασίες συντορισμού χωρίς να χρειάζεται εκ των προτέρων συγκατάθεση του Συμβουλίου. Και αν το Συμβούλιο λάβει απόφαση, μετά, μετά προχωρά χωρίς να χρειάζεται να λάβει υπόψη τη ψήφο της ενδιαφερόμενης χώρας. Επίσης προβλέπεται απόφαση για την κατάρτιση αυτών των κανόνων. Αυτή είναι η βελτίωση. Πολύ σημαντική αυτή η αναβάθμιση του άρθρου. Δεύτερον, ο τίτλος για τις διατάξεις ε, για τις χώρες για τις οποίες ε, το νομίζουμε το ευρώ. Άρθρο 36. Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία τη Οικονομικής και Ένωσης το Συμβούλιο δίνεται να λάβει μέτρα ειδικά για τα κράτη-μέλη που έχουν ως νόμισμα το ευρώ με στόχο την ενίσχυση του συνοδοτορισμού και τη υποπτία, ε, τη δημοσιονομική πεθαρχίας και έκδοση οικονομικών κατευθυντηρίων γραμμών από το Μάστερ τις είχαμε τις κριτήριες γραμμές, αλλά τώρα ενισχύεται το θέμα της δημοσιονομικής πειθαρχίας για τα μέλη της Ευρωζώνης. Υπάρχει και το άρθρο 138 που λέει ότι και η Κομισιόν και η Ευρωευρωζώνη δίνεται συγχωνεύσονται εκπροσώπηση του ευρώ στα διεθνή, στους διεθνείς οργανισμούς. Αν ληφθεί τέτοια απόφαση από την Ένωση, τι σημαίνει αυτό, ότι δεν θα έχουμε πλέον στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κατακαιρματισμένη εκπροσώπηση. Θα ήταν μεγάλο άλμα προς τα εμπρός. Να δούμε τώρα πώς έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Συνέταξα το έγγραφό μου στα τέλη Απριλίου Ξέρετε τι συνέβαινε. Τρεις ήταν οι επιλογές κυρίως. Η πρώτη ήταν να εκδιωχθούν οι ένοχοι. Κάποιοι εξέχοντες ε, καθηγητές πήγαν στη Γερμανία και μίλησαν για εκδίωξη της Ελλάδας. Μετά την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Γαλλία, όλους. Με εξαίρεση τις Παρθένες. άκουσα και άλλες προτάσεις. Διάβασα στην εφημερίδα, γαλλική εφημερίδα Le Monde να διώξουμε τη Γερμανία γιατί είναι υπερβολικά καλή η απόδοσή της. Άλλη πρόταση. Αναβαθμίζουμε τη Γερμανία και τις χώρες Μπενελούξ, ιδίως τις κάτω χώρες, γιατί είναι διαφορετικές. Ένα είναι το κοινό στοιχείο σε αυτές τις προτάσεις. Είναι έκκληση για συλλογική αυτοκτονία και καταστροφή της Ευρώπης. Συμφωνώ απόλυτα με τον πρώην καγκελάριο Χέλμουντ Σμιτ πως άμα δεν το είχαμε το ευρώ τότε οι αγορές και οι κερδοσκόποι θα έπαιζαν ποδόσφαιρο με τα νομίσματά μας. Δεν θα χρειαζόταν καν να πάει κανείς στην Νότια Αφρική. Αυτή είναι η πρώτη πρόταση Άλλη πρόταση, την ανέφερε ο πρόεδρος Μπαρόσο το πρωί, όταν μίλησε για κυρώσεις. Κίνητρα για συμμόρφωση, έτσι τα αποκάλυψε. Πολύ λεπτή και κομψή η έκφρασή του. Αυτή τη στιγμή ήδη υπάρχουν διατάξεις για κυρώσεις και εφαρμόζονται κυρώσεις, επιβάλλονται κυρώσεις για τις απάτες ας πούμε, στη Γεωργία. Επιβάλλονται σε κάθε κράτος μέλος, προβλέπονται πρόστιμα. Το μοναδικό πρόβλημα ποιο είναι. Αυτό που οι οικονομολόγοι αποκαλούν προκυκλικές συνέπειες. Είναι σαν να προχωρούμε σε πόλεμη κατάσταση. Είναι λεπτό, πάντως η συνθήκη το προβλέπει και βεβαίως και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Τρίτο στοιχείο, βελτίωση της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Προσέξτε την απόφαση του ΕΚΟΦΗΝ της 9 η Μαΐου. Πρώτο σημείο, του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών. Ο πρόεδρος Μπαρόσο εξήγηλε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό σύνταξη κάποιες προτάσεις. Δεν θα πρέπει να τροποποιήσουμε τη συνθήκη, να την εφαρμόσουμε τη συνθήκη πρέπει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι κάθε φορά που έχουμε μία ύφεση στην Ένωση λέμε «Α, πρέπει να τροποποιήσουμε τη συνθήκη». Και τελικά είναι χαζό, διότι πριν από την ύφεση είναι που θα πρέπει να προβληματιστούμε. Από αυτή την άποψη πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να τροποποιήσουμε τη συνθήκη. μετά, ε, συντονισμός οικονομικής πολιτικής. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση αυτή που κυκλοφορεί εδώ και καιρό. Πράγματι, θέλουμε πραγματικά την νομισματική ένωση. Ε, τότε το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συντονίσουμε τις οικονομικές μας πολιτικές και τις δημοσιονομικές μας διαδικασίες. Τίθεται θέμα χρονοδιαγράμματος. Χρειάζεται τροποποίηση συνθήκης διότι αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει πολύ κακό κλίμα σε θέματα εθνικής κυριαρχίας κτλ. Οπωσδήποτε χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματικό συντονισμό όλων των μελών ε, της Ευρωζώνης. Τρίτον, διαχείριση της ε, κρίσης του ευρώ. Η απόφαση που ελήφθη για σύστημα εγγύσεων από το ΕΚΟΦΗΝ ήταν ένα πολύ σημαντικό πολιτικό βήμα. Το επόμενο βήμα τώρα ποιο είναι. Η δημιουργία Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Βρίσκεται γι' αυτό υπό συζήτηση. Να επιβληθούν κάποια τέλη για να βρεθεί μία λύση, μία διέξοδος από την παγκόσμια κρίση. Ακούγεται γι' αυτό. Υποσυζήτηση βρίσκονται όλα αυτά, άρα δεν μπορώ να σα δώσω περαιτέρω λεπτομέρειες. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι ορθή κατεύθυνση για διέξοδο από την κρίση. Υπάρχει λεγόμενη πρόταση Blue Bone που έγινε στον Μπρούγκελ από δύο εξέχοντες οικονομολόγους, ένα Γάλλο και ένα Γερμανό, μου φαίνεται σοφή αυτή η πρόταση. Έκδοση ευρωομολόγων μέχρι το όριο του 60% που το προβλήμα η δική του Μάστρεχτε και μετά το να πάμε παραπέρα αυτό θα είναι ευθύνη της κάθε κυβέρνησης ξεχωριστά. Αν ακολουθηθεί αυτή η οδός τότε θα δημιουργήσουμε τη μεγαλύτερη αγορά ομολόγων στον κόσμο. Πιστεύω ότι αυτό θα ενίσχυε την Ευρώπη. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει θετικό αντίκτυπο βεβαίως στις διαπραγματεύσεις της Ντόχα. Πάντως τι είδα την περασμένη εβδομάδα. Ο Επίτροπος Τεκιούχτ, το αντίστροφο μάλλον. Τα κράτη-μέλη το αναλάβουν μέχρι 60% και μετά να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βλέπω επικίνδυνο, λέει ο κύριος Μπαρόν Κρέσπο. Βλέπω ότι είστε πρώην μέλος ε, του Συμβουλίου. Ε, το βλέπουμε από αυτά που είπατε. Δεν νομίζω να περνούσε και κάτι τέτοια ιδέα όμως. Υπάρχει και η δέσμη βεβαίως οικονομικών ρυθμίσεων. Και υπάρχουν οι προτάσεις Λαγοζιέρ. Θα πρέπει να τις παρουσιάσουμε και ενώπιον του G20 Υπάρχουν και ρυθμίσεις για τα hedge funds. Υπάρχει σχετική οδηγία που πέρασε την περασμένη εβδομάδα μόλις στο Συμβούλιο. Καταψήφισε το νούμερο Βασίλειο που δεν αντιλαμβάνομαι, αλλά θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούλιο. Αυτό είναι σημαντικό. Κατά τη γνώμη μου, Και δεν θα ξεπεράσω το τεταρτάκι. Η συνθήκη της Λιζαβόνας μπορεί να μας βοηθήσει σε θέματα οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης. Όπως γνωρίζετε, οι συνθήκες, οι συνθήκες είναι και τα συντάγματα συντάγματα, αλλά υπάρχει πολιτική βούληση και οι πολιτικές αποφάσεις δεν μπορούν να μπουν σε ένα μόνο έγγραφο. Είναι μέρος της ε, διαδικασίας όμως πράγματι δεν ισχύουν αυτά που ίσχυαν στο παρελθόν και το πρωί ακούστηκε αυτό. Γίνεται λόγος για αλλαγές στις θεσμικές ισορροπίες. Τώρα έχουμε πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για δυόμιση χρόνια. Μεγάλη αλλαγή, σπουδαία αλλαγή. σε αυτή, τη νέα, σε αυτή τη νέα κατάσταση ζούμε όπου έχουμε σύνοδο κορυφή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κάθε μήνα. Μια σύνοδο κορυφή το μήνα. Όπου ο πρόεδρο Βάρα Μπόι στην ημερήσια διάταξη πάντα συμπεριλαμβάνεται οικονομικά ζητήματα. Αν μου το επιτρέπει ο Κάρλ Ντεγκιούχτ, να πω ότι οι Βέλγοι στο δικό τους επίπεδο ε, κάνουν μεγάλη συζήτηση αλλά σε επίπεδο ευρωπαϊκό μιλούν με μία, με μία φωνή. Σαν τον Κάρολο τον Πέμπτο. Τώρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι πλέον θεσμικό όργανο. Για να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον της κοινωτικής μεθόδου και πώς διαμορφώνεται ο νέος ρόλος της Κομισιόν, που δεν μπορεί να είναι ο ίδιος όπως στο παρελθόν. βρισκόμαστε στα μέσα αυτή τη περίπλοκη διαδικασία, διότι η Κομισιόν εξασφαλίζει κάποιε πολύ σημαντικέ εξουσίε χάρη στη συνθήκη τη Λισαβόνα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πάντω καθίσταται κύριο παίκτη στην Ένωση. Και όχι μόνο για θέματα εξωτερικών υποθέσεων, για θέματα εκπροσώπηση, αλλά και ω προ τα μέσα και ω προ τι ε, καθημερινέ αποφάσει για οικονομικά ζητήματα. Και ένα τελευταίο στοιχείο, αλλά εξίσου σημαντικό, καταλήγοντας. Από τη στιγμή που αποφασίσαμε, την, ε, αποφασίσαμε ε, να ακολουθήσουμε κοινή μοίρα με την δημιουργία του ενιαίου νομίσματος, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η νομισματική ένωση δεν είναι δυνατόν να διαρκέσει στην ιστορία. Κάποια παραδείγματα υπάρχουν. Μακροπρόθεσμα χρειάζεται και οικονομική ένωση και πολιτική ένωση. Αυτό είναι το κύριο δίδαγμα στο οποίο καταλήγουμε. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ίσως και να ζούμε ιστορικές στιγμές, διότι κατά διάρκεια αυτών των μηνών ελήφθησαν κάποιες ιστορικές αποφάσεις. Ελπίζω δηλαδή. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much Ευχαριστώ πολύ, διότι θέσατε πολλά ενδιαφέροντα και εύστοχα ερωτήματα για οικονομική διακυβέρνηση, ειδικά όσον αφορά την Ευρωζώνη και διότι τηρήσατε και το χρονικό όριο, το χρονικό περιορισμό που ευγενικά προσπάθησα να πείσω τους ομιλητές να τηρούν. Διαφορετικά θα... δεν θα προλάβουμε όχι καφέ να πιούμε, αλλά ούτε καν το βραδινό μας. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Στέφαν Γκρίλερ ο εδραζόμονες στο Πανεπιστήμιο της ε, Βιέννης για οικονομικά θέματα και επιχειρήσεις, ο κύριος Γκρίλα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα δείτε στην οθόνη το πρόγραμμα, αλλά μου ζητήθηκε να συντομεύσω λίγο λόγω χρονικών περιορισμών και αποφάσισα να κρύψω πολλές από τις διαφάνειες και να σας παραπέμψω στο έντυπο που υπάρχει που μπορείτε να βρείτε έξω μετά από την ομιλία μου και να ε, περιορίσω και τις παρατηρήσεις μου για την οικονομική σταθερότητα των κρατών μελών. Με μία εξαίρεση βέβαια. Επιτρέψτε μου με όλο το σεβασμό, θα ήθελα να διαφωνήσω για την ποιότητα του νέου πλαισίου για την οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι, πιστεύω ότι είναι πολύ αδύναμες οι προϋποθέσεις και ο ανοιχτός, η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού είναι πολύ αδύναμες για να αντιμετωπίσουν την κρίση. Τίποτα βέβαια δεν ε, μιλά κατά της ευρύτερης, ενός ευρύτερου συντονισμού, αλλά τα κράτη-μέλη διστάζουν και τίποτα δεν γίνεται και αυτό αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια. Οπότε υπ' αυτή την έννοια πιστεύω ότι η συνθήκη της Λισαβόνας δεν μας δίνει νέο έδαφος. Ούτε τα νέα μέσα είναι επαρκή. Υποσχέθηκα βέβαια να μην τα πω αυτά, αλλά αυτό που δεν θα τηρήσω, αυτό το οποίο θα περά, που θα πω, είναι οι προκλήσεις, οι οποίες ε, που ε, αντιμετωπίζουν, ε, τις οποίες μάλλον αντιμετωπίζει η δυναμική της παγκόσμιας οικονομίας. Ήδη ο Επίτροπος Δικούχτ είπε ότι η Επιτροπή ήδη το 2006 εξέδωσε ανακοίνωση για την Ευρώπη, παγκόσμιο ανταγωνισμός ε, με τον υπόλοιπο κόσμο και αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα και τονίζει δικαίως ότι οι προκλήσεις που ε, αντιμετωπίζει η Ευρώπη όχι μόνο στα πλαίσια ανταγωνισμού με τη ΣΥΠΑ και με την Ιαπωνία αλλά και με τις χώρες BRIC δηλαδή Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και άλλες ε, χώρες και επίσης υπάρχει και το πλαίσιο ότι ο γύρος της Ντόχα δεν επέτυχε ε, οπότε οι πολυμερείς λύσεις, ακόμη και αν είναι πρώτη προτίμηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν περιορισμένη προοπτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλο και περισσότερο επιλέγει διμερείς λύσεις η Ένωση ε, ως προς ε, κάτι το οποίο κάνουν και οι κύριοι ανταγωνιστές, είπα και η Ιαπωνία, ή με λύσεις τη νέα γενιά ε, των συμφωνιών ελευθερ... εμπορίου, ελευθέρων συναλλαγών που καλύπτουν και μη οικονομικά θέματα αλλά και καλύπτουν και νέους χώρους όπως την Κορέα, Μερκοσούρ. Όλα αυτά όμως ήδη αναφέρθηκαν. Είναι σαφές ότι αν αυτή είναι η πρόκληση, δηλαδή ότι υπάρχει μια νέα δυναμική στην παγκόσμια οικονομία, τότε είναι σημαντικό το νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών να ενισχυθούν. Ε, και έχουμε νομικούς μηχανισμούς που είναι αποτελεσματικοί για εξωτερική δράση. Αυτό που ισχυρίζομαι είναι ότι η συνθήκη της Λισαβόνας κάνει πολλά προς την κατεύθυνση αυτή. Όπως ξέρετε όλοι, η συνθήκη γενικώ πως κωδικοποιεί και αποσαφηνίζει τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό ισχύει και για τις εξωτερικές αρμοδιότητες μεταξύ αυτών και τις αποκλειστικές εξωτερικές αρμοδιότητες και πιο, πιο συγκεκριμένα την κοινή εμπορική πολιτική και τις διεθνείς συμφωνίες, δηλαδή το δικαίωμα σύναψης διεθνών συμφωνιών. Είναι πολύ μικρά τα γράμματα. Εδώ δεν το κατάλαβα ότι θα ήταν τόσο μακριά η οθόνη. Το θέμα μου λοιπόν στη διαφάνεια αυτή έχει το, είναι το εξή. Υπάρχει μεγάλη διαφορά εάν μια αρμοδιότητα είναι αποκλειστική ως προς τη φύση της ή αν είναι επιμερισμένη. Αυτό που αποσαφηνίζει η συνθήκη της Λισαβόνας είναι ότι η διευρυμένη κοινή εμπορική ε, πολιτική είναι αποκλειστική ως προς τη φύση της και αυτό σημαίνει ότι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το δικαίωμα δράσης και τα κράτη-μέλη δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να αναλάβουν δράση χωρίς την Ένωση. Αυτό είναι διαφορετικό στον τομέα της επιμερισμένης αρμοδιότητας. Τούτου λεχθέντος, το πιο η πιο εντυπωσιακή μεταρρύθμιση αφορά το δικαίωμα της Ένωσης να συνάπτει διεθνείς ε, συμφωνίες στον τομέα της κοινή εμπορικής πολιτικής. Και αυτό που βλέπετε στη διαφάνεια με κόκκινα γράμματα είναι το ουσιαστικό. Δηλαδή από τώρα και στο εξή, δηλαδή από την 1η Δεκεμβρίου και μετά. Η Ένωση όχι μόνο έχει αποκλειστικό δικαίωμα να συνάπτει συμφωνίες για τα αγαθά και το εμπόριο, αλλά και αποκλειστικό δικαίωμα να συνάπτει συμφωνίες για εμπόριο στον τομέα των υπηρεσιών και εμπορικές πτυχές δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και συμφωνίες για τις ε, ξένες άμεσες επενδύσεις. Αυτό είναι το μεγάλο άλμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σχετικό δηλαδή πλαίσιο το οποίο αφορά τις παγκόσμιες προκλήσεις για να ξεκαθαρίσω τι θέλω να πω. Θα πρέπει να θυμόμαστε πώς είχαν τα πράγματα πριν. Δηλαδή, αυτό που αποκαλώ εγώ το τέλμα του ΠΟΕ με βάση και μια απόφαση του ΔΕΚ του 1994 και τα πράγματα έγιναν και χειρότερα με τη συνθήκη της νίκαιας, αλλά δεν θα μπω σε αυτά για να συντομεύω. Το δικαστήριο το 1994 μας είπε ότι οι υπηρεσίε, ε, το εμπόριο στις ε, υπηρεσίε δεν είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ήταν τότε. Και ούτε και η προστασία των ε, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Μόνο κάποια τμήματα εμπίπτουν στην κοινή εμπορική πολιτική. Ω αποτέλεσμα, η συμφωνία του ΠΟΕ έπρεπε να συναφθεί ω επιμερισμένη, μεικτή αρμοδιότητα, δηλαδή και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κράτη-μέλη η Ένωση μπορεί να ψηφίσει για τα κράτη-μέλη στον ΠΟΕ αναλόγως του πεδίου δράσης και ότι οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις και αυτό βεβαίως εμποδίζει της Ευρωπαϊκή Ένωση διότι υπάρχουν πολλές τεράστιες ε, συμφωνίες και διαπραγματεύσεις που είναι στην αρμοδιότητα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μέλων. Τώρα τα πράγματα άλλαξαν διότι ό,τι ανέφερα, δηλαδή αγαθά, υπηρεσίες, δικαιώματα διανοητικής ε, ιδιοκτησίας και άμεσες επενδύσεις, αλλοδαπές άμεσες ε, επενδύσεις εμπίπτουν στη νέα εμπορική πολιτική και είναι πλέον αποκλειστική αρμοδιότητα και διευρύνεται. Επομένως είναι ε, πιο απλά τα πράγματα, πιο αποτελεσματική η πολιτική αυτή και πιο σαφής και τολμώ να πω ότι αυτή η νέα αρμοδιότητα καλύπτει σχεδόν όλο το πρόγραμμα του ΠΟΕ, δηλαδή με εξαίρεση τις μεταφορές, αλλά δεν θα επεκταθώ σε αυτό το προκλητικό συμπέρασμα είναι το εξή ότι με βάση τη νέα συνθήκη θα μπορούσαν τα κράτη μέλη να ε, σταματήσουν να παύσουν τη συμμετοχή τους στον ποε. δεν ισχυρίζομαι κάτι τέτοιο απλά το λέω για να σας πω πόσο ευρεία είναι η μεταρρύθμιση. Και αφού καλύπτεται πλέον το πρόγραμμα του ΠΟΕ, δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά καλύπτεται και ένα μεγάλο πεδίο της νέας γενιάς ε, συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών. Ε, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και ρήτρε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η προστασία του περιβάλλοντος. Όλα εμπίπτουν πλέον στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης. Και κάτι περισσότερο, οι ξένες ε, άμεσες επενδύσεις. Και θα έλεγα ότι αυτό είναι αμφιλεγόμενο. Ε, υπό την ευρία έννοια και αυτές είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης και όχι μόνο πρόσβαση στην αγορά, αλλά περί κανόνες για την προεγκατάσταση και μετά την εγκατάσταση και μπορούν να συμπεριληφθούν τέτοιοι κανόνες σε συμφωνίες που συνάπτει μόνη της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει το πρόβλημα βέβαια των επενδύσεων χαρτοφυλακίου που ξαναθέτει το θέμα των μεικτών συμφωνιών. όλα αυτά όμως εδώ έχουμε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός και Συνολικά μπορώ να πω ότι η μεταρρύθμιση αυτή είναι η πιο, της κοινή εμπορικής πολιτικής είναι η πιο σημαντική διότι ε, περιορίζει την ικανότητα των κρατών μελών να συνάπτουν συμφωνίες. Η μεταρρύθμιση λοιπόν αυτή μαζί με τη μεταρρύθμιση στον τομέα ελευθερίας δικαιοσύνης και ασφάλειας, αυτές οι δύο, εμπορικής πολιτικής δηλαδή δικαιοσύνης και ασφάλειας, είναι οι μεγαλύτερες ουσιαστικά μεταρρυθμίσεις του ουσιαστικού κοινοτικού δικαίου, ενουσιακού πλέον δικαίου. Το δεύτερο σκέλος τώρα είναι ότι όχι μόνο ότι υπάρχει διεύρυνση των αρμοδιοτήτων, αλλά αυτό σημαίνει ότι συμμετέχει ισότιμα με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναφέρθηκε και το πρωί και το απόγευμα το θέμα αυτό και ισχύει και για την εξωτερική δράση. Με δεδομένα τα χρονικά όρια που έχω όμως, δεν θα εξετάσω τα πάντα που υπάρχουν στη διαφάνεια αυτή. Απλά θα σας παραπέμψω στο συμπέρασμα, στο τέλος. Είναι αρκετά σαφές ότι όλα όλες αυτές οι συμφωνίες εμπορικής πολιτικής που είναι πλέον αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζονται τη συνένεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή, στο μέλλον δεν θα υπάρξουν εμπορικές συμφωνίες χωρίς τη συνένεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και όπως αναφέρθηκε ήδη, προφανώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, όχι μόνο για τις συμφωνίες εμπορικών συναλλαγών, αλλά έχουμε και τις συμφωνίες SWIFT, αλλά το ίδιο θα συμβεί και ε, στο εξωτερικό εμπόριο. Το τρίτο κομμάτι τώρα είναι το εξής. Υπάρχει αυξημένη... Ένα ένας αυξημένος μηχανισμός, ένας ενισχυμένος ε, μηχανισμός. Υπάρχουν ενισχυμένες διατάξεις περί ε, συνεκτικότητας για την εξωτερική δράση συνολικά. Αυτό οφείλεται κυρίως στο κομμάτι 5 της συνθήκης της Λισαβόνας για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνδέει σχεδόν όλες τις εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο την κοινή εμπορική πολιτική, αλλά και την αναπτυξιακή συνεργασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και άλλους τομείς. Με μεγάλη εξαίρεση βέβαια την πολιτική εξωτερικών και κοινή πολιτική ασφάλειας, η οποία δεν διέπεται από τον τίτλο 5 της συνθήκης και έχει ε, τις συνέπειές του αυτό ως προς τα όργανα, τις διαδικασίες και νομικές συνέπειες βέβαια για τα ε, διάφορα μέτρα θέση σε εφαρμογή. Είναι αρκετά θεαματική λοιπόν η μεταρρύθμιση, χωρίς όμως να απαλήφει τις διαφορές μέσα σε αυτά τα συγκεκριμένα πεδία δραστηριοτήτων. Αντιμετωπίζουμε ακόμα, εξακολουθούμε δηλαδή, να αντιμετωπίζουμε σημαντικές διαφορές ως προς τις αρμοδιότητες, τύπους αρμοδιοτήτων, ως προς τις διαδικασίες, πώς δηλαδή μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή δευτερογενής νομοθεσία, ως προς τα όργανα και βεβαίως ως προς τα θέματα ουσίας και επικαλύψεων. Εξακολουθεί λοιπόν να υπάρχει και με τις νέες διατάξεις, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη ανάγκη συνεκτικότητας και η, η συνθήκη προσπαθεί να αντιμετωπίσει και αυτά τα θέματα. Πρώτον, πρέπει να ξέρουμε ότι στη συνθήκη της Λισαβόνας βρίσκουμε τη γενική διάταξη, οι οποίες, οι γενικές διατάξεις μάλλον, οι οποίες αφορούν όλο το εξωτερικό σκέλος δράσης, όχι μόνο την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας που ήδη υπήρχε. Τώρα, οι αρχές αυτές που ε, αναφέρονται ρητά στην διαφάνεια ισχύουν για ολόκληρη την εξωτερική δράση. Και αυτό σημαίνει και είναι σημαντικό ότι από τώρα και στο εξής θέματα ας πούμε προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, πρόθεσης της δημοκρατίας, προστασίας του περιβάλλοντος δεν είναι μόνο θέμα ειδικών ε, συμφωνιών ή ειδικών δραστηριοτήτων με βάση ειδικέ διατάξεις ισχύουν σε κάθε περίπτωση και να θυμηθείτε επίσης ότι και το Κοινοβούλιο, ε, μεταξύ άλλων, έχει αναλάβει την προάσπισή τους. Άρα αυτές οι διατάξεις περιορίζουν κατά κάποιο τρόπο τις αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων τομέων εξωτερικής δράσης, ενώ παράλληλα πολιτικοποιούν τις εξωτερικές δράσεις ε, που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει επίσης και μια οργανωτική κατά κάποιο τρόπο πτυχή του όλου θέματος. Η συνθήκη περιλαμβάνει κάποιες διατάξεις περί συνεκτικότητας μεταξύ των διαφόρων τομέων εξωτερικής δράσης και καλεί το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον είπα το εκπρόσωπο να διασφαλίσουν αυτή τη συνεκτικότητα και να συνεργαστούν προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτή είναι η διατύπωση του νέου άρθρου 21 της ε, συνθήκης. Παράλληλα, η συνθήκη κατανέμει και τις αρμοδιότητες εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δηλαδή, ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί να λάβει δεσμευτικές αποφάσεις για στρατηγικά συμφέροντα και στρατηγικούς στόχους της Ένωσης, όχι μόνο σε θέματα ΚΕΠΑ, αλλά σε όλους τους τομείς εξωτερικών δράσεων. Με την πρώτη ματιά δηλαδή αυτό φαίνεται πολύ εντυπωσιακό. Αν το δει κανείς πιο προσεκτικά, σχεδόν τελείωσα, αν το δει πιο προσεκτικά κανείς μπορεί να αναρωτηθεί, είναι ε, δίκαιη αυτή η συνεκτικότητα. Αν δείτε τα διάφορα όργανα, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον ΥΠΑ, το εκπρόσωπο, δεν είναι και τόσο προφανές ότι όλοι αυτοί θα έχουν τα ίδια καθήκοντα. Είναι προφανές ότι θα υπάρξουν συγκρούσεις. Και αν δεν καταστεί δυνατόν να καταλήξει κανείς σε κάποια συνένεση μεταξύ αυτών Μια πιο προσεκτική λοιπόν ανάλυση δείχνει ότι αυτή η εικόνα δεν είναι τόσο ωραία έτσι, αυτή η εικόνα που προκύπτει και αν δεχτούμε ότι υπάρχει αναπόσπαστη επικάλυψη κατά κάποιο τρόπο μεταξύ πολιτικής και οικονομίας και αν θεωρεί κανείς, αν λάβει υπόψη κανείς ότι η συνθήκη της Λισαβόνας ε, παρουσιάζει μια νέα δομή ε, στην κοινή εξωτερική πολιτική και κοινή ασφάλεια, πολιτική ασφάλεια, τότε θα προκύψουν περαιτέρω αμφιβολίες. Αυτό είναι έτσι μια σύντομη ματιά ε, σχετικά με τις διατάξεις περί εξωτερικής πολιτικής. Από μια έχετε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος στο δικό του επίπεδο υπ' αυτή την ιδιότητα θα διασφαλίσει την εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης για θέματα που αφορούν την κοινή εξωτερική πολιτική και κοινή πολιτική ασφάλειας. Εδώ λοιπόν έχουμε το Συμβούλιο. Μετά έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τον ύπατο εκπρόσωπο που είναι και αντιπρόεδρος της Επιτροπής και παράλληλα ε, προεδρεύει του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και ταυτόχρονα το Συμβούλιο δίνει εντολή στον του εκπρόσωπο που έχει ως καθήκον να έρθει σε επαφή, να συμβάλλει μάλλον με τις προτάσεις στην ανάπτυξη της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Και αυτή η εικόνα αφορά μόνο την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Δεν περιλαμβάνονται εδώ άλλες εξωτερικές δραστηριότητες. Είναι πλέον λοιπόν σαφές, σαφές ότι η οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων θα είναι πολύπλοκη. Και είδαμε και στο πρόσφατο παρελθόν κάποια παραδείγματα για τις εξωτερικές υπηρεσίες. Και είδαμε ότι είναι κάθε άλλο παρά εύκολο το εγχείρημα. Αυτές τις αμφιβολίες θα τις αφήσω για τη συζήτηση και πιθανώς και για, την, ε, για τους ομιλητές αύριο το πρωί. είναι από ό,τι φαίνεται επιτακτική ανάγκη να υπάρχει συνεκτικότητα όχι μόνο για την εξωτερική πολιτική. Ίσως ακόμη πιο δύσκολο είναι αν προσθέσει κανείς την εξωτερική πολιτική και άλλες εξωτερικές δράσεις. Συνοψίζοντας, η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με τη συνθήκη της Λισαβόνας ενισχύεται ουσιαστικά για την εξωτερική δράση, ειδικά στον τομέα της κοινή εμπορικής πολιτικής. Δεν είναι και τόσο σαφές όμως εάν τα κράτη-μέλη και τα όργανα είναι έτοιμα να καλύψουν αυτό το νέο πλαίσιο, να δώσουν σάρκα και οστά σε αυτό το νέο πλαίσιο. Θα το δούμε. Ένα σημαντικό, μια σημαντική παρατήρηση είναι αυτή η εδραίωση που προανέφερα, είναι μάλλον επιφανειακή ε, εξωτερικών πολιτικών όσον αφορά τις εξουσίες, τις ε, ε, διαδικασίες. Είναι ένας ογκόλυφος, να το πούμε έτσι, για το μέλλον και γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ναι, ότι με τη συνθήκη της Λισαβόνας η Ευρώπη στηρίζει κατά κάποιο τρόπο τις ευθύνες της στον τομέα της παγκοσμιοποίησης. Είναι ένα κομμάτι από τη διακήρυξη του Λάκεν, αλλά πολλά μένουν ακόμα να γίνουν. Ευχαριστώ. Θα έλεγα ότι τα νομικά πλαίσια είναι νομικά πλαίσια. Πρέπει να ακολουθήσει και η πολιτική. Και η πολιτική πρέπει να ακολουθήσει. Πρέπει να δούμε. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο Τιμπορ Παλανκάη, ε, τιμημένος με το βραβείο Ζωμονέ για το 2010 και ε, έχει την έδρα Ζωμονέ στο Πανεπιστήμιο Κομβίνιου στην ε, Βουδαπέστη. Τιμπορ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πριν να ξεκινήσω με το θέμα, προσπάθησα να κάνω κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις. Πρώτα-πρώτα προσπάθησα να εμείνω στον τίτλο της συνεδρίας, δηλαδή να μιλήσω κάτι για τις παγκόσμιες προκλήσεις και να μιλήσω και για το νέο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπ' αυτή την έννοια δεν θα περιοριστώ στην συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά θα μιλήσω και για το πρόγραμμα της Λισαβόνας και την συνέχεια αυτού και το πρόγραμμα Ευρώπη 2020. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντικό, δεν είμαι νομικός Δεν θέλω να μειώσω τη σπουδαιότητα του νομικού και του θεσμικού πλαισίου, αλλά πρέπει να γεμίσει αυτό το πλαίσιο με κάποια στρατηγική, με όραμα και πολύπλοκα σχέδια δράσης. Και το 2020, Ευρώπη 2020, είναι μια στρατηγική για το μέλλον της Ευρώπης. Και με βάση αυτό προσπάθησα να μην κάνω μόνο αναλυτικές παρατηρήσεις, αλλά να κάνω και κάποιες προτάσεις. Γιατί το 2020 βρίσκεται υποδιαμόρφωση, δεν έχει οριστικοποιηθεί. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις, κάποιες ενδείξεις που θα μπορούσαν ίσως να βοηθήσουν στην ενίσχυση του προγράμματος αυτού που όπως είπα είναι η υποδιαμόρφωση. Όσον αφορά τις προκλήσεις θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και να τονίσω την πολυπλοκότητα των προκλήσεων. Αντιμετωπίζουμε όντως ποιοτικέ αλλαγές σε όλα τα στοιχεία της ε, κοινωνικο-οικονομικής δομής, ε, τεχνολογία, κοινωνικο-οικονομικές σχέσεις, ε, παγκόσμια ολοκλήρωση. Είναι μια σημαντική εξέλιξη ή τις αλλαγές όσον αφορά τους παράγοντες παραγωγής εκτός από τους παραδοσιακούς που είναι η γη, το κεφάλαιο και η γνώση τώρα έχουμε και την τεχνολογία, συγγνώμη, τώρα έχουμε τη γνώση που είναι ένας νέο παρά, νέος παράγων ε, δυνατοτήτων και θα περιοριστώ ίσως για την ανάγκη να υπάρξουν νέα παραδείγματα όσον αφορά αυτές τις ποιοτικέ αλλαγές. Πρέπει δηλαδή να αλλάξει η οπτική μας για το ΑΕΠ, ας πούμε ή θα πρέπει να επαναξιολογήσουμε τις θεωρίες για το συγκριτικό κόστος ωφέλεια ή την εφαρμοσιμότητα μιας θεωρίας ή την έννοια του ισοζυγίου πληρωμών και διάφορα άλλα. Για τις νέες προκλήσεις λοιπόν, το βασικό πρόβλημα που βλέπω εγώ είναι ότι είναι πολύ ανεπαρκείς οι απαντήσεις που δίνουμε και το θέτω υπείως. Έχουμε μεγάλες κρίσεις. Πέρα από την πρόσφατη παγκόσμια οικονομική κρίση, αντιμετωπίζουμε και μια ενεργειακή και περιβαλλοντική κρίση και φοβούμε ότι αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό από την οικονομική κρίση. Πιο σοβαρή όσον αφορά την πολυπλοκότητα των λύσεων και το μελλοντικό αντίκτυπο που θα έχουν αυτές. Έχω την αίσθηση επίσης ότι θα πρέπει να τονίσουμε και τις κοινωνικές κρίσεις, οι οποίες έχουν ευρύ αντίκτυπο στην κοινωνία. Έχουμε τους, ε, τις διάφορες ακραίες τάσεις, τη, το λαϊκισμό, ε, Προσπάθησα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις ε, για τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ένωση, εκπαίδευση, γεωργία, γύρανση του πληθυσμού. Όσον αφορά τώρα τις παρούσες κρίσεις, η τελευταία κρίση έχει αρκετές διαστάσεις. Μία σημαντική διάσταση ήταν ότι κάθε σύστημα, κάθε χώρα, κάθε φορέας πρέπει να πληρεί κάποιες δραστηριότητες ανάλυσης και πληροφόρησης. Να ξέρεις πού βρίσκεσαι δηλαδή, πώς έχουν τα πράγματα. Και κάθε οργανισμός έχει τις στατιστικές του υπηρεσίες, ή τον σχετικό μηχανισμό ανάλυσης. Και πιστεύω ότι ένα από τα προβλήματα της κρίσης αυτή ήταν ότι σε αυτού του είδους τις πληροφορίες είχαμε αναλυτικές αρμοδιότητες οι οποίες ε, ε, ε, είχαν πολλά κενά και δεν αφορά μόνο τις προβολές, τις προγνώσεις περί κρίσης. Δηλαδή, Μπορεί κανείς να προβλέψει τις ε, προγνώσεις για την Ευρώπη. Όλοι ξέρουμε ότι ήταν, ε, είχαν υποτιμηθεί. Αλλά έλλειψη στατιστικών είναι ένα θέμα. Υπάρχουν προβλήματα για την λογιστική αποτίμηση. Όλα αυτά είναι μέρος της κρίσης. και έπρεπε να επιληθούν. Ίσως θα πρέπει να αναφέρουμε και τις νομικές πτυχές. Υπήρξαν κάποιες δράσεις, οι οποίες όμως ε, από νομικές απόψεις δεν ορίζονται. Δηλαδή έγιναν κάποια εγκλήματα τα οποία όμως νομικώς δεν ορίζονται. Κερδοσκοπία ας πούμε. Και το ίδιο ισχύει και για τις ηθικές πτυχές της οικονομικής κρίσης. Και πάλι θα πρέπει να τονίσουμε ότι μπορούμε να κατηγορήσουμε τους κερδοσκόπους για την απληστία τους. Αλλά συνένοχος ήταν όλος ο πληθυσμός των κερδοσκόπων. Όλοι θέλαν κατά κάποιο τρόπο, έπεσαν οι θελημένα θύματα της απάτης. δεν θα αναλύσω ιδιαίτερα τις απαντήσεις. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες ότι ένα από τα κεφαλώδη συμπεράσματα είναι ότι δεν αρκεί η νομισματική ένωση. Χρειαζόμαστε και μια οικονομική ένωση και πολιτική ένωση. Οι τελευταίες αποφάσεις για νέα ταμεία, νέους μηχανισμούς είναι σημαντικές αποφάσεις και πρόσδεκτες. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεπεράσουν, να πάνε πολύ πιο πέρα από το να δημιουργήσουν ένα μηχανισμό διάσωσης. Πρέπει να γίνουν μηχανισμός πρόληψης. Πρόληψη όχι μόνο της νομισματικής ε, αηφορίας και σταθερότητας, αλλά πραγματικής σύγκλησης θα έλεγα. Θα τόνιζα το θέμα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Όσον αφορά τώρα την ενεργειακή κρίση. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της εποχής μας είναι ότι έχουμε μια τεχνολογική επανάσταση χωρίς ενεργειακή επανάσταση. Οι προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις ήταν και ενεργειακές. Αυτή τη φορά έχουμε τεχνολογική επανάσταση χωρίς όμως να έχουμε ποιοτική αλλαγή στις ενεργειακές δομές. Και είναι προφανές ότι οι ισχύουσε δομές δεν μπορούν να προχωρήσουν. Όλοι συμφωνούμε ότι αν συνεχίσουμε με αυτές τις δομές θα καταστρέψουμε, θα καταστραφούμε. Είναι θέμα κοινή λογικής ότι υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις για την ενέργεια. Πρέπει να είναι καθαρή, φτηνή και ασφαλής. Και δεν ισχύει αυτό για τις υπάρχουσες δομές. Θα έλεγα ότι ειδικά το πρόγραμμα Ευρώπη 2020 καλεί κάποια σημαντικά συμπεράσματα και περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία, αλλά δεν αρκούν είναι αρκετά αόριστα, δηλαδή νέες ενεργειακές αποκρίσεις, αυξημένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενεργειακή ασφάλεια, αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, ολοκλήρωση των αγορών. Αλλά αυτό που χρειάζεται για να αντιμετωπιστεί σοβαρά η ενεργειακή κρίση είναι πολύ περισσότερο. Χρειάζονται πόροι Χρειάζονται, χρειάζεται έρευνα και υποδομές. Υποδομές για να αλλάξει η υπάρχουσα ενεργειακή δομή. Συμφωνώ απόλυτα με το σχέδιο Delors που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, το οποίο τονίζει τη σπουδαιότητα του προβλήματος και θα έλεγα, θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα των υποδομών. Πρόσφατα ε, έχουμε ε, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, Τεχνικό είναι δυνατά, χρειαζόμαστε υποδομές. Έχουμε βενζινάδικα, αλλά θα πρέπει να δημιουργήσουμε σταθμούς φόρτισης μπαταριών. Και αυτό προϋποθέτει πολιτικές χρηματοδότησης. Γιατί οι ενεργειακές εταιρείες δεν ενδιαφέρονται και οι κυβερνήσεις δεν ενδιαφέρονται. Οι κυβερνήσεις εισπράττουν πολλούς φόρους με βάση τις υπάρχουσες ενεργειακές υποδομές. Και αυτό θα πρέπει να αλλάξει και να προβλεφθούν νέοι δρόμοι μία, μάλλον κάποιες σύντομες παρατηρήσεις και για την κοινωνική κρίση. Οι ανισότητες μεταξύ των τάξεων, περιφερειών, των χωρών αυξάνουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως είναι κάπως διαφορετική ως προς αυτό, αλλά Όσον αφορά τα νέα κράτη-μέλη, πρέπει να πω ότι τα κοινωνικά προβλήματα επιδεινώθηκαν λόγω των ε, αποτελεσμάτων της, των διαφόρων μεταρρυθμίσεων. Και αυτό οδηγεί οδηγεί σε κόπωση, όχι μόνο την κόποση της διεύρυνσης ε, ή των μεταρρυθμίσεων. Ε, εμφανίζονται, εμφανίζεται μια κόποση πάντως που ενισχύει τα προβλήματα και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και ένα άλλο θέμα επίσης που είναι σημαντικό η μεταρρύθμιση του κράτους προνοίας. Είναι ένα πολιτισμικό επίτευγμα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κράτος προνοίας. Δεν πρέπει να, να, να, απαλληφθεί, πρέπει να μεταρρυθμιστεί, να προσαρμοστεί στις νέες προκλήσεις για να γίνει πιο ανταγωνιστικό αντί να είναι μόνο προστατευτικό και αναδιανεμητικό. Θα ήθελα να πω κάτι ακόμα αν μου δίνετε το περιθώριο, να πω δύο λόγια για τη γύρανση του πληθυσμού, που είναι ένα μεγάλο, μια μεγάλη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και μιλώ για αυτό το πρόβλημα γιατί αισθάνομαι κάπως συνένοχος. Δεδομένης της ηλικία μου. Είμαι σε ηλικία συνταξιοδότησης. θα έπρεπε να είμαστε χαρούμενοι. Ζούμε περισσότερο. Αλλά τώρα μιλάμε για σοβαρή κρίση. Και μας ανησυχεί αυτό βεβαίως. Πρέπει κάπως να αντιμετωπιστεί. Και πιστεύω ότι σε αυτό το τομέα δεν δώσαμε επαρκείς απαντήσεις. Είναι πολύπλοκο θέμα. Πρώτον είναι η αναδιάρθρωση του, ε, της εργασιακής ζωής. Τον 19ο αιώνα δουλεύαμε 140.000 ώρες, τώρα δουλεύουμε λιγότερο, 74.000 ώρες λόγω της αύξησης παραγωγικότητας Έχουμε περιορίσει το, τις εβδομάδες εργασίας, αλλά ε, ε, έγινε παράταση στα χρόνια. Και πολλές φορές τις μεταρρυθμίσεις βλέπουμε το, να γίνεται το αντίθετο, δηλαδή περιορίζεται ο χρόνος εργασίας, δηλαδή η σύνταξη έρχεται νωρίτερα αντί να έρχεται αργότερα. Είναι πολύ πολύπλοκο το θέμα και αυτό δεν αφορά μόνο τη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών ταμείων αλλά και τη διαβίου εκπαίδευση, τη φορολογική πολιτική. Η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως υπόδειγμα δεν νομίζω ότι πρέπει να δεχτούμε αυτό που λένε, δηλαδή ε, παρακμή της Ευρώπης. Η Ευρώπη μπορεί να δώσει ένα θετικό παράδειγμα για τον υπόλοιπο κόσμο. Thank you Now a logistical problem. Ευχαριστώ. Έχουμε ένα τεταρτάκι το πολύ για ερωτήματα, για απαντήσεις και για να δώσουμε και λίγα λεπτάκια στον ε, συντάκτη της ε, συνόδου, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, να μας μιλήσει. Ε, ίσως πριν θέσετε τα ερωτήματά σας, να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο σύντομο. Αυτή η σύνοδος έχει να κάνει με τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει παγκόσμιες οικονομικές προκλήσεις. Ακούσαμε πολλά για το νομικό πλαίσιο και το πώς έχει αλλάξει. Ακούσαμε επίσης πολλά για την πολιτική βούληση ή την έλλειψη αυτής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Μία πτυχή που τουλάχιστον για μένα δεν αναφέρθηκε επαρκώς είναι η πραγματική οικονομία. Γιατί μπορεί να έχουμε το κατάλληλο νομικό πλαίσιο, μπορεί να έχουμε την επαρκή πολιτική βούληση, αλλά μπορεί να έχουμε και μια λιμνάζουσα οικονομία. Και αυτό μπορεί να είναι πολύ αποφασιστικό παράγοντα στο πόσο και πώ μπορείτε να αντιμετωπίσετε το οποιοδήποτε πρόβλημα. Και αυτό δεν είναι θεωρητικό, ούτε φανταστικό ερώτημα. Γιατί βραχυπρόθεσμα, οι βραχυπρόθεσμες και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι καλές σε σύγκριση με άλλα μέρη του κόσμου. Και αν αυτές οι προοπτικές όντως βγουν πραγματικές, θα επηρεάσουν ε, πάρα πολύ τη δική μας δυνατότητα, είτε μεμονωμένη είτε συλλογική, να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο τις παγκόσμιες οικονομικές προκλήσεις, αλλά ακόμη και τις προκλήσεις που αφορούν μόνο εμάς, την Ευρώπη. Τούτου λεφθέντος έχετε το λόγο για να θέσετε ερωτήματα, σας παρακαλώ πείτε μας το όνομά σας και από πού είστε. Ευχαριστώ από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Ε, μία ερώτηση για τον καθηγητή Γκρίλερ. Η δική σας εκτίμηση για την περίπτωση Μερκιούρ που συζητείτε τώρα γίνεται συζήτηση και στα Ηνωμένα Έθνη και στους κόλπους της Κομισιόν και με τον, με τον υπατή εκπρόσωπο της Κομισιόν για το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, ανταγωνιστικότητα, είναι ανταγωνιστική γιατί στην, σε όλη αυτή την ε, περίοδο που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Καλύτερα να ακούσουμε πρώτα όλα τα ερωτήματα και μετά να σας απαντήσουν ε, σύντομα η κυρία εδώ Tengo tres Τρεις ερωτήσεις. Έγινε λόγος για σύσταση Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Ερωτώ. Σημαίνει ότι αποσυρώμαστε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή θα έχουμε διπλή ιδιότητα. Να έχουμε και το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, να συμμετέχουμε και στο Διεθνές Νομισματικό θα μπορούσαμε να καλύψουμε και τα δύο. Έχουμε, έχουμε επαρκή μέσα. Άλλη ερώτηση. Τι γίνεται με την πραγματική οικονομία. Τι γίνεται με τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μιλώ κυρίως για τα κράτη της Ευρωζώνης. Αν πάρουμε την παραγωγικότητα, ας πούμε, οι διαφορές μεταξύ κρατών μελών μεσοπρόθεσμα δεν επηρεάζουν θέματα δαπανών και εσόδων. Δεν θα οδηγηθούμε, σας ερωτώ, σε νέα πάλι κρίση του ευρώ. Επόμενη ερώτηση, ευχαριστώ. Άντζελο Σαντακοστίνο λέγομαι, από την Μπρέσα, από το κέντρο μελετών της Μπρέσα. Στα Ιταλικά μιλώ γιατί έχουμε εξαιρετικού διερμηνείς, λέει ευγενικό αγορητής. Έχω κάμποσε ερωτήσεις, να θέσω τουλάχιστον μία. Για το είναι εμπορική πολιτική. Έχουμε μια σημαντική συνέπεια από τη συνθήκη μόνο δύο ομοφωνία πλέον περνάνε οι συμφωνίε με τρίτε χώρες. Δεν τίθεται πλέον θέμα άρνηση κυρίας. Αυτές τις μέρες, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, άρχισε η συζήτηση του θέματος για μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών. Μιλάμε και μια εμπορική συμφωνία τέλο πάντων. Με το ψευδοκράτος οπότε να επιβλακεί το θέμα της Τουρκίας, η οποία Τουρκία αρνείται να ανοίξει τους λιμένες της. Πώς βλέπετε αυτό το σημείο? Μία τέτοια συμφωνία σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε τη λεγόμενη Βόρεια Κύπρο, όπως λέει ο μιλητής. Οπότε, de facto, δεχόμαστε τη διοχοτόμηση της νήσου ή κάτι τέτοιο θα διευκόλυνε την επανένωση της νήσου. I shall leave this question to my Austrian friend to answer. Μάλλον ο συνάδελφος από την Αυστρία θα σας απαντήσει σε αυτό. Από το Πανεπιστήμιο στην, από Πανεπιστήμιο στην Πορτογαλία έχω κάποια ερωτήματα. Είπατε πολύ σωστά ότι στην συνθήκη της Λισαβόνας, στο πέμπτο τμήμα για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζονται οι προποθέσεις για την οικονομική συνεργασία, τη συνεργασία γενικώ, τα προαπαιτούμενα της δημοκρατίας και κάτι που ίσχυε και στην Ίκαια ήταν η βιώσιμη ανάπτυξη. Όχι απλώς να δίνουμε έτσι λεφτά, αλλά να ζητούμε να γίνεται και κάτι. Τώρα βρισκόμαστε στο... Αυτά τα, αυτά τα, αυτά τα προαπαιτούμενα βρίσκονται στο αντίστοιχο σημείο της ε, Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να ζητήσουμε το, περισσότερο, το δυνατόν περισσότερο να σέβονται οι χώρες αυτές τους κανόνες του παιχνιδιού. Γιατί διαβάζουμε την προηγούμενη συνθήκη, διαβάζουμε και τούτη και νομίζω ότι υπάρχει ασυνέπεια. Γιατί ε, δεν φαίνεται σαν να ζητούμε ότι την ανάπτυξη όντω, δεν τονίζεται τόσο πολύ αυτό. Νομίζω ότι κάναμε ένα βήμα προ τα πίσω. Και δεύτερο, είπατε σε κάποια στιγμή ότι υπάρχει προοπτική για την Τόχα. Μάλλον και στον Επίτροπο Ντεχούχτ πρέπει να θέσω το ερώτημα αυτό. Είπατε ότι είσαστε απεσιόδοξο για το πώ θα εξελιχθεί ο, ο γύρος της Δόχα δύο ερωτήματα γιατί, ακόμη γιατί αλλιώ δεν θα έχουμε χρόνο να απαντήσουμε. Χάνα πήρε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο στην ε, Βιέννη. Για την ομοφωνία που είπατε, ακούστηκε από τα τελευταία ε, πάνελ, ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει ε, αναγκάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιταχύνει είτε να ενοποιηθεί περισσότερο, να μην έχει δηλαδή μόνο το ευρώ, να έχει η φορολογική πολιτική, διάφορα μέτρα, εν πάση περιπτώσει, μεγαλύτερη συνέπεια, μεγαλύτερη ένωση, εν πάση περιπτώσει, ή να διαλυθεί. Αυτό υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να δει ποιο είναι το νέο μοντέλο που θα μπορούσε να πτυχθεί. Και εδώ θέτω το ερώτημά μου. Για τα τελευταία δύο σχόλια που ακούστηκαν, ακούστηκε το ερώτημα εάν στο μέλλον θα υπάρξει ανάπτυξη. Αυτό ήταν το τελευταίο ερώτημα. Φτάνουμε σε ένα σημείο στασιμότητας. Και κατά πάσα πιθανότητα θα συμβεί, θα υπάρξει αυτή η στασιμότητα. Οπότε, ερώτηση, πρέπει όντως να αναπτυχθούμε και πρέπει να το δούμε αυτό σοβαρά. Δηλαδή, αυτό αυτό δεν είναι ένα από τα βασικά καθήκοντα των πολιτικών, των θεσμικών οργάνων, να εγγυηθούν την αναπαραγωγή με πολιτικούς όρους, χωρίς αυτό να εμποδίζει την κοινοτομία. Δεν θα πρέπει να πάμε σε μια καινοτόμα αναπαραγωγή αντί για μια ποσοτική ανάπτυξη. το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο δεν είναι κάτι που ξεπερνάει αυτό το παλιό όραμα της ποσοτικής ανάπτυξης των περισσότερων αυτοκινήτων, των περισσότερων ε, ποσοτικά πραγμάτων. Δεν πρέπει να είναι ποιοτική η αλλαγή ώστε να εξασφαλίσουμε αναπαραγωγή. Και σε σχέση με αυτά που είπε ο συνάδελφος στο τέλος για, την, ε, για τον πληθυσμό. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Βέβαια, πρόεδρε, τώρα μπορεί να μην θέτω το σωστό ερώτημα 6 ώρα το απόγευμα, αλλά το πάνελ μίλησε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς μπορούμε να λύσουμε, να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, εντάξει. Αλλά το πρόβλημα στην Αφρική, ας πούμε, είναι η υποανάπτυξη και η φτώχεια. Δεν ξέρω κατά πόσο θεωρείτε ότι υπάρχουν τα συστήματα για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, αλλά με τους, με τους στόχους της χιλιετίας τι γίνεται. Είμαστε πολύ μακριά από την εκπλήρωσή τους. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό γιατί η Αφρική είναι η γειτονική ήπειρος. Θα μιλήσουμε για τη μετανάστευση βέβαια, αλλά πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε αυτό το παγκόσμιο πρόβλημα της υποανάπτυξης και της φτώχειας. Ευχαριστώ. Στα Ισπανικά από το Πανεπιστήμιο της Μάλαγα. Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ τους αγορητές και των τριών ε, συνόδων σήμερα. Μία ερώτηση για τον τίτλο της διάσκεψης. Νέο, Νέο πλαίσιο της Λισαβόνας για αντιμετώπιση των προκλήσεων και γίνεται λόγος για το νέο θεσμικό πλαίσιο, για τις νέες θεσμικές σχέσεις. Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Αυτό έχουμε δει σήμερα. Μακάρι να λειτουργήσει το σύστημα να του δώσουμε και ένα νόμπελ. Μιλάμε για νέα θεσμική θεωρία. Μιλάμε για κοινωνικό κεφάλαιο, για να υπάρχει θεσμική εμπιστοσύνη, αλλά πίσω από όλα αυτά τι κρύβεται. Θέλουμε να πετύχουμε την ευημερία των πολιτών. Αυτά μας είπε σήμερα ο πρόεδρος Μπαρόσο. Σκεφτείτε το, γιατί είναι ήδη αργά, δεν θα πρέπει να γίνει και αυτός ο προβληματισμός. Πέραν του να κάνουμε απολογισμό των θεσμικών ισορροπιών θα πρέπει να κάνουμε ένα απολογισμό για να δούμε κατά πόσον η νέα δομή βελτιώνει την παλιά. Γιατί συνήθως τις αλλαγές γι' αυτό τις κάνουμε. Το νέο θεσμικό πλαίσιο βελτιώνει την λειτουργία του συστήματος. Ακούστηκαν διάφορες προκλήσεις περιβαλλοντικές, απασχόληση κτλ κάνουμε πίσω, οπισθοχωρούμε ή βελτιώνουμε τα πράγματα. Okay, I propose, uh, Θα ζητήσω από τον κάθε μιλητή να απαντήσει σε τρία λεπτά. Γιατί οι διερμηνείς θα μας παρατήσουν και είναι σημαντικό να τους έχουμε σε μια τέτοια συνεδρίαση με τόσες πολλές γλώσσες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τον κύριο Κίνγκ και μετά ούτως ή άλλως σου χρωστάμε χρόνο για παρέμβαση. Μήπως να απαντήσουν καλύτερα οι υπόλοιποι και να παρέμβω εγώ σε ό,τι περισσέψει. Εντάξει, οπότε αλλάζουμε σειρά. Πολύ σύντομα για το αν θα πρέπει να αναπτυχθούμε περισσότερο. Πολύ καλό το ερώτημά σας. Μία πτυχή που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι η φτώχεια. Έχουμε αρκετά προϊόντα, έχουμε αρκετές υπηρεσίες για την ευημερία όλου του πληθυσμού. Οπότε νομίζω ότι είναι αδύνατο να σκεφτούμε πάυση ανάπτυξης. Και κάτι άλλο με το οποίο συμφωνώ είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αναπτυσσόμαστε και την ποιότητα της ανάπτυξης. Εγώ είπα ότι τώρα, έτσι όπως έχουν οι δομές, η ανάπτυξη οδηγεί σε καταστροφή. Οπότε πρέπει να αλλάξουμε. Και νομίζω ότι όντως πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Τρία λεπτά. Τρία λεπτά. Ένα για την υπόθεση Mercury. Δεν μπορώ να το λύσω. Σε ένα λεπτό δεν μπορώ να το λύσω σίγουρα. Το μόνο που θέλω απλώς να πω είναι ότι από ό,τι καταλαβαίνω εγώ αυτό δείχνει ακριβώς τις ε, ασυνέπειες που υπάρχουν στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια και σχετικό, σχετικό μηχανισμό. Υπάρχουν πολλοί παίκτε που θα ήθελαν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο. Νομικώ μιλώντα, είναι σαφέ ότι το Συμβούλιο είναι επικεφαλή. Αυτό πρέπει να καθορίσει τη θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την περίπτωση. Τα κράτη-μέλη η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προσωπείται σε επίπεδο ΙΕ, θα πρέπει να λάβουν θέση σε επίπεδο ΙΕ. Μόνο όμω αν υπάρξει ή αν χρειαστεί ομοφωνία είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να φτάσουμε σε ομοφωνία στο Συμβούλιο και μετά θα παρέμβει η εκπρόσωπο και θα έρθει η Κομισιόν και θα προσπαθήσει να λάβει τον ηγετικό ρόλο. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που απορρέουν από την ομοφωνία σε θέματα ΚΕΠΑ και από την ε, πολυμορφία των παικτών που δεν την ενοποιεί καθόλου η συνθήκη της Λισαβόνας. Ένα λεπτό λοιπόν για αυτό. Τώρα για το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες ε, για αυτή την συμφωνία που αναφέρατε. Χωρίς ε, μικρόφωνο κύριο, κύριος Κίνγκ. Νομικός και πάλι δεν υπάρχουν εξωτερικές σχέσεις με το ψευδοκράτος. Είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο στο βαθμό που δεν εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο εκεί. Αλλά δεν γίνεται να, συνάψουμε συμφωνία σαν να θεωρούσαμε το βόρειο τμήμα της Κύπρου τρίτη χώρα. Και τρίτο σχόλιο, αιρεσιμότητα. Αν κατάλαβα καλά, για την ε, αναπτυξιακή συνεργασία. Νομίζω ότι έχετε δίκιο. Αν πάμε στο κείμενο της συνθήκης, η διατύπωση που, που δημιούργησε, τις προκάλεσε τις ε, αποφάσεις του ΔΕΚ, ήταν ότι είναι ε, αίρεση ε, ο σεβασμός του, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ανάπτυξη. Αλλά αυτό δεν υφίσταται πια. Με δεδομένο με δεδομένη τη σημασία και τη σχέση των γενικών αρχών στις διατάξεις για την αναπτυξιακή συνεργασία και τη σχετική πολιτική, άρθρο 208, Λαμβάνοντα αυτό υπόψη, μπορεί να καταλήγαμε σε διαφορετικό αποτέλεσμα. Εγώ αμφιβάλλω. Θα έλεγα ότι με βάση εκείνη τη διατύπωση και τι γενικέ διατάξει θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στον ίδιο, στο ίδιο σημείο. Αλλά συμφωνώ ότι δεν είναι όσο σαφέ ήταν στο παρελθόν. Θα σας απαντήσω στα ε, ισπανικά. Για το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο δεν έρχεται σε αντίφαση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είπαμε ότι προβλέπεται ήδη και στη συνθήκη. Όμως αντιθέτως οι Ευρωπαίοι θα αναλάβουμε την ευθύνη μας διότι έχουμε κατά κάποιο τρόπο βαλκανοποιηθεί στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο το δημιουργούμε για να ε, προστατεύσουμε την ικανότητά μας αλλά να δημιουργήσουμε και ένα διεθνές νόμιμο νομισματικό ε, πλαίσιο ε, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε ε, την κομμουνιστική Κίνα που είναι ο μεγαλύτερος πιστωτής των ΗΠΑ. Δεν ξέρω αν είστε από την Αργεντινή εσείς. Είδαμε ότι η Αργεντινή, το Μεξικό, η Βραζιλία μεταξύ άλλων βρίσκονταν σε δραματική κατάσταση το δεκαετία του 90, τώρα είναι μέλη του ΠΟΕ. Άρα υπάρχει περιθώριο. Το θέμα των προκλήσεων τώρα, Ντόχα. Ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής ε, τέτοιων σχέσεων, ε, ε, σχέσεων του Κοινοβουλίου. Εμείς ανοίγουμε τις αγορές. Η περιορίζουν τις συμβάσεις. Οι χώρες BRIC και οι υπόλοιπε ανοίγουν τις αγορές τους για τα, διεθνή, για τα βιομηχανικά προϊόντα και τις υπηρεσίες, αλλιώς δεν θα υπάρξει συμφωνία. Εμείς πρέπει να επιβιώσουμε η Κοπενχάγη και το Μεξικό. Κοιτάξτε, ε, οι δύο που μολύνουν περισσότερο, που είναι η ΙΠΑ και η Κίνα, μπλοκάρουν μία πρόταση που είναι το 2020-20, πρόταση που κάναμε, ε, και πρέπει και αυτοί να περιορίσουν τις εκπομπές διότι υπάρχει ένα θέμα που είναι ξεκάθαρο η μεγαλύτερη πρόκληση του Προέδρου Ομπάμα που θα πρέπει να τώρα μεταρρυθμίζει το σύστημα υγείας ε, το πρόβλημα στην Ευρώπη δεν ισχύει. Στην Ευρώπη καλύπτεται όλος ο πληθυσμός. Στην Κίνα δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει πρόσβαση όλου του πληθυσμού σε βασικά προϊόντα όπως είναι η υγεία. Εμείς δεν είμαστε άσχημα και οι υπόλοιποι πρέπει να συμβάλλουν. Και κλείνω κύριε Πρόεδρε αναφέροντας, ε, με μια αναφορά στους στόχους της ε, χιλιετίας. Πιστεύω ότι όλα αυτά συνδέονται με τους στόχους της χιλιετίας. King. Ο κύριο Tim King έχει το λόγο τώρα, συντάκτης του European Voice και θα απαντήσει και στα ερωτήματα που δεν τολμούσατε να θέσετε αλλά που πάντα θέλατε να θέσετε. Όπως τι είναι ο συντάκτης συνεδριάσεων. Ούτε εγώ ακριβώς ξέρω, γιατί έτσι περνάω μια υπαρξιακή κρίση μου την, έχει, μου την έχουν προκαλέσει πολλά πράγματα. Ε, ένα από αυτά ήταν και οι κρίσεις που ανέφερε ο προηγούμενος ε, συνάδελφος ε, για την ενέργεια, για τον γυράσκοντα πληθυσμό, μετά διάφοροι θέλετε να προσθέσετε και τη μετανάστευση και τις κλιματικές αλλαγές και πολλά άλλα προβλήματα. Άλλη υπαξιακή κρίση προέκυψε από αυτά που είπε ο Κάρελ Ντεχούχτ για, το, για αυτά που είπε για τον Ζαν Μονέ, που ήταν κάποιο, που ήθελε να είναι κάποιο και ήθελε να κάνει κάτι. Εγώ ούτε κάποιο είμαι, ούτε τίποτα κάνω. Ποτέ δεν με προσκάλεσα να δείπνήσω στον ε, Λευκό Οίκο. Την τελευταία φορά που ήμουνα στην Ουάσιγκτον όμως, πήγα σε ένα εστιατόριο που ε, μου είπαν ότι έπαιζε και σε μια σειρά, στην σειρά The West Wing που έπαιζε στην τηλεόραση. Αυτό ήταν το πιο κοντινό που έφτασα ποτέ εγώ στον ε, Λευκό Οίκο. Στις 9 Μαΐου μας είπατε ότι έγινε η Επανάσταση. Δεν ήταν η 9η Μαΐου, ήταν η 10η Μαΐου. Και σε το λέει κάποιος που περίμενε την επιτυχία από τους ε, Υπουργούς Οικονομικών. Να σας θυμίσω κάποια από τα πράγματα που είπε ο κύριος ε, Κρεσπόν στα σχόλιά του για την ε, πρόσκληση σε συλλογική αυτοκτονία. Είπε ότι οι Βέλγοι είναι σαν τον Κάρολο τον Πέμπτο. Ο Κάρολος ο Πέμπτος όμως έφτιαχνε στη όταν πήρε σύνταξη ρολόγια στην Ισπανία. Δεν ξέρω πώς συνδέεται αυτό με τους Βέλγους. Δεν θέλω τώρα να λέω τα προφανή, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν είναι τόσο νέο. Γιατί οι θεσμικές αλλαγές, όπως γίνεται συχνά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκαλούνται από κρίσεις. Ο κύριος Σαρκοζή συχνά αναφέρεται στις συνεδριάσεις ε, του Eurogroup. Αυτό έγινε είτε στις 7 είτε στις 8 Μαΐου και το γεγονό ότι η εκπεριτροπή Προεδρία των, ε, στο, των Υπουργών ήταν, είχε τόσο μεγάλο άγχο για το αν θα επιτύχει η συνθήκη τη Λισαβόνα. Ε, έχει, η Ισπανική λοιπόν αυτή η εκπεριτροπή Προεδρία έχει μπει λίγο στο παρασκήνιο σε σχέση με την μόνιμη τώρα Προεδρία που έχουμε. Η Ισπανία πάλι αυτή τη στιγμή δεν είναι και στην καλύτερη θέση για να υποδεικνύει στους άλλους τι θα κάνουν. Σήμερα λοιπόν υπάρχει μια διάσκεψη και αύριο που γίνεται στο κτίριο Σαλεμάνι της Κομισιόν που την οργανώνει το τμήμα για την, το Υπουργείο Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Η συζήτηση ήταν όμως πιο επίγουσα και είχε και περισσότερες ενοχές από τα μέλη που συμμετείχαν. Εντάξει, συμμετείχαν και κάποιοι ακαδημαϊκοί, κάποιοι οικονομολόγοι που ένιωθαν και αυτοί αυτές τις ε, τύψεις. Ε, τώρα είναι και οι πολιτικοί που, έχουν, που νιώθουν τις τύψεις και οι τραπεζικοί. Εκεί όμως μιλούσαν για αποσύνδεση των ε, θεσμικών οργάνων και των αγορών. Ο Μπαρόζο ζητούσε γιατί έβλεπε ότι υπάρχει μια ευκαιρία και ετέθη ως προερώτηση αυτό από εσάς, ότι το θέμα δεν είναι ότι η κρίση μας έφερε σε κάτι καινούριο. Ε, είναι μια ευκαιρία να ενισχύσουμε τις εξουσίες κάποιων θεσμικών οργάνων και θα ήθελε αυτό να γίνει υπέρ της Κομισιόν και όχι του Συμβουλίου. Για τη Λισαβόνα τώρα. Η συνθήκη είναι ακόμη σε μια ενδιάμεση κατάσταση. Και για το ερώτημά σας για το Mercury, για την υπόθεση Mercury, που ήταν στη δεύτερη σελίδα του, της European Voice αυτής της εβδομάδας, η νομική, ο νομικός ορισμός δεν, ε, δεν λειτουργεί, γιατί όταν η Κομισιόν αποσύρει την πρότασή της, τι γίνεται. Ακόμη παίζονται θεσμικά παιχνίδια και νομίζω ότι αυτό θα μου δώσει ψωμί εμένα για, πολύ, για αρκετό καιρό ακόμα. Και στην πρώτη σελίδα έχουμε την άλλη υπόθεση για το εμπόριο με, την, με το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Γιατί με, την, με τις αλλαγές της, της, της συνθήκης της Αβώνας η πρόταση μιας, της είναι η πρόταση της Κομισιόν να έχει άμεσα, άμεσα εμπορικές σχέσεις με το υπόλοιπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, το βόρειο τμήμα της Κύπρου, το ψευδοκράτος. Και μετά η πρόταση αυτή περνάει στην, ε, στο κοινοβούλιο για την, ε, για τη συναπόφαση, γιατί εμπίπτει στη συναπόφαση. Οι αλλαγέ λοιπόν ακόμη εξελίσσονται. Και μια άλλη ακόμη αλλαγή που δεν ακούστηκε πολύ, το G20. Υπάρχει και εκεί αγωνία. Το G20 είναι, αποτελεί απειλή στα τα νέα θεσμικά όργανα απειλούν τα παλαιά, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεούται να υποβάλει νέα νομοθεσία, να αναλάβει αποφάσεις που αλλιώς θα λαμβάνονται σε επίπεδο G20. Και ακούσαμε τι είπε ο κύριος Δεχούχτ για το ότι αν δεν δουλέψει η Ντόχα θα πάμε σε διμερεί, σε εμπορικές σχέσεις κλπ. Και τι γίνεται αν αυτό ξαναπροκύψει και όπως είπε για την ε, πραγματική οικονομία ο στην πραγματική πολιτική. Μιλούμε για κοινωνικέ συνέπειε. Και στην άλλη διάσκεψη περιγράφουν πώ μια οικονομική κρίση οδηγεί σε μια κρίση στην πραγματική οικονομία, στις, στα δημόσια οικονομικά. Αλλά δεν προχωράνε για να πούνε ότι η κρίση στα δημόσια οικονομικά μπορεί να οδηγήσει σε, πολι... σε κρίση πολιτική νομιμοποίηση και μπορεί να αρχίσει να, αμφι, αμφισβητεί και τις, ε, το θεσμικά μας όργανα. Νομίζω ξεπέρασε το χρόνο μου και σας ευχαριστώ. Well, Κυρίες και κύριοι, θα έκανα μία μεγάλη μακροσκελή ομιλία στα ελληνικά για να κλείσω, αλλά θα μας φύγουν οι διερμηνείς, οπότε δεν θα σας πω τίποτα. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ και τους ομιλητές μας και καλό σας απόγευμα.